Rozumiem, Από ό,τι ξέρω μπορούμε να αρχίσουμε χωρίς άλλη καθυστέρηση. Η ημερήσια διάταξη είναι πολύ φορτωμένη σήμερα. Με κύριο θέμα την ακρόαση για τη δέσμη των γαλακτοκομικών και τις προοπτικές του γαλακτοκομικού τομέα που είναι πολύ επίκαιρο και σημαντικό θέμα. Συμφωνείτε νομίζω. Από ό,τι κατάλαβα μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη αφού έχουμε μόνο ένα θέμα υπάρχει αναμετάδοση και έχουμε διερμηνία σε 20 γλώσσες. Εκτός δηλαδή εστονικά, μαλτέζικα και σλοβακικά. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Με μεγάλη χαρά κηρύσω την έναρξη της ακρόασης αυτής για την αποτίμηση αξιολόγηση του τρέχοντος δημοσιονομικού ε, νομοθετικού πλαισίου και των, προοπτικών του γαλακτοκομικού τομέα μετά την, το τέρμα των ποσοστώσεων. Δεν υπάρχει πάρα πολύ χρόνος, οπότε πρέπει να πούμε ότι όσο πλησιάζει η μέρα λήξης των ποσοστώσεων τίθενται όλο και περισσότερα ερωτήματα και ανησυχίες. Υπάρχουν φόβοι για πιθανή κρίση στο γαλακτοκομικό τομέα και αγορά ελπίζω αφού ακούσουμε τους εξέχοντες εμπειρογνώμονές μας να μπορέσουμε να μάθουμε κάτι περισσότερο για τον πολύπλοκο χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητες του τομέα ίσως και για πιθανές λύσεις. Ο James Nicholson είναι ο εισηγητής μας, είναι για έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας και ασχολείται με το θέμα αρκετά χρόνια. Είχε αναλάβει εκθέσεις πολλές φορές Έχουμε εννέα ομιλητές στην ακρόαση, εμπειρογνώμονες. Θα δώσω δέκα λεπτά στον καθένα και παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο σας. Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα. Πρώτο θέμα εφαρμογή της γαλακτοκομικής δέσμης. Τρεις εμπειρογνώμονες μετά σύντομη συζήτηση. Θα μιλήσουν οι συντονιστές και όσοι θέλουν να θέσουν ερωτήματα ή έχουν απορίες. Επαναλαμβάνω ότι στο δεύτερο γύρο θα μιλήσουν κατά προτίμηση όσοι δεν μίλησαν στον πρώτο. Δεν είχαν ερωτήσεις να θέσουν. Φαντάζομαι λοιπόν ότι δεν θα θέσετε διπλά ερωτήματα. Πριν αρχίσουμε λοιπόν το πρώτο θέμα ή πάνελ θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο James Nicholson. Πεστε μας μερικά λόγια σας παρακαλώ για το θέμα και την ακρόαση ολόκληρη. Καταρχήν σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας καλωσορίζω όλους εδώ τους εμπειρογνώμονες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα. Το ενδιαφέρον φαίνεται ότι είναι υψηλό και αυτό δεν με εκπλήσει καθόλου, διότι ο γαλακτοκομικός τομέας έχει ζήσει μεγάλες ε, διαταραχές με μειώσεις των τιμών και πολλοί αναρωτιούνται τι μέλλον μπορεί να έχει ιδίω μετά την 1η Απριλίου και την κατάργηση των ποσοστώσεων. Γνωρίζουμε το παρελθόν του τομέα, το γνωρίζουμε από πολλά χρόνια, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε με την κατάργηση των ποσοστώσεων. Αφού η απόφαση λήφθη πριν από πολλά χρόνια, πρέπει τώρα να εφαρμοστεί. Η μέση τιμή των γαλακτοκομικών τους τελευταίους 12 μήνες έχει πέσει πάρα πολύ σε βαθμό που αρχίζουν να φαίνονται σημαντικές επιπτώσεις. Αυτό είναι το κύριο θέμα της έκθεσης μας, αλλά νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και γενικότερα για το καλακτοκομικό τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη διότι δεν έχω πιστεί μετά από αυτά που είδαμε τους τελευταίους 6 μήνες δεν έχω πιστεί από την αύξηση της παραγωγής γάλακτος γιατί δεν υπάρχει ανάλογη αύξηση της κατανάλωσης και επομένως υπάρχει πρόβλημα για την βιομηχανία. Η έκθεση λοιπόν αυτή είναι ιδιαίτερα επίκαιρη για την ιστορία του γαλακτοκομικού τομέα και η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε όλοι σήμερα είναι ότι παρά τις συζητήσεις που έγιναν επανειλημμένως και πρόσφατα στο Κοινοβούλιο για την κατάσταση και το μέλλον του γαλακτοκομικού τομέα πρέπει να σας πω με όλο το σεβασμό που σας οφείλω ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους οργανώνεται σήμερα η ακρόαση είναι ότι όλοι μπορούν να μας πούν ότι είναι απέσια και τρομερή η κατάσταση, αλλά εγώ αυτό που θέλω να μάθω, γιατί σε αυτό, επ' αυτού έχουμε ευθύνη ως ευρωβουλευτές, είναι να δούμε πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα και να βρεθεί ένα μέλλον για το γαλακτοκομικό τομέα και τους ακρότες που ασχολούνται με αυτόν. Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε δεν θα σας απασχολήσω άλλο θα ακούσω περισσότερο, αυτή είναι η δουλειά μου σήμερα και στα τέλη Φεβρουαρίου θα έχουμε μπροστά μας μια έκθεση που θα συζητηθεί, θα τροπολογηθεί και ελπίζουμε να έρθει η προσυζήτηση στο Κοινοβούλιο τέλη Απριλίου ή αρχές Μαΐου. Απλώς δεν μπορούμε να πούμε ότι στο εξή θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια, ούτε να με τα σχήρας μας γιατί είναι ε, θέμα του Συμβουλίου, γιατί και εμείς είμαστε συνομοθέτες και έχουμε και εμείς ένα τμήμα ευθύνης και συνυπευθυνότητας στα μάτια των εκλογέων μας και ιδίως των γαλακτοπαραγωγών που αντιμετωπίζουν τέτοιες δυσκολίες. Γι' αυτό κύριε Πρόεδρε θα σταματήσω εδώ και προσμένω τη συμβολή των εμπειρογνωμόνων που προέρχονται από πολλά μέρη της Ευρώπης και ανυπομονώ να τους ακούσω. πολύ καλή πρόταση. Να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες και μετά να θέσουμε τα ερωτήματα. Μ' αρέσει αυτή η πρόταση του κυρίου Νίκολσον. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες με τη σειρά. Πριν όμως από αυτό, ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας για την Κόπα Κοντζέκα, ο κύριος Μάνζελ Ρεϊμό, να μας κάνει μια εισήγηση. Ορίστε και παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο σας. Πρόεδρε, μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να σας απευθυνθώ. Το γάλα είναι ένα θέμα που μου είναι προσφυλές και νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για σας. Έχω εργαστεί σε γαλακτοπαραγωγικό αγρόκτημα στην Ουαλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτή τη στιγμή ο γιος μου και ο ανιψιός μου θα ακολουθήσουν την ίδια καριέρα. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαι πρόεδρος του Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΟΠΑ ΚΟΖΕΚΑ για το γάλα όπου συγκεντρώνονται γαλακτοκομικές, ε, γαλακτοκομικές συνεταιρισμοί από όλα τα κάτι μέλη. Περίπου 7.500 γαλακτοκομικά αγροκτήματα, γαλακτοπαραγωγικά αγροκτήματα από τα πλέον πολυπληθή σημεία μέχρι τις πιο ορεινές περιοχές της ε, Ευρώπης. Είναι μεγάλες οι προκλήσεις για το γαλακτοκομικό τομέα και είναι βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποκλήσεις. Πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα μπορεί να παρουσιαστούν ευκαιρίες, αλλά βράχυπρόθεσμα βλέπουμε δυσκολίες από την πίεση της κοινή αγοράς. Αυτό έχει σωρευτικό αντίκτυπο στο διεθνές ε, σκηνικό με σημαντικές γεωπολιτικές αποφάσεις και την προσωρινή έξοδο της Κίνας από την αγορά. Η, η μείωση των τιμών στην αγορά έχουν πλήξει όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παγκοσμίω έχουν φέρει αλλαγέ. Ωστόσο, το γεγονό ότι δεν έχει πλέον αγορά εξαγωγών η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, με μείωση 13,4% προ την αξία, αυτό έχει σοβαρές ε, συνέπειες και εσωτερικώ όταν μιλάμε για έμεσες ή άμεσες συνέπειες από την λειτουργία του γαλακτοπαραγωγικού τομέα και της αλυσίδας του με πιέσεις που ασκούνται καθημερινά στους παραγωγούς από τη μια και την άλλη άκρη αυτής της αλυσίδας παραγωγής. Σήμερα βλέπουμε μείωση των τιμών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με τους ε, γαλακτοπαραγωγούς, ιδίως στις χώρες κοντά στη Ρωσία, να έχουν πληγεί ιδιαίτερος. Ήδη έχουν ε, επιχειρηθεί κάποια βήματα, κάποιες λύσεις για να αντιμετωπιστεί η πίεση της αγοράς με κάποια εργαλεία της κοινή αγροτικής πολιτικής στην περίπτωση που πιέζεται η αγορά. Η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς αυτό ήταν λοιπόν ευπρόσδεκτη, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Και ακόμη υπάρχουν κίνδυνοι. Η εσωτερική αγορά μπορεί να φτάσει σε τόσο χαμηλά επίπεδα τιμών που θα φτάσουν τα, ακριβώς τα επίπεδα παρέμβασης. 274, 217 ε, λεπτά τον τόνο σε ισοδύναμα γάλακτος. Το κόστος λοιπόν έχει αυξηθεί ε, τον τελευταίο χρόνο, ε, αλλά το σταθερό κόστος είναι αυτό που έχει αυξηθεί περισσότερο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η εσωτερική αγορά λειτουργεί σωστά δεδομένη τη συνολική κατάσταση. Οι γαλακτοπαραγωγοί θα πρέπει να έχουν ε, πραγματικά κέρδη από την αγορά για να καλύπτεται το κόστο παραγωγή και να μπορέσουν να ε, συνεχίσουν την ανάπτυξη των επιχειρηματικών των δραστηριοτήτων. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η μεγάλη ε, αβεβαιότητα στην αγορά και στις τιμές και η αβεβαιότητα των παραγωγών για αυτή την αγορά, η καλύτερη λειτουργία της αλυσίδας παραγωγής γάλακτος και η διασφάλιση των γαλακτοπαραγωγών, επίσης όλες οι φάσεις της παραγωγής από την παραγωγή γάλακτος μέχρι την επεξεργασία των προϊόντων, εφόσον όλα αυτά διατηρηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή είναι η πραγματική πρόκληση για τον γαλακτοπαραγωγικό τομέα και εκεί θα πρέπει να βρούμε απαντήσεις μετά την ε, λήξη του συστήματος των ποσοστώσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες. Τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την ζήτηση για γάλα παγκοσμίω που αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,1% μέχρι το 2024. Πρέπει λοιπόν να δράξουμε αυτή την ευκαιρία για τους γαλακτοπαραγωγούς και πρέπει να επενδύσουμε σε υποδομές για να είναι πιο αποτελεσματική, πιο ανταγωνιστική παραγωγή γάλακτος. Εμείς λοιπόν στην ΚΟΠΑ αναζητούμε περιθώρια ευελιξίας όπως ε, στην περίπτωση των προστήμων και των ε, δασμών που θα επιβληθούν σε κάποια κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσουν το κόστος αυτό μέσα σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Η γαλακτοπαραγωγική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πλέον έρθει πολύ κοντά στη διεθνή αγορά. Έχει, είναι εκτεθειμένη στις παγκόσμιες τιμές και στη μεγάλη αυτή αβεβαιότητα των τιμών. Επειδή λοιπόν υπάρχει τέτοια μεγάλη διακύμανση στις τιμές και επειδή υπάρχουν διεθνείς παράγοντες πλέον που καθορίζουν την αγορά, υπάρχουν και περιορισμοί στην παραγωγή που δεν αρκούν πλέον. Δεν είναι επίκαιροι σε αυτή την παγκοσμιοποιημένη αγορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν καθαρός εξαγωγέας γαλακτοκομικών προϊόντων επί δεκαετίες. Με τον διεθνή ανταγωνισμό πλέον ως δεδομένο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ένας μεγάλος πρωταγωνιστής στη διεθνή αγορά. Σήμερα έχουμε ήδη κάποια μέτρα που μπορούν να προστατεύσουν τους γαλακτοπαραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις συνέπειες της μεγάλης αυτής διακύμανσης των τιμών στην παγκόσμια αγορά. Προς στιγμήν όμως δεν έχουν προστατευτεί αρκετά οι γαλακτοπαραγωγοί. Ίσως χρειάζονται περισσότερα μέτρα για να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσκολίες και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι εθελοντικού χαρακτήρα για τους γαλακτοπαραγωγούς. Τα μέτρα αυτά, το δίκτυο ασφαλείας με την δημόσια παρέμβαση και την ιδιωτική αποθηκεύση θα πρέπει να γίνει αποτελεσματικότερο και πιο ε, εύστοχο με την αλλαγή στα επίπεδα των τιμών παρέμβασης και τα διάφορα ανώφλια δίκτυα, τα δίκτυα ασφαλείας που ισχύουν αυτή τη στιγμή για τον παραγωγικό τομέα δεν αρκούν για να προστατεύσουν τους γαλακτοπαραγωγούς σε στιγμές κρίσης ή δυσχεριών, όπως τώρα με την αύξηση του κόστους παραγωγής. Επίσης, χρειάζονται πιο στοχευμένες αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένου του περιφερειακού επίπεδου, εφόσον χρειαστεί. Εδώ θα πρέπει να δούμε κατά πόσον τα ανώφλια και τα όρια μπορεί να πρέπει να ισχύουν αναπεριοχή και αναπεριφέρεια εφόσον υπάρχει ανάγκη. Επίσης, οι εξαγωγές επιστροφές είναι ένα, ένα εργαλείο που θα πρέπει να αποτελεί την τελευταία λύση και το Ταμείο για την Αντιμετώπιση της Κρίσης με την διακοπή των άμεσων ενισχύσεων προς τους γαλακτοπαραγωγούς θα πρέπει να είναι μια από τις τελευταίες λύσεις. Όμως αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνθήκες κρίσης και δεδομένη τη ε, ακραία διακύμαση των τιμών στο γαλακτοπαραγωγικό τομέα, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται δυναμικό εργαλείο για τι εξαγωγέ, για την ενίσχυση των εξαγωγών που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί όποτε χρειάζεται. Υπ' αυτήν την προοπτική, η εναλλακτική των ε, ασφαλίσεων των εξαγωγικών πιστώσεων στην περίπτωση των επιστροφών από τις εξαγωγές είναι κάτι που θα πρέπει να διερευνηθεί και από οικονομικής πλευράς για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να προσελκύσουμε και νέες αγορές σε μέρη του κόσμου που τώρα ε, βρίσκονται σε συνθήκες μεγάλης αβεβαιότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται επιπλέον να αναζητήσει εργαλεία αντιμετώπιση του κινδύνου, όπω το τι ε, μορφή θα πάρει η μελλοντική αγορά ή τι σταθερέ συμβάσει που αυτή τη στιγμή δεν διατίθεται τόσο πολύ και είναι εναλλακτικέ λύσει για του γαλακτοπαραγωγού. Τελικώ δεν χρησιμοποιούνται ε, σε, ε, για να αντικαταστήσουν το δίκτυο ασφαλεία. Το δίκτυο ασφαλεία λοιπόν <clears throat> έχει εμποδίσει την κατάρρευση τη Ευρωπαϊκή Αγορά και την πτώχευση κάποιων γαλακτοπαραγωγών, όμω θα πρέπει να υπάρχουν και άλλε ελλακτικέ λύσει για να αντιμετωπίσουμε του κινδύνου. Οι συνεταιρισμοί γαλακτοπαραγωγών έχουν καθοριστικό ρόλο στην μείωση τη ε, μεγάλη διακύμανση των τιμών στην αγορά για τα, για τα, μέλη, για τα μέλη των συνεταιρισμών. Και ανάλογε συζητήσει υπάρχουν και σε άλλη μέρη του κόσμου, όπου η κατάσταση είναι πολύ πιο προχωρημένη, όπω στη Νέα Ζηλανδία, όπου υπάρχουν ε, σταθερές συμβάσει, ή στι Ηνωμένε Πολιτείε, που υπάρχει ασφαλιστική πολιτική. Πέραν της διακύμανσης των τιμών που προκαλείται από εξωτερικούς παράγοντες, η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα πρέπει να διερευνήσει τη λειτουργία της ε, γαλακτοκομικής αλυσίδας παραγωγής. Η γαλακτοπαραγωγή είναι ο πιο αδύναμος κρίκος αυτής της αλυσίδας. Πρέπει να αντιμετωπίσουν την πρόσθετη πίεση λόγω ε, των αναταράξεων αυτής της ε, περίοδου. Η κόπα Κοζέκα ασχολείται με την πλήρη υλοποίηση του γαλακτοκομικού πακέτου της μέτρων ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή αυτή βρίσκεται ακόμη στα προκαταρκτικά στάδια. Υπάρχουν πολλέ νέε διατάξει που θα πρέπει να εφαρμοστούν. Όμω, ήδη τα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι το πακέτο αυτό, η δέσμη αυτή, έχει βελτιώσει τι εξειδικευμένε συμβάσει που σκοπό έχουν την, ε, να αντιμετωπίσουν, να καλύψουν τι ανάγκε των δομών των ενώσεων γαλακτοπαραγωγών και να αυξηθεί η αγοραστική δύναμη των επιμέρους παραγωγών. Αυτό πρέπει να συνεχιστεί ως προσπάθεια και ή δυνατόν να βελτιωθεί. Επιπλέον πρέπει να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία της αλυσίδας παραγωγής γάλακτος που συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του γαλακτοκομικού πακέτου. Ο μεγάλος φόβος των παραγωγών είναι η μείωση των τιμών και οι ε, καταχρήσει στην περίπτωση πώληση προϊόντων. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρεμβαίνει και να επιβάλλει πρόστιμα σε περίπτωση τέτοιων εμπορικών πρακτικών. Για τους λιανοπολιτές και τους ε, πολιτές χονδρικής πρέπει να ε, αναλογεί μεγαλύτερη ευθύνη από ό,τι για τους ίδιους τους γαλακτοπαραγωγούς. Επίσης, διαφανείς πληροφορίες για όλη την αλυσίδα παραγωγής γάλακτος θα πρέπει να ισχύει με ένα παρατηρητήριο για τον τομέα αυτό. Θα χρειαστούμε περισσότερες πληροφορίες που να είναι ευθυγραμμισμένες ώστε να μπορούμε να καταλαβαίνουμε ανα πάσα στιγμή γιατί υπάρχουν αναταράξεις την αγορά του γάλακτος. Επίσης η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση χρειάζεται μια σαφή στρατηγική για να μελετήσει την κατανάλωση των προϊόντων γάλακτος από τα πρώτα στάδια της ζωής. Ο γαλακτοκομικός ε, τομέας χρειάζεται εργαλεία προώθησης με την ανάλογη στήριξη από τον προπολογισμό και λιγότερο διοικητικό άχθος. Εφόσον ισχύσουν όλε αυτέ οι προποθέσει ταυτόχρονα, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η επεξεργασία γαλακτοκομικών προϊόντων και η παραγωγή του θα παραμείνει ένα ζωτικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια πρόκληση που αφορά όλους μας για το μέλλον του γαλακτοκομικού τομέα. Ευχαριστώ για την προσοχή σα και είμαι στη διάθεσή σα για ερωτήσει. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι όλοι οι ομιλητές έχουν 10 λεπτά ο καθένας και μετά τα 9 λεπτά θα σας κάνω κάποιο νόημα. Λοιπόν, τώρα η κυρία Ιζαμπέλ Βιλάλμπα Σεϊμπάν που είναι γαλακτοπαραγωγός από την Καλήθεια και πρόεδρος της Βία Καμπεσίνα με την ομάδα πολιτικού διαλόγου για τα γαλακτοκομικά. Έχετε το λόγο. Καταρχάς ευχαριστώ την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξη Πέτσων για τη δυνατότητα που μου δίνει να ακουστεί εδώ η φωνή των παραγωγών, ανδρών και γυναικών και να αναλύσουμε τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας μιλήσω για τους στόχους αυτού του πακέτου για το γάλα για να δούμε εάν είναι χρήσιμα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Μετά τη βαθιά κρίση του 2009 ο στόχος μας είναι να έχουμε τα αναγκαία μέσα για να αποφύγουμε μελλοντικές κρίσεις, χαμηλές τιμές και να ενισχύσουμε τις δυνατότητες ε, των παραγωγών, την εξουσία των παραγωγών και τις συνθήκες ζωής που ε, να αποφύγουμε τις συνθήκες ζωής που επιβάλλουν οι χαμηλές τιμές και να αποφύγουμε την κυρίαρχη θέση των μεγάλων σούπερ μάρκετ που υποβάλλουν ε, τέτοιες χαμηλές τιμές που έχουν επιπτώσεις στους παραγωγούς. Να βελτιώσουμε λοιπόν το εισόδημα των ε, παραγωγών, να ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία του κόστους παραγωγής, να υπάρξει σταθερότητα, ούτως ώστε να έχει βιώσιμο μέλλον ο κλάδος. Να αποφύγουμε τις μεγάλες ανισορροπίες. Αυτή είναι η στόχη του πακέτου γάλα και έτσι δημιουργήθηκε. Μετά από τρία χρόνια εφαρμογή τι βλέπουμε. Πρώτον, σε σχέση με τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, καμία αλλαγή. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, οι μεγάλοι διανομή, δεν επηρεάστηκαν καθόλου. Τα συμβόλαια που υπεγράφησαν κυρίως είχαν επιπτώσει στους παραγωγού Η ισχύ, η κυρίαρχη θέση των μεγάλων σούπερ μάρκετ δεν έχει αλλάξει καθόλου από το 2009. Οι δυσλειτουργίες και ανισορροπίες στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι παρόμοιες. Κανείς δεν υποχρεώνει κανέναν να λάβει υπόψη το πραγματικό κόστος παραγωγής και δεν υπάρχουν και ουσιαστικές κυρώσεις. που να τιμωρούν αυτούς που υποχρεώνουν τους παραγωγούς να πολλούν το γάλα τους κάτω του κόστου. Επίσης, το πακέτο αυτό που στην ουσία ήταν η ιδιωτικοποίηση της πολιτικής γαλακτοκομικών αγνόησε σε μεγάλο βαθμό τους Ευρωπαίους παραγωγούς. Ε, υπήρχε μία δυνατότητα για τους συνεταιρισμούς που δεν ήταν υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν στις λογικές διαπραγματεύσεις ούτε σε οργανώσεις παραγωγών. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης οι συνεταιρισμοί συλλέγουν το 90% του γάλακτος. Να τους εξαιρέσουμε λοιπόν τι αποτελεσματικότητα αφήνει στο πακέτο γάλακτος, διότι εξαιρούμε τεράστιες περιοχές και ένα μεγάλο αριθμό παραγωγών. Η εκτίμηση που κάνει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έκανε στις 13 Ιουνίου 2014, καθιστά σαφές ότι μόνο σε τέσσερα κράτη-μέλη, Γερμανία, Τσεχία, Ισπανία, Γαλλία, υπήρξαν κάποιου τύπου διαπραγματεύσεις με συμμετοχή των οργανώσεων παραγωγών. Να σας πω τι έγινε στην Ισπανία. Έχουμε 7 ε, αναγνωρισμένες ε, οργανώσεις παραγωγών στον τομέα αλλά δεν απέκτησαν ποτέ ουσιαστικές δυνατότητες η παραγωγή διαπραγματεύσεων. Ούτε είχε αυτό καμία επίπτωση ουσιώδη στις τιμές. διότι οι οργανώσει αυτές καλύπτουν λιγότερο από το 1 τρίτο τη παραγωγή Συμπέρασμα. Δεν ενισχύθηκε η πραγματική διαπραγματευτική θέση των παραγωγών. Εξακολουθούν τεράστιες ανισορροπίε ε, δυνάμεων μεταξύ των παραγωγών και των μεγάλων πολυεθνικών όπως Λακτάλη, Άρδα, Καμπίνα. Αυτοί απέχουν χιλιάδε χιλιόμετρα από του παραγωγού και ασχολούνται με πολύ γενικότερες ε, παραμέτρους της κατάστασης αγοράς από ό,τι μικρή παραγωγή. Είχαμε κάποιες, ε, κάποιους δείκτες ε, όπου συμφώνησαν όλες οι επαγγελματικές οργανώσεις, αλλά κατόπιν δεν έγιναν σεβαστοί οι δείκτες αυτές. Οι δείκτες αυτοί από τους μεγάλους οργανισμούς ε, διανομής. Αυτές λοιπόν οι οργανώσεις είτε υποχρεωτικές είτε εθελούσιες δεν βοηθούν. Οι μεγάλοι διανομής επιβάλλουν τους όρους τους. Αν είμαι υποχρεώσει λοιπόν να υπογράψω μια, ένα συμβόλαιο ε, όπου είμαι υποχρεωμένος, ε, υποχρεωμένη να δέχομαι τιμή ε, πώληση χαμηλότερη από το κόστος τότε με πιέζουν υπερβολικά και δεν βελτιώνεται καθόλου η κατάσταση των παραγωγών. Δεν υπάρχει υποχρέωση υπογραφής συμβολέων από τους διανομής και αυτό το αξιοποιεί η διανομή. Μας επιβάλλουν τιμές που μας καταστρέφουν σε πολλές περιπτώσεις. Και τι πήρε είχαμε και με τα συμβόλαια. είναι διαφορετικών διαστάσεων και πολλές φορές ε, ο μηχανισμός αυτός ε, στρεβλώνεται. Έχουμε συμβόλαια για ένα μήνα πολλές φορές. Μας επιβάλλουν τιμές και συνθήκες και προδιαγραφές ποιότητας που είναι χαμηλότερες από αυτά που έχουν συμφωνηθεί από τις δημόσιες αρχές. Δεν υπάρχει σύστημα διατησίας μεσολάβησης, άρα στην ουσία περισσότερο αυτός ο μηχανισμός ωφελεί τους διανομής. Η κατάσταση των τιμών είναι δραματική. Ούτε καν 30, 30 λεπτά. Έχουμε πολλά συμβόλαια στη χώρα μας, στην Ισπανία, αλλά οι τιμές, όπως είπα, είναι χαμηλότερες από 30 λεπτά. Άρα δεν ε, μας εξυπηρετεί. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν. Έχουμε πλεονάσματα και δεν υπάρχει επαρκής προσφορά. Άρα το πακέτο, λέτσε, το πακέτο γάλα δεν είναι αποτελεσματικό. Η κατάσταση και με τους άλλους παραγωγούς ε, Νέα Ζηλανδία, Ηνωμένε Πολιτείες Υπάρχει υπερπαραγωγή. Δεν υπάρχει επαρκή ζήτηση. Αυτό λοιπόν ε, πιέζει τις τιμές, οι οποίες πέφτουν κάτω του κόστους. Και η μόνη δυνατότητα που έχουμε είναι να πτωχεύσουν οι επιχειρήσεις για να μειωθεί η παραγωγή. Γιατί ξέρετε, όπου γίνονται αυξήσεις παραγωγής δεν είναι ομοιόμορφες. Άλλοι λένε πως είναι 12, άλλοι λένε πως είναι 5% σε επίπεδο ευρωπαϊκό, αλλά είναι πολύ άνηση η αύξηση. Σε κάποιες περιοχές που υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση θα έχουμε πολλά ζώα, σε άλλες θα εξαφανιστούν. Οπότε η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν κάνει μια αποτίμηση των επιπτώσεων που θα έχουν για τις μειονευτικές περιοχές αυτές οι καταστάσεις και για την απασχόληση και γενικά για την οικονομική και κοινωνική δομή των περιοχών αυτών. και δεν γίνεται καμία ανάλυση για το πόσα γαλακτοκομικά αγροκτήματα θα εξαφανιστούν. Δεν είναι δυνατόν να μα λένε ότι η μόνη δυνατότητα που έχετε είναι να βάλετε λουκέτο. Ο μόνο μηχανισμό για να ε, μειωθεί η προσφορά. Και οι δυνατότητε διαμεσολάβηση είναι πολύ ε, περιορισμένε, πολύ λίγο αξιοποιούνται. Οπότε, έχουμε μια διαδικασία συγκέντρωση παραγωγή σε συγκεκριμένε περιοχέ με όλα τα προβλήματα που προκαλεί αυτό η υψηλή συγκέντρωση για παράδειγμα νητρικών και η μόνη δυνατότητα που έχουμε είναι μια δημόσια πολιτική ελέγχου της παραγωγής και διαχείρισης των αγορών. Να ληφθεί υπόψη όχι μόνο η παραγωγή αλλά και ο τρόπος παραγωγής. Δεν μιλάμε πολύ για την εσωτερική αγορά. Πάνω από 90% της ευρωπαϊκής παραγωγής ε, καταναλώνεται εσωτερικά. Και γιατί μειώνεται ε, η, κατανάλωση, υπάρχουν προβλήματα με τη λακτόζη, με, τα, με την αντίσταση σε αντιβιωτικά. Αυτά δημιουργούν προβλήματα γενικότερα στην ε, ευρωπαϊκή κτηνοτροφία και ευρύτερα. Όλα αυτά έχουν επιπτώσει στην ε, υγεία. Οπότε μειώνεται η κατανάλωση για τέτοια προβλήματα, όπως υπάρχουν και οι αφλατοξίνες. Οπότε η εσωτερική κατανάλωση πρέπει να αξιοποιηθεί περισσότερο. Να μην υπάρχει τέτοια έκθεση σε αυτήν την ε, παγκόσμια αγορά που έχει τόσο χαμηλές τιμές και ε, ισχυρές διακυμάνσεις τιμών. Σας ευχαριστώ. γιατί επιδείξατε και την απαραίτητη πειθαρχία και σεβαστήκατε το χρόνο σας. Θεωρώ ο κύριος Ντάνκαν Μαν Άγγλος γαλακτοπαραγωγός. Λέγομαι όπως ακούσατε Duncan Mann. Είμαι τρίτης γενεάς γαλακτοπαραγωγός από την Κούμπρια, από την Ουαλία. Το αγρόκτημά μου έχει 106 εκτάρια και 20 από αυτά είναι καλλιεργήσιμα. Το 2007 έλειφε η απόφαση να σταματήσουμε την καλακτοπαραγωγή και να πουλήσουμε το κοπάδι μας, αλλά μετά από τρία χρόνια αποφάσισα να ξαναρχίσω την γαλακτοπαραγωγή. Μέσω διεθνών και τοπικών αγορών γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων μπόρεσα να μαζέψω 240 αγελάδες από το 2012 όμως χρειάστηκε να τις μειώσω και πάλι γιατί ξέσπασε μία επιζωτία και το τέλος του 2014 μου έμειναν πολύ λίγες. Παρ' όλα αυτά ξανααποφάσισα να επιστρέψω στη γαλακτοπαραγωγή παρά τη ζημιά που μου επέβαλε το μικόπλασμα, μικόπλασμα Μπόβης. Απευθύνθηκα σε ένα συνεταιρισμό γαλακτοπαραγωγών που χρηματοδοτεί όχι με τον όγκο της παραγωγής αλλά αναγρόκτημα και έτσι μπόρεσα να έχω κάποιο εισόδημα. 0,47 πένες πληρώνομαι για κάθε πρόσθετο 0,1% πρωτεϊνών στην παραγωγή του γάλακτος. Και αυτό το φροντίζω μέσω πολύ προσεκτικής επιλογής. Έτσι έχω μεγαλύτερο έλεγχο στο εισόδημά μου. Το έψαμε την Εστλέ. Ήταν ουσιώδες για να μπορέσω να επιβιώσω. Αυτή τη φορά θα ξαναγοράσω αγελάδες αλλά από κάποια άλλη ποικιλία που παράγει περισσότερες πρωτεΐνες γιατί μάθαμε πολλά μαθήματα από την εμπειρία μας με την επιζωτία μικρόπλασμα μπόβης και έτσι αυξήσαμε την βιοασφάλεια του αγροκτήματός μας. Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη αν δεν μας είχε βοηθήσει ένας αγοραστής που ενδιαφέρεται για την εχλαισιμότητα και την ποιότητα του προϊόντος. Στο Ηνωμένο Βασίλειο απαιτείται να εφαρμόζεται ένας εθελοντικός κώδικας Αυτό είχε λειτουργήσει σωστά, αλλά αυτή τη στιγμή η οργάνωση αυτή, η περιοχή μου μάλλον, υποφέρει εκ νέου γιατί δεν υπάρχουν πια συμβόλαια. Ο τρόπος λειτουργίας του συμβολέμου με την Εστλέ νομίζω είναι καλό πρότυπο. Οι γεωργοί επενδύουν στην επιχείρησή τους, είτε είναι μεγάλη είτε μικρή, αν έχουν την εμπιστοσύνη ότι θα υπάρχει κάποιο εισόδημα. Η επένδυση δεν αυξάνεται απλώς μέσω μεγαλύτερης παραγωγής, αλλά μπορεί να αυξηθεί λόγω περισσότερης αποτελεσματικότητας ή καλύτερης ποιότητας γάλακτος ή καλύτερης τεχνολογίας. Μια τιμή παρέμβασης δεν στηρίζει τέτοιου είδους επενδύσεις, αλλά μόνο τη στήριξη περισσότερου γάλακτος, μεγαλύτερης παραγωγής γάλακτος στηρίζει. Όπως ξέρουμε το σύστημα των επιχορηγήσεων δεν ισχύει πια και μόνο εταιρείε σαν τη Λεστλέ που αρχίζουν να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την, ε, το σύστημα μπορούν να επιβιώσουν. Νομίζω ότι η μικροπαραγωγή και οι καταναλωτές γάλακτος είναι σε καλύτερη θέση τώρα για να στηρίξουν τα εισοδήματα των γαλακτοπαραγωγών. Φροντίζοντα περισσότερο τη διαδικασία παραγωγής Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια ασφάλεια της ε, προμήθειας, της παραγωγής και ενδιαφερόμαστε όλο και περισσότερο και για θέματα περιβαλλοντολογικά όπως την μείωση του ρυθμού παραγωγής αερίων με εφέ θερμοκηπίου. Προ η διανομή στο Ηνωμένο Βασίλειο υποτιμούν πολύ τα γαλακτοκομικά οι τωρινές λιανικές τιμές είναι χαμηλές, 89 πένες για 4 pints, περίπου 2,2 λίτρα. Το γάλα είναι φτηνότερο αυτή τη στιγμή από ότι το νερό. Αυτό είναι απαράδεκτο αφού είναι κάτι τόσο χρήσιμο και υγιεινό για τους καταναλωτές από τις καλύτερες πηγές βιταμινών και πρωτεϊνών ασβεστίου, καλίου, φωσφόρου, ιωδίου, βιταμινών Β2, Β1 και Β12 και συνεισφέρει κατά 19% στην ε, διατροφή σε ασβέστιο των ενηλίκων. Για να έχουμε την ίδια ποσότητα ασβεστίου από άλλα τρόφιμα θα έπρεπε να τρώμε 63 λαχανάκια βρυξελών, 11 μερίδες σπανακίου και τέσσερις μερίδες μπρόκολα. Και όμως η τιμή είναι εξευτελιστική. Αυτά που κάνει η Coca-Cola αυτή τη στιγμή θα μπορούσαν να είναι υπόδειγμα. Δηλαδή οι καταναλωτές της Ένωσης είναι συνηθισμένοι να αγοράζουν γνωστά προϊόντα, γνωστές μάρκες και θα μπορούσαν επομένως οι πολυεθνικές να κάνουν κάτι παραπάνω για να επενδύσουν στη διανομή και προώθηση των γαλακτοκομικών ιδίω υψηλή ποιότητα και με τις καινούργιες ποικιλίε που χρησιμοποιούνται όπως πρόσθετα ωμέγα 3 κλπ. Πώς, πώς. Δεν είναι δυνατόν να μας κάνει ένας ομιλητής διαφήμιση για την Εθλέ και την Coca-Cola. Είμαστε κοινοβούλιο. Δεν είναι ε, διαφημιστική εκδήλωση εδώ. Είναι απόλυτα παράδειγμα να γίνονται αυτά τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο αυτό, αλλά παρακαλώ τον ομιλητή να συνεχίσει ο ομιλητής Κοιτάξτε, ο μιλητής αυτός λέει τι κάνει για να επιβιώσει. Αυτό πρέπει να ακούσουμε. Τα ονόματα είναι άσχετα. Τα έδωσε των εταιριών για να μας δείξει τι ακριβώς κάνει για να παραμείνει ενεργός. Αυτά πρέπει να πάρουμε ως μαθήματα. Ναι, ναι, θα τον ακούσουμε, θα τον ακούσουμε. Συνεχίζει. Η μεγαλύτερη προώθηση των γαλακτοκομικών θα σημαίνει ότι και οι διανομής θα έχουν καλύτερη προμήθειες και θα μπορούν να επενδύσουν και αυτοί με πρόσθετα ωφέλη ώστε οι αγρότες, οι παραγωγοί να μπορούν να πληρώνονται δικαιότερη τιμή και να μπορούν να επενδύσουν. Παραδείγματος χάρη, εμείς συνεργαζόμαστε με την ΕΣΤΛΕ για να παρακολουθούμε και πώς τι εκπομπές αερίων δημιουργούνται από την παραγωγή μας. Δεν πιστεύω ότι οι ε, αγρότες που συνεργάζονται σε συνεταιρισμούς θα μπορέσουν να πουλήσουν περισσότερο τα γαλακτογμικά τους προϊόντα. Έχουμε μεγάλη ιστορία και παρελθόν συνεργατισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά ακόμη και με τις συνεδερισμούς η ποιότητα είναι αυτή που λείπει από την γαλακτοκοπική αγορά. Οι αγρότες στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη παλαιότερα στο Milk Marketing Board και υπήρχαν πολύ μεγάλοι συνεταιρισμοί όπως οι Dairy Farmers of Britain θα ήταν πολύ δύσκολο να συνηθίσουν ξανά οι αγρότες του Ενωμένο Βασίλειο να εμπιστεύονται τέτοιους συνεταιρισμούς και πρέπει να βρεθούν διαφορετικές λύσεις. Γίνεται πολλής λόγος αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο για το κατά πόσον θα υπάρξει μέλλον στην αγορά των γαλακτοκομικών. Υπάρχουν παραδείγματα από άλλους τομείς, αλλά θα έπρεπε να υπάρξει περισσότερη διακύμανση στο Δημονό, λιγότερη. Άλλη ιδέα είναι ένα συμβόλαιο ποσοστώσεων α συν β, όπως γίνεται με τα ζαχαρότευτλα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερο μερίδιο και ίσως και ψηλότερη τιμή για το φρέσκο γάλα. Ως παραγωγός έχω καθημερινά προβλήματα για να φροντίσω τα ζώα μου και τις ζωοτροφές μου. Δεν πιστεύω ότι πρόσθετες ευθύνες θα μπορούσαν να με βοηθήσουν αν αναλάβω πρόσθετες ευθύνες. Δεν νομίζω ότι οι παρεμβάσεις που στρεβλώνουν την αγορά ζημιώνουν τελικά τον παραγωγό και θα ήθελα να υπάρξει ένα μέλλον όπου περισσότεροι διανομής θα αναλάβουν κάποια ευθύνη και αυτή και επομένως θα επενδύσουν σε εναλλακτικά γαλακτοκομικά προϊόντα που να διασφαλίζουν ένα εισόδημα στο γεωργό και περισσότερη ασφάλεια για όλους από τον παραγωγό μέχρι τον καταναλωτή. Σας ευχαριστούμε για την δική σας ε, εμπειρία. Φαντάζομαι ότι δεν προσπαθήσατε να διαφημίσετε κάτι, αλλά να παρουσιάσετε τις θετικές πτυχές της, ε, του γαλακτοκομικού τομέα. Τώρα η κυρία Πιλάρ Ουλάουα από την Γαλλική στην Ισπανία για 10 λεπτά έχετε το λόγο.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 gdybyśmy się Państwo nie obrazili, to byśmy poprosili o pierwsze wystąpienia naszych koordynatorów. Ίσως τους συντονιστές να ζητήσουμε να μιλήσουν πρώτα και μετά μέχρι να διορθωθεί το τεχνικό πρόβλημα και να γίνει η παρουσίαση. Α, δούμε. Ο κύριος δεν ζήτησε το λόγο πρώτος, αλλά έφυγε. Έχουμε όμως τον πρόεδρο Ντεκάστρο. Μήπως εκείνος να μιλήσει τώρα. <laughs> Ευχαριστώ πρόεδρε. Ήθελα να ακούσω πρώτα τους εμπειρογνώμονες στο δεύτερο τμήμα της ακρόασης και μετά να τοποθετηθώ. Ωστόσο, επειδή μου δώσατε το λόγο, παρακαλώ. Ένα λεπτό παρακαλώ μόνο. Εντάξει, κερδίζουμε χρόνο έτσι. Με την παρέμβαση αυτή ήθελα να πω το εξή. Ακούγοντας τις πρώτες ε, σκέψεις των εμπειρογνωμόνων μας, η κατάσταση μου φαίνεται αρκετά σαφής. Ζούμε μια δύσκολη στιγμή. Μια στιγμή που έχει περισσότερο συνέπειε για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Δεν ξέρουμε εάν μακροπρόθεσμα θα αντέξουν στι χαμηλέ τιμέ. Βλέπουμε ότι η αύξηση τη παραγωγή στην Ευρώπη και νομίζω θα μα το πούν και οι μετά, μα φέρνουν στο 5% αύξηση γάλακτο το 2014 τα στοιχεία, με ε, μείωση τη κατανάλωση. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έπαιξε εδώ σίγουρα το ρόλο της. Και, αν, και σε να μην έφτανε αυτό, έχουμε και το εμπάρκο της Ρωσίας που περιόριζε τις ε, εισαγωγές ε, πολλών γαλακτοκομικών προϊόντων. Η συνδυαστική, ο συνδυαστικός αντίκτυπος αυτών των τριών στοιχείων έχουν δραματικές συνέπειες για την αγορά, φέρνοντας την τιμή του γάλακτος σε σταδιακή μείωση και σε δυσχερή θέση της επιχειρήσης. Η δουλειά του Τζιμ Νίκολσον με την ε, έκθεση που συντάσσει και ακούγοντας τις παρατηρήσεις των διάφορων συζητήσεων στο Κοινοβούλιο θα είναι να μας πει τι είδους διαχείρισης της προσφοράς μπορεί να προτείνει το Κοινοβούλιο χωρίς και το λέω με μεγάλη σαφήνεια, χωρίς να αφήσει από το παραθυράκι να ξαναμπούν οι ποσοστώσεις γάλακτος που ξέρουμε πολύ καλά ότι φεύγουν από την πόρτα κανονικά και με τον νόμο τον, την 1η Μαρτίου 2015. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι ο κύριος Νταντέν θα καθορίσει με την παρέμβασή του ε, τα θέματα αυτά, διότι με την ε, κοινή οργάνωση αγοράς και τη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής είχε κάνει μια πρόταση που όμως δεν έτυχε πλειοψηφία στο Συμβούλιο και την Επιτροπή. Τότε όμως είχε συντάξει μια πρόταση το Ευρωκοινοβούλιο που κάποια στιγμή θα πρέπει να την ξαναδούμε, ίσως προσαρμοσμένη, ε, αλλά είχαμε συντάξει επί χάρτου ένα υποθετικό σενάριο διαχείρισης της ε, προσφοράς που θα μπορούσε να είναι μια απόκριση ε, στο όλο πρόβλημα. Να είναι περισσότερο σε εναλλακτικέ που διατίθενται στου γαλακτοπαραγωγού μα και για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τι αλλαγέ στι τιμέ, όπω είδαμε και από τα γραφήματα. Οι διακυμάνσει στι τιμέ ε, εντείνονται, δεν εμβλύνονται, δεν περιορίζονται. Άρα είναι απαραίτητο νομίζω να προβλέψουμε τέτοιες προτάσεις γιατί προφανώς θα περιμένουμε βεβαίως και από τους ε, εμπειρογνώμονες κάποιες πρόσθετες ιδέες αλλά μιας και τώρα λειτουργεί ο προβλέας ας δώσουμε την... Ε, το λόγο στην εμπειρογνώμονά μας την κυρία Ολό Αλόνσο. Τρία λεπτά πρόεδρε. <laughs> Panie Przewodniczący, ma Pan wyjątkowe szczęście, bo zamiast dwie minuty mówił Pan... Είστε πολύ τυχερός, γιατί όντως ε, τρία λεπτά πήρατε αντί για δύο. Και θα έχετε κι άλλο χρόνο μιλίας μετά. Είστε πραγματικά τυχερός. Τώρα να δώσω το λόγο στην εμπειρογνωμονά μας. Ε, buenas tardes. Καλησπέρα. Ως εκπρόσωπος μιας περιφέρειας της Ευρώπης που έχει μεγάλο βάρος ε, στη γαλακτοκομική παραγωγή να σας δώσω μερικές πινελιές για το πώς έχει λειτουργήσει το πακέτο για το γάλα στην ε, περιφέρειά μου, τη Γαλλικία κατά την περίοδο εφαρμογής του μέχρι τούδε και τι προτείνουμε για βελτιώσεις για μια περιφέρεια όπως η Γαλλικία. Αυτό είναι ο χάρτης της Ευρώπης. Βλέπετε που είναι η Γαλλικία εδώ, βόρειο-ανατολική Ισπανία, βορειοδυτική συγγνώμη, όπου υπάρχουν πολλοί παραγωγοί γάλακτος, ή περισσότεροι παραγωγοί γάλακτος και μεγάλη πυκνότητα παραγωγής γάλακτος, που με βάση τα στοιχεία της Κομισιόν παράγει το περισσότερο γάλα και έχει την υψηλότερη πυκνότητα παραγωγών και στα πλαίσια της Ισπανίας, του Ισπανικού κράτους. Είμαστε η σημαντικότερη γαλακτοπαραγωγική περιοχή. 56% των παραγών στην Γαλλικία, 10.500 παραγωγή. Και έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της παραγωγής γάλακτος της Ισπανίας. 2,3 εκατομμύρια τόνους. έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε συμβατικέ σχέσει Και τα κράτη-μέλη αποφασίζουν αν θα είναι υποχρεωτικέ αυτέ οι σχέσει και ποια θα πρέπει να είναι η διάρκεια ισχύω. Έτσι έχουμε περισσότερε δυνατότητε ε, να διαπραγματευτούμε με του ε, μεταποιητέ, ούτω ώστε σε όλη την αλυσίδα να είναι πιο ισότιμε οι σχέση. Οι επαγγελματικέ οργανώσει, για να διευκρινίσουν την κατάσταση, προσπαθούν σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας να υπάρχει διαφάνεια. Αυτό επιθυμούμε όλοι. Το πακέτο έχει επιτύχει τους στόχους του στη Γαλλικία. Τίθεται η ερώτηση. Τους έχει ε, επιτύχει. Σε ένα βαθμό αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Για παράδειγμα οι συμβατικές σχέσεις. Τι αποφασίστηκε. Αποφασίστηκε να είναι υποχρεωτικές ή συμβάσεις. Υποχρεωτικά τα συμβόλαια με ελάχιστη διάρκεια ενός έτους και μόνο για τον νοπό γάλα όπως το ορίζει η κανονιστική ενωσιακή νομοθεσία. Έχουμε τρία, τρία τμήματα της ε, διατροφικής αλυσίδας. Παραγωγή, ε, αγοραστές, μεταποιητές και διανομής. Εδώ είναι διαφορετική η κατάσταση από ότι σε άλλα μέρη της Ευρώπης όπου οι παραγωγοί πουλούν απευθείας του διανομής. Έχουμε τρεις διαφορετικούς εμείς, ε, τρεις φάσεις, τρία τμήματα. Οι παραγωγοί δεν έχουν υψηλή συνειδητότητα, δεν έχουν υψηλό επίπεδο οργάνωσης, δεν κατανοούν το ρόλο που πρέπει να παίζουν για τα συμβόλαια. Οι μεταπιτέ, οι γαλακτοβιομηχανίες θεωρούν ότι με το να έχουν αιτήσια συμβόλαια έχουν δυσχέρες τις σχέσεις τους με την διανομή. Και γι' αυτό ακριβώς οι μεταπητές είναι πολύ ισχυρότερες σε σχέση με τους παραγωγούς. Τους επιβάλλουν συμβόλαια με την διάρκεια που επιθυμούν. Εμείς θα θέλαμε ε, όλα τα συμβόλαια να είναι αιτήσια και για την παραγωγή και για τη μεταποίηση και τη διανομή. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Η διαπραγματευτική ισχύ είναι πολύ σημαντική. Οι παραγωγοί πρέπει να μπορούν να διαπραγματευτούν με τους μεταποιητές, με τις βιομηχανίες. Όπως πόθηκε προηγουμένως, οργανώσεις παραγωγών που παίζουν βασικό ρόλο στην Γαλλικία εκπροσωπούν το 35% της παραγωγής αλλά δεν μπόρεσαν να παίξουν το ρόλο τους. Γιατί θα έπρεπε να μπορούν να διαπροτευτούν για όλα τα συμβόλαια. Τα δικαιώματα των παραγωγών περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να καταγγείλει κάποιο συμβόλαιο. Αυτός είναι ένας όρος όμως που μειώνει τη σταθερότητα των συμβολέων αυτών μακροπρόθεσμα. Τι συμβαίνει δηλαδή. Η τιμή του γάλακτος καθορίζεται από τα συμβόλαια. Ούτε η παραγωγή, ούτε οι βιομηχανίες δεν θέλουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια που να βασίζονται σε δείκτες για το καθορισμό της τιμής. Σε τι βαθμό επιτύχαμε τους στόχους μας. Συζητούμε με τις επαγγελματικέ οργανώσεις όπως η INLAX στην Ισπανία και θα έπρεπε να εκπροσωπείται, γιατί δεν εκπροσωπείται και ο τομέας της διανομής. Όλα τα τμήματα της αλυσίδας θα έπρεπε να μπορούν να συζητήσουν γύρω από ένα τραπέζι για να ενισχυθεί ο τομέας για το μέλλον. Η διαφάνεια θεωρούμε ότι είναι σημαντική, οπότε θεωρούμε ότι το παρατηρητήριο γάλακτό, το ευρωπαϊκό, παίζει ζωτικό ρόλο, το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο, ε, που μπορεί να βοηθήσει τη λήψη αποφάσεων και από τους παραγωγούς και από τη βιομηχανία και από τη διανομή. Από όλο τον τομέα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πληροφόρηση που μας δίδεται. Αλλά θεωρούμε ότι θέλουμε να έχουμε πληροφορίες όχι μόνο σε επίπεδο κρατών αλλά και σε επίπεδο περιφερειών από το παρατηρητήριο. Οπότε η Γαλλικία προτείνει να έχουμε στοιχεία για επίπεδα παραγωγής και τιμές σε επίπεδο περιφερειών. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να βασίζονται βέβαια στον ε, προκαθορισμένο ορισμό για το τι είναι γάλα. Η συνεργασία μεταξύ παραγωγών και γαλακτοβιομηχανιών είναι θεμελιώδης. Όπως είπα, ένα μεγάλο τμήμα του γάλακτος στη Γαλλικία παράγεται από παραγωγούς που δεν είναι συνδικαλισμένοι, ούτε πολύ μεγάλοι. Μόνο 20% του γάλακτος στη Γαλλικία παράγεται από συνεταιρισμούς, οπότε η συνεργασία μεταξύ παραγωγών και μεταπητών είναι πολύ σημαντική. Αλλά είναι περίπλοκη αυτή η πρόκληση. Γιατί δεν έχουμε επαρκές επίπεδο οργάνωσης στη Γαλλικία. Πρέπει να ανέβει το επίπεδο συμμετοχής στους συνεταιρισμούς. Η παραγωγή, όπως είπα, είναι το πιο αδύναμο τμήμα της αλυσίδα. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί η θέση τους. Όπως είπα, δεν θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ε, διακοπής των συμβολέων που έχουν υπογραφεί για ένα χρόνο. Γιατί αυτό το αξιοποιούν οι βιομηχανίες σε πολλές περιπτώσεις. Ει βάρο των παραγωγών. Και μια άλλη πρόταση, να απαγορεύεται. Αν ένας παραγωγός ανήκει σε οργάνωση παραγωγών να μην μπορεί να διαπραγματευτεί από μόνο του την πώληση γάλακτος τη γαλακτοβιομηχανία. Θα πρέπει να περνάει από το συνεταιρισμό του. Το πακέτο αυτό είναι χρήσιμο και αναγκαίο για μειονεκτικέ περιοχέ όπω η Γαλλικία, αλλά όπω είπα μπορεί να βελτιωθεί και επειδή επίκειται η λήξη των ποσοστώσεων είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτές τις βελτιώσεις ζωτικής σημασίας, όπως ήδη υπόθηκε, είναι να έχουμε και άλλους μηχανισμούς στήριξης, όπως είναι οι βοήθειες μέσω των ε, απευθείας πληρωμών και οι επιδοτήσεις για την ανάπτυξη της πέτρου για περιοχές που έχουν ειδικά ναι, ναι, ναι. χαρακτηριστικά. Α, με συγχωρείτε, να δω σε, σε ποια διαφάνεια πρέπει να πάω. Ε, ε, Πώ ah, Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το πακέτο για περιοχές όπως η Γαλλικία το παρατηρητήριο να μας δίνει στοιχεία για σε επίπεδο περιφέρειας με βάση τον στάνταρ ορισμό του γάλακτος να μην μπορεί ο παραγωγός να καταγγείλει το συμβόλαιο που πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα χρόνο και οι πολιτές να μην μπορούν να πουλήσουν απευθείας ε, την παραγωγή τους αν συμμετέχουν στο οργάνωση παραγωγών και να συμπεριληφθεί ο τομέας της διανομής στις ε, διεπαγγελματικέ οργανώσεις και άλλες πολιτικές. Να αυξηθεί η τιμή παρέμβαση για τα γαλακτοκομικά, να υπάρχουν μηχανισμοί για την προστασία των περιθωρίων, να συμμετέχουν οι παραγωγοί σε οργανώσεις που να είναι σε θέση να μεταπίσουν το γάλα, ούτω ώστε να μειώσουμε τον αριθμό διαδικασιών, να πολλούν περισσότερο γάλα οι συνεταιρισμοί, όλα τα συμβόλαια σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας εφοδιασμού να είναι τουλάχιστον ενός έτους, να υπάρξουν ανανεώσεις, να μειώσουμε το κόστος παραγωγής, να προωθήσουμε την εσωτερική κατανάλωση και οι ετικέτες να δίνουν σωστή πληροφόρηση και να μην μπορούν οι διανομείς να αξιοποιήσουν ε, το, προϊόν του, το γάλα και τα προϊόντα ω ειδικέ προσφορές κάτω του κόστου για να προσελκύσουν ε, πελάτες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ποιο από τους συντονιστές θα ήθελε τώρα να πάρει το λόγο σε αυτόν τον γύρο και ποιο στο δεύτερο. Κύριε Ντες. Δύο λεπτά για κάθε συντονιστή και ένα λεπτό για λοιπούς βουλευτάς. Ο κύριος Ντες με αργότερα. Σάντα. Ευχαριστώ. Καταρχάς, ο γαλακτοκομικός τομέας είναι τομέας όπου διακυβεύονται πολλά. Είναι θέματα διατροφής, απασχόλησης και ανάπτυξης της υπαίθρου. Είναι σαφές ότι η αποτυχία των μέτρων που έχουν ληφθεί για τα γαλακτοκομικά είναι γνωστή. Και επίσης ε, χώρες όπως η Ελβετία εγκατέλειψαν τις, τους μηχανισμούς ελέγχου της παραγωγής και αυτό είχε επιπτώσεις. Οπότε πρέπει να σκεφτούμε σε βάθος σε αυτή τη συγκυρία τι θα κάνουμε στο μέλλον. Για μένα ειλικρινά δεν θεωρώ ότι είναι αποδεκτό να λέγεται όπως είπε ο εκπρόσωπος της ΚΟΠΑ να λέει ότι έχουμε τεράστιες δυνατότητε ε, στη διεθνή αγορά και να ζητάει τώρα μέτρα στήριξης της παραγωγής, των εξαγωγών. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εάν μας δίνει τόση δυνατότητα η διεθνής αγορά και όλοι ε, εγκομιάζουν τη φιλελευθεροποίηση, τότε γιατί χρειάζονται ε, δημόσιες πολιτικές για να ευνοήσουμε τις εξαγωγές. Πρέπει να στρέψουμε την ε, προσοχή μας στην εσωτερική κατανάλωση, να διατηρήσουμε τα συστήματα προογής, να υπάρχουν μηχανισμοί που να επιτρέπουν στους παραγωγούς να λαμβάνουν δίκαιες τιμές, που να επιτρέπουν να επιζούν, να ζουν. Και πρέπει να επιτρέψουμε σε μία κατάσταση που θα μας επιτρέψει να επανεξετάσουμε την εγκατάλειψη των μηχανισμών παραγωγής ούτως ώστε ο κλάδος αυτός να είναι δυναμικός, ζωντανός, πολλοί αγρότες να μπορούν να ζουν από αυτή τη δραστηριότητα και ούτως ώστε να επιζήσει και η ύπεθρος. Γιατί αυτά που μας λέγονται εδώ θα οδηγήσουν στην καταστροφή του κλάδου που σήμερα είναι σημαντικός και μπορεί να είναι και πολύ πιο σημαντικός. Ευχαριστώ πολύ και να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Ο κύριος Χάψελ. Με εκπλήσει το ότι δεν λέμε ότι έχουμε πολλά προβλήματα στην αγορά. Αυτά πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το πακέτο γάλακτος, πρέπει να πω ειλικρινά, νομίζω ήδη από την αρχή ήταν καταδικασμένο να αποτύχει. Διότι η ανισότητα μεταξύ των παραγωγών ε, και των υπόλοιπων ε, στοιχείων φάσεων της ε, διαδικασίας εφοδιασμού αυξήθηκε. Κύριε εκπρόσωπε του Κόμπα Κοζέκα, χρόνια μας λέγατε ότι η ελπίδα μας είναι η παγκόσμια αγορά για τους Ευρωπαίους παραγωγούς γαλακτοκομικών. Και παίξατε ρόλο στη φιλελευθερωποίηση. Παίξατε ρόλο στο ότι ήδη εδώ και χρόνια στην πράξη έχει καταργηθεί το σύστημα ποσοστώσεων. Και τώρα να έρχεστε να μα λέτε ότι α, δεν λειτουργεί αυτό. Και ότι πρέπει πάλι να πληρώσει ο φορολογούμενος. Νομίζω ότι είναι λιγάκι αφθάδε. Τώρα να πούμε ότι χρειαζόμαστε πάλι επιστροφέ για τι εξαγωγέ. Μα αυτή ήταν η πολιτική σα όλα αυτά τα χρόνια. Απέτυχε η πολιτική σα τι φιλεπτροπής. Και ήταν η πολιτική και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάλιστα την εφάρμοσε πολύ επιθετικά. Οπότε, ειλικρινά, τίθεται το ερώτημα. Υπάρχουν ιδέες για να επανέλθει η αγορά στην, ε, σε μια ισορροπία. Αλλά μέσω επιδοτήσεων από τους φορολογούμενους θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η πολιτική της δεκαετίας του 70. Έχει ξεπεραστεί. Δεν θα ξεπεράσουμε έτσι την κρίση στον τομέα αυτό. Δεν θέλουμε να επανέλθουμε στο παλιό σύστημα ποσοστώσεων, αλλά θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα όρια τη παραγωγή στην Ευρώπη. Πώ μπορούμε να επανέλθουμε σε ισορροπία στην αγορά, πώ μπορούμε να επικεντρωθούμε στην εσωτερική αγορά και όχι σε τύπους όπω ο Πούτιν και οι Κινέζοι. Αυτά είναι μέτρα μέλλοντο. Σα παρακαλώ και το λέω και στου ειδήμονε, Στραφείτε στην εσωτερική αγορά και να μην μα πείτε ότι η σωτηρία μα είναι στην Κίνα και στη Ρωσία. Αυτά έχουν αποτύχει ήδη. Και θα αποτύχουν και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσει. Η μία προ τον κύριο Ρέιμοντ. Μπορείτε να μα δώσετε ένα παράδειγμα του πώ νομίζετε ότι οι εξαγωγικέ πιστώσει και το ασφαλιστικό του σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει και δεν θέλω να τα καλύψω όλα όσα θα μπορούσα να πω στον κύριο Ντάνκαν Μον. Ε, λυπάμαι που τόσο αγενό σα διέκοψαν στο δεκαλεπτό σα. Προσπαθήσατε να πείτε την αλήθεια σα για αυτά που κάνατε εσεί στο δικό σα αγρόκτημα για να παραμείνετε στην αγορά και να διατηρήσετε την παραγωγή σα. Απλώ είπατε την αλήθεια. Αν κάποιοι έχουν αντιρρήσει εδώ, καλό θα ήταν να μην έρχονται καν σας έπληξε μια καταστροφική ασθένεια, μια επιζωτία πριν από 2-3 χρόνια, θα μπορούσατε ίσως να μας εξηγήσετε τα συμπτώματα ε, για όσους εδώ ενδιαφέρονται για τις γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες και να μάθουν από τις δικές σας ε, εμπειρίες ως, ε, σαν να ήσασταν ένα ειδικό χειρίδιο. Και εδώ όταν ξαναρχίσετε τη παραγωγική δραστηριότητα, τη ζωοτροφική, θα έχετε διαφορετικό τρόπο για, να, για τις αγελάδες σας, για να τις τρέφετε. Πρόεδρος. Και τώρα ερωτήσεις από τους συναδέλφους. εκεί Δία Γκαρσία. Ευχαριστώ πολύ ως υπεύθυνη του ΕΛΚ για την έκθεση αυτή του κ. Νίκολσον θέλω να ρωτήσω την κυρία Ουγιώα αναφέρθηκε στην κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις των παραγωγών για ποιο λόγο μόνο το 30% των παραγωγών συμμετέχουν σε αυτούς τους οργανισμούς που τους δίνουν ε, περισσότερη διαπραγματευτική ισχύ. Δεν γνωρίζουν την κατάσταση. Είναι θέμα αδράνεια, δεν είναι επαρκή ο επαγγελματισμό των οργανώσεων παραγωγών. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι ή άλλω πρέπει με σεβασμό να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Ξέρουμε ότι λύγει το σύστημα των ποσοστώσεων. Νομίζω ότι με μια σωστή συζήτηση θα ήθελα να ρωτήσω τους εκπροσώπους των παραγωγών. Βεβαίω, να μας πείτε, θέλουμε να σώσουμε τον τομέα αυτό ή θέλουμε απλώς να αξιοποιήσουμε τον τομέα αυτό για να κάνουμε κρατιστική πολιτική. Θα ήθελα παρακαλώ απαντήσεις και από τον κύριο Νίκο. Ευχαριστώ πολύ. Έχω συμμετάσχει σε δύο εργαστήρια του Ευρωκοινοβουλίου και αυτό είναι το τρίτο. Σε όλα ε, τα εργαστήρια μιλήσαμε για την κρίση ε, στον καθένα από τους τομέα και είδαμε, από τους τομείς. Και είδαμε ότι εδώ έχει πολύ σημαντικές συνέπειες όχι μόνο για τους γαλακτοπραγωγούς αλλά και για τον τομέα της ε, σόγιας ας πούμε. Πάντοτε πλήττονται οι παραγωγοί. Εδώ είδαμε τον κύριο ε, Βογκανό να μας μιλάει για θέματα πολύ αρεσικητικά για να ξεπεράσουμε αυτό το ροζ χρώμα που μέχρι τώρα έχει επικρατήσει με την ανανέωση του γαλακτοκομικού ε, τομέα είδαμε ότι η μετατροπή και η μεταρρύθμιση στον τομέα αυτό δεν επέτυχε τους στόχους τους και τα σχόλια, οι παρατηρήσεις που ακούσαμε σήμερα εδώ δείχνουν ότι για την παραγωγή και την επεξεργασία τα μέτρα που έχουν ληφθεί, που έχουν ληφθεί δεν λειτουργούν δεν ήταν αποτελεσματικά τα μέτρα για τη χώρα προέλευσής μου, την Πορτογαλία και πιο συγκεκριμένα για τις Αζόρες. Εκεί όπου ο τομέας έχει πληγεί, πληγεί Εδώ λοιπόν υπάρχει επιτακτική ανάγκη, κάτι που σήμερα έγινε από κάποιους από τους ομιλητές, να λάβουμε υπόψη όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής. Δηλαδή να ευαισθητοποιήσουμε και τους καταναλωτές για τις επιλογές του και να προστατέψουμε τους παραγωγούς. Τους παραγωγούς που έχουν υποστεί τι μεγαλύτερε συνέπειε και αδίκω πλήττονται από την κρίση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Ριμπέιρο. Κυρία Ριμπέιρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ξέρουμε όλοι ότι από την επομένη 1η Απριλίου θα καταργηθούν οι γαλακτοκεντές ποσοστώσεις. Ξέρουμε όμως τι γίνεται με τη μείωση των, ε, εξαγωγών από, την Κίνα, τη μείωση των εξαγωγών προς τη Ρωσία και την πτώση των τιμών που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν λοιπόν δύο αντιφατικά στοιχεία εδώ. Ότι δίνουμε έμφαση στι εξαγωγέ και προσπαθεί το Κοινοβούλιο να στηρίξει αυτή την προσπάθεια με, την, ε, με τα διάφορα μέτρα και δυνατότητε που διαθέτουμε. Αλλά από την άλλη πρέπει να δώσουμε έμφαση και στην εσωτερική αγορά. Αυτό το βλέπουμε τώρα με το καθεστώ ε, τη διανομή λόγου χάρη, με το σύστημα διανομή γάλακτο στα σχολεία. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, να προσέξουμε τι θα γίνει με την εσωτερική αγορά ότι μπορεί να ε, να μην έχουμε λάβει υπόψη τις δημογραφικές αλλαγές, ε, την δημογραφική μείωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για σκοπούς προστασίας λοιπόν του παραγωγού και αυτό θέλουμε, των παραγωγών και αυτό θέλουμε να το συζητήσουμε στο Κοινοβούλιο πρέπει να βρεθούν μηχανισμοί ελέγχου της ζήτησης και για την ποσότητα και για την ποιότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων διότι οι τιμές μειώνονται αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα την, σωστό υπολογισμό της ποσότητας και της ποιότητας των, προϊόντων και για το τρίμηνο που μας μένει και για το επόμενο διάστημα. Τι μέτρα μας επιτρέπετε, τι μας προτείνετε για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά αυτή τη μετάβαση. Λοιπόν, είπατε ότι μέσω των ποσοστώσεων δεν μπορούμε να επιτύχουμε τίποτα διότι ήταν άλλη η κατάσταση όταν ε, εισήχθησαν και τώρα θα καταργηθούν. Άρα πρέπει να προετοιμαστούμε για την επίπτωση της νέας κατάστασης. Υποστηρίζω εκείνους που μίλησαν για μακροπρόθεσμα προγράμματα, δηλαδή σχέσεις ε, σταθερές μεταξύ παραγωγών και μεταποιητών. Και σε εμά όμως ε, είναι πολύ δυσχερής η κατάσταση των παραγών και αν δεν αντιδράσουμε οι μειονεκτικές περιοχές θα αντιμετωπίσουν όλο και πιο δύσκολες καταστάσεις. Και ξέρουμε φυσικά ότι οι πολυεθνικές ε, έχουν όλο και περισσότερη ε, επίδραση στην εξέλιξη της κατάστασης. mesdames, messieurs, la fin des quotas laitiers, c'est la victoire idéologique. Κυρίε και κύριοι, το τέλο των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων σημαίνει τέλο τη κερδοσκοπία. Όταν πρωτοπάρθηκε αυτή η απόφαση δεν είχε ακόμα σημειωθεί η μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση. Και τότε οι περισσότεροι αναλυτές έλεγαν ότι θα υπήρχε σταθερότητα των τιμών των πρώτων υλών. Σήμερα όμως όπου υπάρχουν τόσες πολλές πολιτικές πολιτικές και γεωπολιτικές πιέσεις πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των συμπολιτών μας ιδίως στη Γεωργία. Γιατί σήμερα να μην κάνουμε ό,τι κάνουν και οι άλλοι στρατηγικοί αναλυτές, δηλαδή για να σώσουμε μεγάλο τμήμα του ευρωπαϊκού μας παληθισμού. Ο κύριος Λουαζόν, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο τερματισμός των ποσοστώσεων σημαίνει ότι ο τομέας πάει καλά και ότι άρα η κρίση ήταν ελάχιστη. Αυτό όμως είχε υπολογιστεί πριν, σημειωθούν, πριν σημειωθεί η χειροτέρευση των διεθνών σχέσεων και το ρωσικό εμπάργκο. Πράγματι το τέλος των ποσοστώσεων ανησυχεί τους ασχολούμενους στον τομέα και εδώ και 10 περίπου χρόνια στη Γαλλία χάσαμε 40% των γαλακτοκομικών μας εξαγωγών, πράγμα που αποτελεί ρεκόρ. Ιδίω οι μικροί παραγωγοί αναγκάζονται να συνεργαστούν μεταξύ τους και να συνεταιριστούν δημιουργώντας τις λεγόμενα αγροκτήματα εργοστάσια με συγκέντρωση μέχρι και 2.000 ζώων από μερικούς παραγωγούς. Αυτό είναι πρωτοφανές. Σε γεωγραφικές περιφέρειες όπου υπάρχουν λίγα αγροκτήματα, η λύση θα ήταν να επιστρέψουμε στην εθνική κυριαρχία, τουλάχιστον για τις τροφές στη Γαλλία, με την εφαρμογή μιας γαλλικής αγροτικής πολιτικής. κυρίες και κύριοι. Αν ο καθένας μιλάει τόση ώρα, τότε μερικοί δεν θα λάβουν το λόγο. Ένα λεπτό είπα, κύριε Ρόμπης. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική από χώρα σε χώρα. Σε ορισμένες χώρες το πακέτο λειτουργεί καλά, σε άλλες όχι. Το Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα δεν είναι τόσο άσχημη φαίνεται η κατάσταση. Αυτό πρέπει να το πρότυπό μα. για να λύσουμε ορισμένα προβλήματα. Σε άλλες χώρες, στις βαλτικές χώρες για παράδειγμα, είναι πολύ διαφορετική κατάσταση. Αν δεν ληφθούν αποφάσεις για μηχανισμούς, ε, αν δεν είχαν ληφθεί αποφάσει για μηχανισμού επιστροφών, τότε δεν θα υπήρχε πλέον παραγωγή γαλακτοκομικών. Έγιναν διάφορε προσπάθειε από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και από άλλους. Όμως η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται. Γιατί? Γιατί υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Γιατί λοιπόν δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερες οι τιμές του γάλακτος όταν έχουν πέσει οι τιμές των καυσίμων, για παράδειγμα. Γιατί να μην είναι χαμηλότερο η τιμή του γάλακτος στο σούπερ μάρκετ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που έχουμε δει ως τώρα είναι να υπάρχουν τεράστια προβλήματα με την επεξεργασία ε, είτε λόγω της διακύμαση των τιμών είτε λόγω της διάρκεια των συμβάσεων. Αυτό που θέλω να ρωτήσω όμως είναι ε, δεν νομίζετε ότι οι οργανώσεις παραγωγών και η συνένωσή τους επιτρέπει να δημιουργήσουν τα δικά τους σχέδια για την μεταποίηση και την επεξεργασία προϊόντων. Δεν είναι καλύτερο αυτό για τη δημιουργία μιας αλυσίδας διανομής που να είναι καινούργια και να ανεξαρτοποιηθούν από τις, από τις σημερινές δεσμεύσεις Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω αυτό είναι και το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μποβέ. Κύριε Πρόεδρε. πριν από δύο χρόνια η πολιτική μας ομάδα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεώρησε ότι ήταν προβλέψιμα αυτά που γίνονται σήμερα, <laughs> διότι ο τρόπος εφαρμογής των συμβολέων και των τιμών δεν έχει καμία εγγύηση, ούτε καμία διαφάνεια. Δεύτερον, δεν έγινε τίποτα εκτός από τις ε, ετικέτες προέλευσης. Τίποτε για το συνδυασμό του όγκου της παραγωγής με τις τιμές και γι' αυτό καταλήξαμε σε κρίση τον Απρίλιο και το ξέρανε όλοι. Τρίτον, οι σημερινοί δείκτες είναι πάρα πολύ φλού και σε μεγάλη καθυστέρηση σε σύγκριση με τους διεθνείς δείκτες. Ας παραμείνω εδώ. Αλλά πρέπει πρώτον να ορίσουμε τι είναι κατάσταση κρίσης, δεύτερον ποια είναι η μέθοδος υπολογισμού των δικτών και με τι διαφάνεια και τρίτον πώς θα δημιουργήσουμε μια σωστή διαχείριση των τιμών σε σύγκριση με την παραγωγή. Αν δεν καταλήξουμε σε ένα κοινοβουλευτικό ψήφισμα που να το αναλάβει η Κομισιόν τότε πάλι οι γεωργοί στο τέλος θα πληρώσουν την ύφη. Ο κύριος Βιέγκας, ευχαριστώ. Από την πλευρά μας συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι το σύστημα ποσοστώσεων πρέπει να διατηρηθεί. Η απόφαση έχει ληφθεί βέβαια, μέσω πρόθεσμα να ε, εξελιχθεί, όμως ας ε, σήμες του ας θυμηθούμε τι έγινε με έναν μελοθάνατο που δέχτηκε την απόφαση χάριτος ε, στα 37 του λίγο πριν εκτελεστεί. Ε, τελικά σώθηκε. Άρα ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ακόμα δυνατότητες για λίγη δικαιοσύνη στην κατανομή των δικαιωμάτων και των ωφέλων, των ωφελών από την μεταρρύθμιση του γαλακτοκομικού τομέα το εσωτερικό των κρατών μελών και στι διάφορε περιφέρειε. Όσο αυξηθούν οι τιμέ, θα επιτρέψει αυτού του παραγωγού να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Η, στην Πορτογαλία αυτό που επιθυμούμε είναι να διατηρηθεί η παραγωγή γάλακτο για όσου έχουν κρατηθεί στην αγορά. Αυτό που θέλουμε λοιπόν το Κοινοβούλιο είναι μια γραπτή δήλωση, ε, ώστε ε, όσοι έχουν αντίρρηση με το σύστημα ποσοστώσεων να μπορέσουν να συνυπογράψουν. Θα συνεχίσουμε να αντιστοιχόμαστε, διότι αυτή η μεταρρύθμιση, αυτό το πακέτο, είναι μια οπισθοχώρηση. Ουσιαστικά τι λέμε, ότι είναι μέτρα ασφαλεία αυτό που υπήρχε πριν από τις ποσοστώσεις και που οδήγησε στην επιβολή των ποσοστώσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ταραμπέλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τέσσερι γρήγορε παρατηρήσει. Πρώτον, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι τώρα βρισκόμαστε στα πρόθυρα μια μεγάλη κρίση ή θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγο να είμαστε σε επιφυλακή, διότι στην περιοχή μου ήδη από τον Ιανουάριο πωλείται το γάλα 25 λεπτά. Εδώ για τι εξαγωγέ και τα σχόλια που έγιναν, αν θέλουμε να ανταγωνιστούμε τι λιγότερο προηγμένε χώρε, είναι απαράδεκτο αυτό. Θα πρέπει να είναι συνεκτικέ οι πολιτικέ ανάπτυξη που έχουμε με τι αγροτικέ πολιτικέ. Τρίτον, η μόνη οργάνωση παραγωγών που είναι αποτελεσματική όπως τη γνωρίζω είναι το, η, ο Καναδε, Καναδέζικος φορέας γάλακτος. Είναι όμως δημόσιος φορέας. Μπορούμε να φανταστούμε σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων ότι θα γίνει ο δημόσιος κλάδος το χροφύλακα των αγορών ή θα αφήσουμε τις αγορές να κάνουν ό,τι θέλουν τις εταιρείε να μεγαλώνουν και να συγκεντρώνονται όλο και περισσότερο. Και τέσσερα, πολύ γενικότερα. Όλοι οι μεγάλοι γεωργικοί παράγοντες επιδοτούν πλέον, τις, ε, συνδέουν ξανά τις ε, βοηθειές τους και στηρίζουν τους παραγωγούς τους. Εμείς από τότε που αποσυνδέσαμε την παραγωγή και δεν επιδοτούμε τους παραγωγούς έχουμε πολύ ε, μεγαλύτερη και οξία κρίση. Αυτά ήθελα να διαπιστώσω και να τα λάβουμε υπόψη. Ευχαριστούμε η κυρία Πετήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω τη λύπη μου γιατί δεν μπορέσαμε σήμερα να ακούσουμε γαλακτοπαραγωγούς από καμία καινούργια χώρα μέλος. Θα ήταν σημαντικό να τους ακούσουμε και αυτούς για να καταλάβουμε όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για την εφαρμογή της δέσμης γάλα, του γάλακτος, του γαλακτοπαραγωγικού τομέα. δεν έχει νόημα να προσωμιάζουμε την κατάσταση των μικρών με τους μεγάλους παραγωγούς. Δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια οικονομικά προβλήματα. Οι Κροάτες γαλακτοπαραγωγοί δεν είναι μέτοχοι ή συνειδιοκτήτες βιομηχανιών μεταποίησης όπως γίνεται στα περισσότερα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Γι' αυτό θα ήθελα να σας αναφέρω ποια είναι η κατάσταση στην Κροατία. Στη χώρα μας δεν παράγουμε αρκετά, αρκετό γάλα και είναι και οι τιμές απαράδεκτες πολύ υψηλέ, διότι υπάρχουν υπόλοιπες χώρες μέλη των οποίων η παραγωγή στηρίζεται από εθνικά μέτρα. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Ρεμόν μήπως δεν θα μπορούσαμε σε ενωσιακή κλίμακα όπως έλεγε και η Κόπα Κοζέκα να γίνουν συμφωνίες, να συναυθούν συμφωνίες προστασίας της μικρής παραγωγής γάλακτος όπως της Κροατίας για να προστατευτεί από γαλακτοκομικά προϊόντα που τα στηρίζουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και που άρα αποτελούν αθέμητο λίγο ανταγωνισμό. Άντριου. Μερικά ερωτήματα για τους εμπειρογνώμονες. Μετά από αυτά που είπε ο Ταραμπέλα, νομίζω ότι μια ανακατανομή προς τις ε, πιο ευαίσθητες και προβληματικές ζώνες θα μπορούσε να συζητηθεί και μια κάποια επιστροφή σε επιχορηγήσεις. Επίσης, οι μηχανισμοί αντιμετώπισης κρίσεων για τη λεγόμενα κυκλικά συμβόλαια. Η επιστροφή σε αποθήκευση με υψηλότερη τιμή και με έλεγχο παράλληλα του όγκου της παραγωγής, τι θα σας έλεγε. Μήπως σε αυτή τη φάση θα έπρεπε να πάρουμε μαθήματα, να τα αποτιμήσουμε και να συγκρίνουμε με την κατάσταση στην Αμερική για να βρούμε μια λύση. Σας ευχαριστώ. Μετά θα μιλήσει ο κύριος Διευθυντής για πέντε λεπτά και μετά θα ξαναρχίσει η απαντήσεις Ορίστε. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ευκαιρία να σας απευθυνθώ πολύ γρήγορα και να αντιδράσω στις παρουσιάσεις που έγιναν για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα και επικαιριά ακρόαση και να καλωσορίσω το γεγονό ακριβώ ότι λαμβάνει χώρα η ακρόαση αυτή. Να πω αυτή εξ αρχή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει επακριβώ ποια είναι η κατάσταση στο γαλακτοπαραγωγικό τομέα και γνωρίζει ότι τα πράγματα αλλάζουν είναι λοιπόν πολύ καλή και κατάλληλη στιγμή για να δούμε τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων. Ε, τα πράγματα αλλάζουν. Γιατί, γιατί μετά από 30 χρόνια ποσοστώσεων ε, καταργούνται. Η απόφαση για την ε, εξαλειφθή του συλλήφθη το, 2003 και με την μετέπειτα μεταρρύθμιση επιβεβαιώθηκε. Αυτό που δεν είδαμε ακόμα και μου πρώτος αυτό το παραδεχτή είναι ότι Τότε δεν ξέραμε στις αρχές του 2014 ότι οι τιμές θα πέσουν και μάλιστα τόσο γοργά. Αυτό μας ευνηδίασε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ο αλληλεσχετισμό μεταξύ των δύο δεν, των δύο δεν αποδεικνύεται. Είχαμε κρίση στο γαλακτοπαραγωγικό τομέα και στα έτη των ποσοστών τιμών το 2009 και το ανέφεραν πολλοί από του ομιλητέ εδώ. Ε, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν προβλήματα. Δεν ήταν επανάκια για την διακύμαση των τιμών ή το σύστημα των ποσοστώσεων. Νομίζω όμω ο συνδυασμό, όπω είπε και ο κ. Νίκολσον, τη εξάλληψη των ποσοστώσεων από τη μια και τη πτώση των τιμών δυστυχώ ανησυχεί. Αυτό δεν θα το αρνηθώ αλλά οι τιμές έχουν μειωθεί βάσει των αριθμών μας μεταξύ 34 ε, λεπτών το κιλό το 2000, με συγχωρείτε 40 λεπτά ε, το 2013 σε 42 τον Δεκέμβριο του 2014. Και αυτό γιατί υπάρχει ε, αλλαγή, υπάρχουν μεταβολές στην παγκόσμια αγορά, αλλά και η παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί κατά 5%. Όλα αυτά έχουν ενταθεί από το ρωσικό εμπάργκο. Κάτι που δεν βοηθά καθόλου την κατάσταση. Σε αυτό το τοπίο σημαντικό είναι να επισημάνουμε ότι οι μακροπρόθεσμε προοπτικέ για το γαλακτοπαραγωγικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένουν πολύ καλέ. Και αυτό δεν είναι άποψη μόνο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των ειδικών τη, αλλά και του ΦΑΟ και τη Παγκόσμια Τράπεζα και πολλών άλλων. Τώρα, για, το, για τη δέσμη μέτρων για το γάλα. Ε, νομίζω ήταν πολύ καλέ οι προκατακτικέ παρατηρήσει του κ. Νίκολσον. Τι θα κάνουμε, αυτό είναι το σημαντικό να ρωτήσουμε. Οι τιμέ εντάξει πέφτουν, αλλά τι κάνουμε. Το πακέτο που προτάθηκε, ο σκοπό ήταν να προτείνει λύσει, να προτείνει λύσει στη μεταβαλλόμενη κατάσταση και στη μεγαλύτερη έκθεση των παραγωγών στην διακύμαση των τιμών στην αγορά. Ε, έτσι λοιπόν, ε, λιγότερο οι κανονισμοί, λιγότερε διακυμάνσει και περισσότερη ελευθερία για του ανθρώπου να λάβουν τι δικέ του αποφάσει. Έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Νομίζω είναι σαφέ από την έκθεση ότι δεν είμαστε ιδιαίτερω ικανοποιημένοι έχουν γίνει με το πακέτο για το γάλα. τα αριθμητικά στοιχεία μπροστά σα. Να πω στην κυρία Χέραν Σάντσεφ και βεβαίω θέλω να ακούσω και τι απόψει των ε, όσων εργάζονται επί τόπου και των ε, εμπειρογνωμόνων ειδικών ε, γιατί δεν ήταν σωστή η υλοποίηση, γιατί ήταν αρκετά ισχυρή. Γιατί οι τιμέ το γαλακτοπραγικό τομέα αυξάνονταν μέχρι πρόσφατα. Μήπω πρέπει να αναδιοργανωθούμε καλύτερα. Μήπω πρέπει κανεί να λειτουργήσει με τη λογική ισχύ εν τη ενώση. Ε, και αυτό μάλλον χρειάζεται τώρα περισσότερο από ποτέ. Επίση, να επαναλάβω κάτι που έχει πει και ο Επιτροπό μου ε, σε επανειλημμένε ευκαιρίε και χθε στο Συμβούλιο των Υπουργών, ότι Βεβαίω η απάντηση κλειδί εδώ είναι η παραγωγή να γίνουν ισχυρότερη στην όλη αλυσίδα και όχι μόνο μέσω του πακέτου για το γάλα, αλλά και τη πρωτοβουλία για την διατροφική αλυσίδα και άλλων πρωτοβουλίων που έχουν αναλυθεί. Και θα επιδιώξουμε. Άλλα πράγματα, πολύ σύντομα, που θέλω οπωσδήποτε να αναφέρω, είναι πόσο χρήσιμο είναι το παρατηρητήριο για την αγορά του γάλακτος και για μας, γιατί συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τους εμπόρους και τους χρήστες σε αυτό το νέο οργανισμό για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά δεδομένα στη διάθεσή μας για τις εξελίξεις στην αγορά. Πραγματικά γίνεται έρευνα για να έχουμε τι καλύτερε δυνατέ πληροφορίε, ώστε να είναι ο μηχανικό κλάδο ενήμερο για το τι αποφάσει να λάβει. Και τέλο, γιατί και αυτό αναφέρθηκε, οι άμεσε πληρωμέ ακόμη υπάρχουν και για τον γαλακτοπαραγωγικό τομέα και τη συνδεδεμένη εθελοντική βοήθεια. Προβλέπετε αυτό. Προβλέπετε και σύντομα θα ξαναγυρίσουμε σε εσά για να σα δώσουμε μια συνολική επισκόπηση για το πώ ε, υλοποιούν το σύστημα αυτό τα κράτη-μέλη. 18 από τους 28 ήδη έχουν αυξημένη εθελοντική συνδεδεμένη βοήθεια για το γαλλικό τομέα. Και υπάρχει και το εργαλείο για την ε, ε, στήριξη των παραγωγών, γιατί αναγνωρίζουμε ότι περνάνε μια δύσκολη περίοδο. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Θυμηθείτε, υπήρχε το σύστημα των ποσοστώσεων και υπήρχαν και τότε κρίσεις και γνωρίζαμε ότι οι ποσοστώσεις μια μέρα θα καταργηθούν και πρέπει να δούμε πώς θα ενδυναμωθεί η όλη τροφιμική αλυσίδα με τι εργαλεία, με τι μέσα έχουμε τώρα δύο λεπτά για τους εμπειρογνώμονες όχι παραπάνω Ευχαριστώ πρόεδρε Μία σύντομη απάντηση προς τον κύριο εκεί πίσω που αφορούσε επιστροφές. Εγώ είπα ότι αυτά χρειάζονται μόνο σε περιπτώσεις κατεπίγουσας ανάγκης, όπως γίνεται και στην Αμερική, όπου δίνονται διασφαλίσεις εγγυήσεις για εταιρείες που θέλουν να αγοράσουν ένα προϊόν αλλά φοβούνται να το πράξουν. Είναι μια πολιτική στήριξη λοιπόν για να μπορέσουν οι δοσοληψίες να συνεχίσουν με νέες αγορές, νέες χώρες. Γι' αυτό μιλάμε, για να κινηθεί η αγορά. Δεν είμαστε υπέρ των συστηματικών τέτοιων επιστροφών στην κόπα Κοζέκα για αυτά που είπατε εσείς κύριε Πρόεδρε για τις ποσοστώσεις. 30 χρόνια κράτησαν. Χρειαζόμαστε διαφοροποιημένη βιομηχανία και οικονομία. Θα υπάρξουν ευκαιρίες, υπήρχαν και άλλες κρίσεις. Και εγώ είχα ένα ακρόκτημα γαλακτοπαραγωγικό και αντιμετώπισα κρίσεις και καταστροφές δύο-τρεις φορές. Δεν είναι λοιπόν η απάντηση σε όλα τα ερωτήματα ή ποσοστώσεις Πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε ένα διαχειριζόμενο σύστημα ή ένα αναπτυσσόμενο σύστημα. Αλλά και τα δύο χρειάζονται μια βιομηχανία που να λειτουργεί και να αυξάνεται. 5% αυξήσεις παραγωγικότητας και στο γαλακτοκομικό τομέα σημειώθηκαν στην Ευρώπη, 2% μειώθηκαν λόγω της ρωσικής κρίσης, υπάρχουν λοιπόν ακόμη προβλήματα. Βίλα Είναι σαφές ότι μια πολιτική που δίνει τιμές για τους παραγωγούς χαμηλότερες από το κόστος παραγωγής οδηγεί στην άβυσο. Τι θέλουμε να κάνουμε. Αυτό που ανταποκρίνει και σε αυτό που απαιτούν οι πολίτες είναι να διατηρηθούν όλα τα αγροκτήματα και να υπάρχει γαλακτοπαραγωγή σε όλες τις περιφέρειες με βιώσιμο τρόπο. Δεν είναι δυνατό να δεχθούμε τεράστιες εισαγωγές και να γίνονται επιστροφές μέσω χρήματος των φορολογουμένων. Στην ουσία δηλαδή ευνοούμε τρίτες χώρες. Πρέπει λοιπόν να αναθεωρηθεί αυτή η πολιτική καταστροφή της παραγωγής. Έχουμε σαφές πρόβλημα με τις ποσότητες. Υπάρχει πρόβλημα και παίζει ρόλο στις τιμές. Ως αποτέλεσμα χάνονται χιλιάδες εκμεταλλεύσεις. Πρέπει να μείνουν ζωντανές αυτές οι περιοχές με βιώσιμη λειτουργία των εκμεταλλεύσεων. Θέλουμε επίσης ένα εντατικό σύστημα. Συγγνώμη. Αν προωθούμε εντατικό σύστημα μπορεί να έχουμε μεγάλες ε, συγκεντρώσεις νητρικών. Σε μια διαδικασία διαβούλευσης είπαμε ότι κάθε χρόνο πεθαίνουν 25.000 ε, άτομα από τα προβλήματα αντίστασης στα αντιβιωτικά. Επίσης υπάρχει ένα πρόβλημα δυσανεξίας στη λακτόζη που έχουν πολλοί πολίτες, αλλεργίες. Πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσουμε για ποιότητα, γιατί είναι τρόφιμα αυτά, αλλά και απασχόληση διατήρηση της υπαίθρου. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Δεν είναι δυνατόν απλώς να παράγουμε πρώτη ύλη χαμηλού κόστους για, τους, για τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Ο κύριος Μάουγκεν. την ερώτησή σας για το τι μου συνέβη εμένα ως κτηνοτρόφου. Είχα το πρόβλημα της λιμόδους πλευροπνευμονίας στο αγρότημά μου που ε, μόλυνε τα πάντα. Αν αυτό ε, συμβαίνει, συμβεί και σε άλλες χώρες θα είναι πολύ δύσκολο να σκεφτεί κανείς τι θα κάνει με το πλεόνασμα του άλεκτο, διότι θα ξέρει πια από πού θα πάρει γάλα. Ε, ε, υπάρχουν τέτοιες επιζωοτίες ασθένειες που θα παρει γαλα ε υπαρχουν τετοιε επιζωοτιες ασθενειες που πρεπει να τις ελέγξουμε. Δεν θα ήθελα κανείς να περάσει αυτό που πέρασε εγώ την τελευταία διετία. Ήταν ε, φρικτό. Ε, το μισό κοπάδι να σου πεθαίνει στα χέρια. Δεν είναι κάτι ευχάριστο. Είμαι πολύ τυχερός που έχω μία σύμβαση με κάποιον αγοραστή αλλά θα ένα καλύτερη τιμή αν μπορούσα να παράγω αυτά που ήθελε. Μία κυρία είπε ότι δεν έπρεπε να αναφερθούν οι μάρκες, αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Ε, ε, είναι πώς θα προωθηθούν καλύτερα τα γαλακτοκομικά προϊόντα στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πάει το γάλα και στα σχολεία, στα παιδιά. Και πρέπει να είμαστε σαφέστεροι για την ασφάλεια των καταναλωτών, πώς θα τους πείσουμε και πώς μέσω των αγοραστών μας θα καταλήξουμε στον τελικό χρήστη. Όχι να προσπαθήσουμε με αριθμητικά σκευάσματα να ξεφύγουμε από το πρόβλημα. Πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να βρούμε λύσεις. Ευχαριστούμε. Και τώρα η κυρία Ουλούα. Θα παρακαλέσω το επόμενο πάνελ πρέπει να ετοιμαστεί. Έχουμε τον ε, καθηγητή Λούντβιχ Τόισεν Δύο λεπτά για την ώρα για τον κύριο Ολούα. Ως περιφερειακή υπεύθυνη για την γαλακτοκομική πολιτική στην Γαλλικία θέλω να τονίσω αυτό που ήδη υπόθηκε ότι διαπιστώσαμε μείωση των ε, τιμών δημόσιας παρέμβασης και αλλού στην Ισπανία και στη Γαλλικία. Οπότε υπάρχουν πολύ ισχυρέ διακυμάνσει στην τιμή του γάλακτος που εξαρτάται αυτό από εξωτερικούς παράγοντες της παγκόσμιας αγοράς. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα θέλουμε πρώτα απ' όλα αύξηση τη τιμή παρέμβαση, αλλά και άλλα μέτρα για να ενισχυθεί το πακέτο γάλακτος, να έχουμε τις σωστές σχέσεις μεταξύ των διαφόρων συμμετεχόντων στην παραγωγή και να είναι ισότιμες οι σχέσεις τους, όχι ανισότιμες όπως σήμερα. Όπως υπόθηκε, στην Ισπανία τα συμβόλαια είναι υποχρεωτικά και υποχρεωτική διάρκεια στον Για το νοπό γάλα όπως το ορίζει ο κανονισμός της Ένωσης. Θέλουμε αυτό να επεκταθεί όχι μόνο στο νοπό γάλα αλλά και το μεταποιημένο, αυτό που καταλήγει στα σούπερ μάρκετ. Έτσι θα ενισχυθεί η θέση των άλλων συμμετεχόντων να μην είναι η παραγωγή πιο αδύναμη. Στις σχέσεις τους με τις βιομηχανίες και τους ε, διανομής. Γιατί δεν υπάρχουν συμβόλαια σε όλες τις φάσεις διαδικασίας. Αυτό σημαίνει συχνά ότι ο παραγωγός παρετείται του δικαιώματός του να έχει μακροχρόνια συμβόλαια. Γι' αυτό θέλουμε τα συμβόλαια να περάσουν και στη σχέση με τους διανομής και όχι μόνο για τον οπό για τις άμεσες ενισχύσεις θεωρούμε ότι επειδή το καθεστώς των ποσοστώσεων βοήθησε την αναδιάρθρωση πολλών εκμεταλλεύσεων χρειάζεται ακόμη βοήθεια η περιοχή μέσω αμέσων ενισχύσεων γιατί είναι η μειονεκτική περιοχή η Γαλλικία για να μπορέσει να συνεχίσει να παράγει και να είναι επικερδής η παραγωγή γάλακτος. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους μας τους εμπειρογνώμονες ε, αυτού του πρώτου πάνελ. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, ομιλίες σας. Με συγχωρείτε που ήμουν τόσο αυτερός με τον χρόνο, αλλά αυτός είναι ο ρόλος μου. Και τώρα θα έρθουν άλλοι εμπειρογνώμονε εδώ γύρω από το τραπέζι του Προεδρείου και όπως αλλάζετε θέσεις να κάνω μερικές ανακοινώσεις. Η έκθεση του κυρίου Ντόφμαν αλλά και η δική μου για τις μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις βλέπουμε ότι οι μικρομεσαίες εκμεταλλεύσεις χρειάζονται κάποια βοήθεια. Επίσης ε, και οι εκμεταλλεύσεις που είναι σε μειονεκτικές περιοχές, ορεινές, όλοι αυτοί χρειάζονται βοήθεια, οικονομική βοήθεια. Η ενιαία αγορά ίσως δεν κάνει αρκετά για να προωθήσει την κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών. Για πολλές χώρες δεν κάνουμε όλα όσα θα μπορούσαμε για να προωθήσουμε την κατανάλωση γάλακτο. Αυτά ήθελα να πω για να περάσει η ώρα μέχρι να ανέβουν οι άλλοι στο Προεδρείο. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο πάνελ, προοπτικέ για το αγροτικό τομέα. Πρώτος, ο καθηγητή Λούντβιχ Τόισεν από το Πανεπιστήμιο του Γκέρτιγεν στη Γερμανία. Θα έχει 10 λεπτά. Ε, ξέρω ότι ποτέ για πανεπιστημιακό δεν είναι αρκετά, αλλά αυτοί είναι οι κανόνες.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 Herr Vorsitzender. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, μου ζητήσατε να εκφραστώ για ορισμένα θέματα. Για το ποια είναι τα σενάρια μετά τη λήξη ε, των ποσοστώσεων και ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες από τις διεθνείς εξαγωγές και το μέλλον της παραγωγής γάλακτος σε διάφορες ε, μειονεκτικές περιοχές και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις για τα σενάρια μετά τις ποσοστώσεις πολλά υπόθηκαν. Νομίζω ότι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για τις αγορές ε, γάλακτος είναι καλές παρά τις ε, εξελίξεις τιμών. Διότι μεγάλες τάσεις όπως η αύξηση του πληθυσμού και οι αλλαγές των συνηθιών διατροφής ισχύουν και θα βοηθήσουν να υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς γάλακτος. Οπότε οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν όπως και στο πρόσφατο παρελθόν να μπορούν να λάβουν χρηματοδοτήσεις. Γιατί η κατάσταση είναι δυσχερή σε αυτή τη συγκυρία. Υπόθηκαν πολλά, υπάρχουν πολλοί λόγοι. Γενικά υπάρχει καλή, ε, καλός εφοδιασμός. Έχει μειωθεί η οικονομική ανάπτυξη της Ανατολικής Ασίας και δύσκολη, και δύσκολη κατάσταση στην Ευρώπη, η κρίση της Ρωσίας και η επέκταση της παραγωγής στην Ευρώπη. Εδώ στην Ευρώπη διαπιστώνουμε ότι οι χώρες που στο, που στο παρελθόν δεν εκπλήρωναν τις ποσοστώσεις ε, τώρα τις εκπληρώνουν επειδή έχει αυξηθεί η τιμή και παράγουν πολύ περισσότερο. Και άλλες χώρες όμως αύξησαν ε, την παραγωγή τους ε, πέρυσι, οπότε έχουμε πολλή προσφορά. Γενικά για τις γεωρικές αγορές, αγορές γεωρικών προϊόντων, Ακόμη και σχετικά μικρές αλλαγές στην ε, ποσότητα παραγωγής ε, ε, προκαλούν μεγάλες διαφορές τιμών γιατί είναι ανελαστική η ζήτηση. Οι τιμές λοιπόν είναι ιδιαίτερα μεταβλητές. Για το γάλα προστίθεται επίσης ότι από τη συνολική παραγωγή μόνο ένα μικρό τμήμα, μόνο 7% εξάγεται παγκοσμίως. Δηλαδή οι διεθνεί αγορές είναι σχετικά μικρές και μικρές αγορές προκαλούν μεγαλύτερε ε, μεταβολές τιμών. Επίσης ε, αυτή η μεταβλητότητα των ε, τιμών θα παραμείνει υψηλή. Το είπανε πολλοί ότι δεν έχει μεγάλη σχέση με την κατάργηση των ποσοστώσεων, αλλά με πολύ γενικότερα φαινόμενα που χαρακτηρίζουν την αγορά γάλακτο. Συνολικά, οι εξαγωγέ προ μη ενωσιακέ χώρες είναι ευκαιρία αλλά και κίνδυνος. Υπάρχουν ε, δυνατότητες γιατί αυξάνεται η ζήτηση για ασφαλή και υψηλής ποιότητας γαλακτοκομικά και σε μεγάλο βαθμό και στο μέλλον αυτά τα προϊόντα θα προέρχονται από την Ένωση. Επιπλέον, οι εξαγωγές προς αυτές τις χώρες, τις τρίτες, είναι ο μόνος τρόπος να μην εγκαταλείψουν ε, τη γαλακτοκομική παραγωγή πολλοί από του παραγωγούς μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν γιατί παράγουμε περισσότερα από όσα καταναλώνουμε εξαγωγές. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε και κινδύνου. Πέρα από τη μεγάλη μεταβλητότητα των τιμών υπάρχουν και προβλήματα ισοτιμιών, ε, μη δασμολογική ε, φραγμή στου εξαγωγέ κτλ. Ιδιαίτερα δύσκολε είναι οι, αυτές οι μεταβαλλόμενες περιοχές για τις ε, μειονεκτικές περιοχές γαλακτοπαραγωγής. Θεωρώ ότι η γενική γαλακτοκομική πολιτική δεν είναι ο σωστός τρόπος για να βοηθήσουμε τις μειονεκτικές περιοχές να σταθεροποιήσουν την τιμή τους. Διότι σε πολλές περιπτώσεις ε, η διαφορά κόστους παραγωγής σε σχέση με τις πιο ευνοημένες περιοχές είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να διατηρηθεί η παραγωγή αυτή. Για τις μειονεκτικές περιοχές θα πρέπει να εξετάσουμε μήπως υπάρχουν καταλληλότερε ε, διαδικασίες παραγωγής που να είναι κατάλληλες για τέτοιες περιοχές. Για παράδειγμα η εκτατική παραγωγή βοήου ή η παραγωγή ε, μητέρων, ε, δηλαδή αγελάδων για αναπαραγωγικούς σκοπούς. Επίσης ο δεύτερος πυλώνας θα μπορούσε να αξιοποιηθεί περισσότερο, να επεκταθεί περισσότερο. Οι τιμές του γάλακτος θα συνεχίσουν να είναι μεταβλητές, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι επαρκές επιχείρημα για να έχουμε προστατευτισμό στην αγορά. Θα πρέπει οι εκμεταλλεύσεις να διαχειρίζονται καλύτερα τις ε, κρίσεις και τους κινδύνους. Είναι επίσης επιχείρημα αυτή η μεταβλητότητα για να αναπτύξουμε τις αγορές επιπροθεσμία και άλλους μηχανισμούς για να περιορίσουμε τους κινδύνους. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι η τιμή παρέμβασης είναι ε, ουσιοδός χαμηλή, όπως είπαν πολλοί, να έχουμε υπόψη μας. Ότι αν ήταν ε, ουσιοδός υψηλότερη η τιμή παρέμβασης, θα είχαμε σοβαρές τρευλώσεις αγοράς. Πολύ ψηλό κόστος και θα ε, αυξάνονταν οι ποσότητες που θα ήταν αποθηκευμένες. Θέλουμε πραγματικά να επανέλθουμε στις ε, λίμνες γάλακτος και βουνά βουτύρου των 80, τη δεκαετία του 80. Δεν μπορούμε επιπλέον να λύσουμε το πρόβλημα μέσω ε, συγκεντρωτικής προσπάθειας καθορισμού των ποσοτήτων που παράγονται. Δηλαδή από την πίσω πόρτα να επανέλθουμε σε ποσοστώσεις. Δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες για το πώς εφαρμόζεται αυτή η συγκεντρωτική προσπάθεια καθορισμού της παραγωγής, αλλά η εμπειρία από άλλες χώρες δείχνουν ότι αυτά τα συστήματα είναι τρομερά ε, γραφειοκρατικά, είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν, γιατί πολύ συχνά δεν έχουμε την επαρκή πληροφόρηση γι' αυτό και δεν μπορούμε να την έχουμε εγκαίρως. Αυτές λοιπόν οι προσπάθειες είναι πολύ ακριβές γιατί οι ποσότητες που βγαίνουν από την αγορά συνήθως είναι πολύ μεγαλύτερε από ό,τι συνήθως ε, θεωρείται και τα συστήματα αυτά πολλές φορές δεν έχουν καμία επίπτωση. Γιατί να αναφέρω το παράδειγμα του Καναδά. Αναφέρθηκε ήδη σήμερα. Εδώ και δεκαετίες γίνεται η προσπάθεια στον Καναδά να ε, ελέγχεται η προσφορά γαλακτοκομικών. Αν δούμε τώρα πώς έχουν μειωθεί η παραγωγή όμως, θα διαπιστώσουμε ότι οι διαστροτικές αλλαγές στην παραγωγή αυτή ήταν τόσο ταχείες όπως και στις ΗΠΑ που έχει ένα πολύ πιο απελευθερωμένο σύστημα. Επιπλέον, να λάβουμε υπόψη ότι η γαλακτοπαραγωγή του Καναδά είναι στο επίπεδο της δεκαετίας του 60 ενώ οι άλλες μεγάλες περιφέρειες και χώρες που παράγουν γάλα έχουν αυξήσει κατά πολύ την παραγωγή τους. Κατά συνέπεια, το τμήμα του Καναδά στην παγκόσμια αγορά αγροτικομικού από το 1996 μέχρι το 2009 πήγε από 3% στο 1%. Ενώ για παράδειγμα το τμήμα των ε, Αμερικανών στην αντίστοιχα περίοδο πήγε από 6% στο 17%. Επιπλέον, στον Καναδά έχουμε πολύ περισσότερες εισαγωγές γαλακτοκομικών λόγω αυτής της πολιτικής. Δηλαδή το 1996 ήταν μόνο 8% ενώ το 2009 έχει ανέβει στο 24%. Τέλος, αυτή η πολιτική του Καναδά οδήγησε σε διάφορα ανεπιθύμητα φαινόμενα. Για παράδειγμα, λαθρεμπόριο τυριού από τις ΗΠΑ στον 21ο αιώνα και πολλές προσπάθειες ε, να παρακαμφθεί η νομοθεσία. Για παράδειγμα, στέλνουν κίτια πίτσα από τις ΗΠΑ του Καναδά με τυρί και κάτι ακόμη. Και έχει προκαλέσει και πολλές διαφορές και συγκρούσεις ε, εμπορικής πολιτικής. Πόρισμα λοιπόν. Βεβαίως ε, θέλουμε ένα δίκτυο ασφαλείας εάν υπάρχουν σοβαρές κρίσεις, αλλά συνολικά δεν θέλουμε κεντρικό καθορισμό του επίπεδου της παραγωγής. Δεν λειτουργεί κάτι τέτοιο. Τέλος, δύο λόγια για το TTIP, γιατί και αυτό ήταν ερώτημα που μας ετέθη. Η πείρα που έχουμε με τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου μέχρι τώρα δείχνει ότι οι επιπτώσεις της αγορές πρέπει να εξεταστούν σε λεπτομέρεια, γιατί φυσικά εξαρτώνται από το επίπεδο προστασίας των επιμέρους προϊόντων, για να δούμε ποια χώρα θα ωφεληθεί και ποια θα ζημιωθεί. Γι' αυτό η εξέταση πρέπει να γίνει αναπροϊόν, πολύ συγκεκριμένα. Αυτό ισχύει και για τα διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα συνολικά, χωρί τώρα να μπούμε σε λεπτομέρειε. Θεωρώ ότι για τα γαλακτοκομικά οι ευκαιρίε από φιλελευθερωποίηση είναι μεγαλύτερες από τους κινδύνου για την Ευρώπη. Ο λόγος είναι ότι έχουμε πολύ πια διαφοροποιημένη προσφορά γαλακτοκομικών. Εμείς ως Ευρωπαίοι εναντίον των Αμερικανών από ό,τι αντίστροφα. Αντίστροφα όμως θα πρέπει να συνεχίσουμε να προστατεύουμε ορισμένα προϊόντα περιφερειακά. Είναι προ το συμφέρον μας αυτό και θα είναι αναγκαίο να έχουμε υψηλότερα επίπεδα. αυτά τα υψηλότερα επίπεδα προδιαγραφών και προστασίας δεν θα πρέπει να τα εγκαταλείψουμε κατά διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε καθηγητά. Και τώρα ο κύριος Σιέτα Φανκέιν Πέμα, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Γαλλό. Να ευχαριστήσω τον ε, καθηγητή Ευσέν για τα αισιόδοξα λόγια του. Παρακαλώ. Thank you very much for the opportunity for European... Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που δίνετε στο European Milk Board να σας περιγράψει τις προοπτικές του κρατικού τομέα. Στο άρθρο 39 της Συνθήκης Λισαβόνας διατυπώνονται ρητά οι στόχοι της γαλακτοκομικής πολιτικής να διασφαλιστεί ένα δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες, ιδιαίτερα μέσω της αύξησης των εισοδημάτων του κάθε γεωργού και της σταθεροποίησης των αγορών. Οι διακυμάνσει των τιμών και πολύ χαμηλέ τιμέ που βλέπουμε σήμερα και το είδαμε και το 9 είναι αποτέλεσμα όλης της παραγωγής χωρίς να λαμβάνεται, που, όπου δεν λαμβάνουμε υπόψη τη ζήτηση. Έχουμε πολύ λίγα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε την κρίση των τιμών στο γαλακτοκομικό τομέα. Αυτό που χρειαζόμαστε τουλάχιστον είναι ένα εργαλείο για να αντιμετώπιση των τρομερών διακυμάνσεων και που το οποίο να κινητοποιείται μόνο σε περίπτωση κρίσης. Αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή είναι η δυνατότητα να αναγνωριστεί η ύπαρξη της κρίσης γιατί δεν έχουμε ορισμό. Τι θεωρούμε κρίση. Μερικοί θεωρούν ότι οι τιμές των γαλακτοκομικών είναι επαρκής δείκτης αλλά παίζουν εξίσου σοβαρό ρόλο και άλλοι παράγοντες. Θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένας δείκτης που να παίρνει υπόψη του όλους τους παράγοντες της αγοράς. Αυτό χρειαζόμαστε. Και αν ο δείκτης ξεπερνάει το 100 τότε να, κινητοποιείται ένα πρόγραμμα ή μηχανισμός. Αν όμως απ' την άλλη δεν καλύπτεται ούτε το, δεν καλύπτεται ούτε το κόστος τότε να αρχίζει ένα πρόγραμμα υπευθυνότητα των αγορών σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση έγκαιρη προειδοποίηση. Αν ο δείκτης πέσει κατά 7,5% θα γίνεται μια ανακοίνωση προειδοποίηση και μέχρι να επιστρέψει στο 100 ο δείκτης θα διατηρείται αυτή η φάση. Δεύτερη φάση. Πέφτει ο δείκτης κάτω από 15%. Η κρίση ορίζεται ως υπάρχουσα επισήμως και αρχίζουν να κινητοποιούνται τα κύρια στοιχεία του προγράμματος υπευθυνότητας των αγορών. Οι παραγωγοί μειώνουν, την παραγωγή τους κατά τουλάχιστον 5%. Όποιος δεν συμμορφώνεται πληρώνει έναν ειδικό φόρο ή πρόστιμο μάλλον. Εάν η κρίση συνεχίζεται παρά τα μέτρα αυτά και τις υποχρεωτικές μειώσεις, τότε για συγκεκριμένη περίοδο όταν ο δείκτης πέσει κάτω από 25% εφαρμόζεται η τρίτη φάση. Όλοι πρέπει να μειώσουν την παραγωγή τους κατά 2 και 3% για την καθορισμένη αυτή περίοδο. Και αν συνεχίσει η επιστροφή προς το 100% και είναι όλα τα άλλα στοιχεία θετικά μπορεί να θεωρηθεί ότι τελείωσε η κρίση. Μέχρι σήμερα όλα τα τότε όλα τα μέτρα περιορισμού της παραγωγής σταματούν και βλέπετε εδώ τις διάφορες γραφικές παραστάσεις. Κάτω από το μπλε είναι η κρίση όπου ο παραγωγός μπορεί να παραγάγει τα ίδια, να παραγάγει περισσότερα πληρώνοντας πρόστιμο ή να μειώσει την παραγωγή του και τότε να έχει κάποιο μπόνους. Όταν το πρόστιμο στη δεύτερη φάση παρα... καταλήξει συνθετικά αποτελέσματα, μπορεί κανείς να αλλάξει την παραγωγή του. Αυτό το είδαμε από μελέτες. Φέτος συσχύει ακόμη ο υπερφόρος. Αλλά αυτό καταστρέφει όπως βλέπουμε τους γαλακτοπαραγωγούς και βλέπουμε από τις τιμές ότι αρχίζουν να ανεβαίνουν. Αυτό είναι σωστό. Σωστό λοιπόν μέτρο το πρόστιμο ή ο υπερφόρος. Τώρα για να λειτουργήσουν όλα αυτά κανονικά πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί το παρατηρητήριο που οργανώθηκε σε ενωσιακό επίπεδο. Η λειτουργία του κανονίζεται εκ των προτέρων από ορισμένα κριτήρια. Λαμβάνονται αποφάσεις με βιώσιμο και διαφανή τρόπο χρησιμοποιώντας τον δίκτυ που είναι η βάση όλων των αποφάσεων. Αλλά επίσης απαιτείται και ένα νομικό υπόβαθρο που να μπορεί να εφαρμοστεί σε ολόκληρη την Ένωση και δεσμευτικά σε ολόκληρη την Ένωση. Ό,τι αφορά τις, το ύψος της παραγωγής θα το αναλαμβάνουν οι παραγωγοί. Σύμφωνα με την αρχή όποιος μολύνει πληρώνει. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει εξοικονόμηση πόρων για την απαραίτητη αποθήκευση. Βασιζόμαστε λοιπόν σε διάφορα κριτήρια. Οι τιμέ δεν είναι επαρκέ γιατί καθυστερούν μερικού μήνε πάντοτε. Χρειάζονται περισσότερα στοιχεία και αριθμοί μεταξύ των οποίων και το κόστος παραγωγής. Μόνο τέτοιου είδους δεδομένα μας δίνουν μια, ένα βιώσιμο δίκτυ. Το πρόγραμμα υπευθυνότητα των αγορών έχει πολλά ωφέλη σε σύγκριση με άλλα προγράμματα. Παραδείγματο χάρη μπορεί να αποφευχθεί η καταστροφή των τιμών. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η έννοια αυτή βασίζεται στη συμπεριφορά των γαλακτοπαραγωγών που πρέπει να συμφωνεί με τις συνθήκες της αγοράς. Στο μέλλον τα αγροκτήματα θα πρέπει να παρατηρούν συνέχεια τις εξελίξεις της αγοράς και να αντιδρούν στις αλλαγές, ιδιαίτερα σε κρίσεις. Τέτοια συμπεριφορά, επιχειρηματική συμπεριφορά, μέχρι στιγμής δεν εφαρμοζόταν και αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί θα αλλάζουν την παραγωγή τους ανάλογα με τη ζήτηση αλλά επίσης θα έχουν συνυπευθυνότητα για αν συμπεριφορά αντιαγοράς και υπάρχουν και οι λεγόμενοι free riders που κάθε φορά μας καταστρέφουν τις προσπάθειές μας από την άλλη φορά, αν είναι θεμητό φυσικά σε περίπτωση κρίσης να δοθεί και κάποια στήριξη. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν τα αγροκτήματα να πιστούν να συμμορφωθούν εθελοντικά. Κάθε φορά βέβαια πρέπει να πληρώνουν και το λογαριασμό αυτά που χρωστάνε σε τράπεζες μπορεί να μην έχουν τα μέσα να μειώσουν την παραγωγή τους μπορεί να είναι αναγκασμένοι και να αυξήσουν την παραγωγή για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους είναι λοιπόν αδύνατον να πούμε ότι με χαμηλές τιμές μπορεί κάποιος μερικές φορές να διασφαλίσει το εισόδημά του Αλλιώ θα ήταν ο νόμος της Ζούγκλας το πρόγραμμα η υπευθυνότητα των αγορών είναι πολύ διαχειρίσιμο και μπορεί να βασιστεί στα υπάρχοντα στοιχεία που τα έχει ήδη η Κομισιόν, αρκεί να συνδυαστούν. Συνοπτικά, το πρόγραμμα υπευθυνότητα των αγορών επομένως μπορεί να περιγραφεί ως τελείως βασισμένο στην αγορά. Ξέρω ότι η παρουσίασή μου ήταν συντομότατη, έχω όμως και άλλα στοιχεία και φέιγ βολάν αν θέλετε για να σας τα εξηγήσω οποτεδήποτε χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Θα καλέσω τώρα τον κύριο David Dobbin υπεύθυνο και διευθυντή της Ένωσης των Γαλακτοπραγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου. Αν θέλετε... Όχι, με συγχωρείτε. Προηγουμένως ο κύριος Βενσόν Σατελιέ. από το Εθνικό Ίδρυμα της Γεωπονικής Έρευνας. Châtelier, Vincent Châtelier. Merci. Merci, Président. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην σύντομη παρουσίαση που θα κάνω, θα σας διαθέσω, θα προσθέσω ένα άρθρο για όσου το επιθυμούν, για την κατάσταση του γαλακτοπορεγωτικού τομέα στην ε, Γαλλία και για το πόσο ποικιλόμορφο είναι, εφόσον έχουμε σωστά αυτές τις απορίες για το μέλλον του τομέα. Ο ίδιος ο τομέα ανησυχεί. Για να δούμε την παραγωγή της Γαλλίας λοιπόν στο γάλα αυτή τη στιγμή πρέπει να λάβουμε υπόψη το μεταβαλλόμενο τοπίο με ή χωρίς μηχανισμούς ποσόστοσης, με ή χωρίς ε, τη, τα εργαλεία της αγορές υπάρχει αναδιάρθρωση των εκμεταλλεύσεων 4-5% ετησίως. Έχουμε 68.000 ε, γαλακτοπραγωγικές μονάδες στη Γαλλία. ραντεζόμαστε ότι γύρω στο 2025 θα έχουμε 40.000. Μιλάμε για τη γεωργία που αναγεννάται. Το γάλα στη Γαλλία ε, προέρχεται από εκμεταλλεύσεις ε, συνεταιριστικές και η ανάπτυξη μεγάλων μονάδων παραγωγής γίνεται με σχετικά αργή ταχύτητα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 16% του συνολικού ζωικού κεφαλαίου γαλακτοπαραγωγών αγελάντων ε, στη Γαλλία με 100 Αγελάδε ε, ισοδύναμο. Έχουμε πολύ μεγάλε διαφορέ μεταξύ των περιφερειών, όχι εδώ και πέντε, αλλά εδώ και δέκα χρόνια και το γάλα συνήθω πάει από τον νότο τη Γαλλία προ τα βορρά και όχι από τα ανατολικά μόνο, αλλά από το σύνολο των περιοχών τη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένων όσων ε, έχουν προσανατολιστεί στην παραγωγή δημητριακών. Έχουμε ενισχυμένη στήριξη τη γαλακτοπαραγωγή ε, στι περιοχέ που ήδη παρήγαν γάλα και αυτή τη στιγμή έχουμε και διαφορά στην οργάνωση τη εργασία ε, σε περιοχές ορεινές ή παιδινές και αυτό ε, επηρεάζει και το εισόδημα. Υπάρχει, υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, στην, ε, στο μοντέλο της παραγωγής γάλακτος λόγω των διαφόρων μεθόδων παραγωγής διότι υπάρχουν στις ορεινές περιοχές ελλείψεις ως προς τις ζωοτροφές και, επειδή, και την παραγωγή τους και επειδή στη Γαλλία έχουμε μεγάλες ομίλους, συνεταιρισμούς, αλλά και μεγαλύτερες εταιρείες. Χρειάζονται λοιπόν εδώ συγκεκριμένες λύσεις, αλλά που να γίνουν και αποδεικτές επιτόπου. Τώρα, για την ε, ε, χρηματοδότηση των γαλακτοπραγικών μονάδων, που είναι καθοριστικό για την ερχόμενη δεκαετία. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι το πλαίσιο στήριξης των γαλακτοπραγωγικών μονάδων δίνει αποτελέσματα κυρίως γιατί ε, έχει θετική δυναμική η διεθνής αγορά και επειδή υπάρχουν πραγματικέ δυνατότητε ανάπτυξη τη εκμεταλλεύση. Έχουμε επίση χαμηλά επιτόκια, οπότε πολλέ εκμεταλλεύσει σήμερα επενδύουν. Η πρόσβαση στην χρηματοδότηση δεν είναι πάντοτε απλή. Πρέπει να διακρίνουμε, ακόμη και σε συνθήκε κρίση, την έννοια τη στήριξη ναι. των περιοχών παραγωγών σε περίοδο διακύμανσης των τιμών, δηλαδή την ανάγκη του ταμείου τους, τις ανάγκες του ταμείου τους και μετά τη χρηματοδότηση των διευθυντικών αλλαγών. Ε, το ποσό του, το κόστος ε, της ε, στήριξης των μονάδων παραγωγής είναι αυτή τη στιγμή πολύ γοργά αυξανόμενο, διότι οι γεωργοί που πιστεύουν στο μέλλον, οι κτηνοτρόφοι που πιστεύουν στο μέλλον, χρεώνονται πολύ, μάλλον προχωρούν πολύ γρήγορα, αν και το ποσοστό χρέωσής τους είναι πολύ χαμηλό. Η χρηματοδότηση Κατάρτιση προγραμμάτων λοιπόν γίνεται σε εκμεταλλεύσει και σε συνθήκε που είναι κάποιε φορέ μέχρι και ακροβατικέ θα μπορούσε να πει κανεί. Έχουμε πολύ μεγάλε λοιπόν αγορέ αυτή τη στιγμή ω προ το κεφάλαιο που συγκεντρώνουν οι εκμεταλλεύσει. Επίση ε, το κατά πόσο αναπτύσσεται ε, ε, η δυνατότητα μίσθωσης γεών ε, γιατί η νέη παραγωγή δεν ε, επενδύουν στα ακίνητα και επίσης πολύ μεγάλες αλλαγές σε σχέση με την τελευταία δεκαετία. Ποια είναι τα εργαλεία που χρειάζονται αυτή τη στιγμή. Πολλά έχουν ε, υποθεί, τιμές παρέμβασης και οι εξαγωγικές επιστροφές είναι εργαλεία του παρελθόντος, παροχημένα. Κάθε φορά λοιπόν που υπάρχει μια κρίση προσπαθούμε να καινοτομήσουμε με παλιά εργαλεία, αλλά προσοχή, προσοχή, διότι το μήνυμα είναι ότι η μεταρρύθμιση τη ΚΑΠ εδώ και 10 χρόνια έχει δώσει μείωση των τιμών παρέμβαση με κάποια σταθεροποίηση πλέον, αλλά το μήνυμα από τι Βρυξέλλε τώρα είναι αυξήστε τι τιμέ για να ξεφύγετε. Νομίζω ότι στην πράξη θα υπάρξουν δυσκολίε. Δεν νομίζω ότι η αύξηση των τιμών παρέμβαση είναι το Α και το Ω, η πανάκια για την ε, μελλοντική επιτυχία του γαλακτοπαραγωγικού τομέα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη στήριξη των εξαγωγών και με τη ρωσική κρίση, καταλαβαίνουμε ότι ακόμη και προσωρινά και ίσω και με την συγκατάθεση του ΠΟΕΝ μπορούσε αυτό να ε, λειτουργήσει. Όμω υπάρχουν και άλλα εργαλεία που πρέπει να συζητηθούν. Είναι πολύ δύσκολο να έχει κανεί ε, τελείω αυτέ τι ιδέε, διότι δεν έχει ακόμη και αρκετή εμπειρία στα χέρια του για να δει όλε οι καινοτόμε λύσει που έχουν ε, επιχειρηθεί στο πακέτο του γάλακτο, τι αποτελέσματα έχουν δώσει. Αυτό που, δεν είναι βέβαιο, που είναι βέβαιο είναι ότι τιμή της κατανάλωσης των γαλακτικών προϊόντων στην Γαλλία σε σχέση με άλλες ε, ευρωπαϊκές χώρες είναι υψηλό. Δηλαδή ε, ο καταναλωτής δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει πάντοτε το κόστος ε, χάρη στις επιδοτήσεις της ΚΑΠ. Από το αποθεματικό αντιμετωπίσεως της κρίσης, από τη διαφοροποιημένη οργάνωση των συνεταιρισμών, αυτά όλα μπορεί να ενθαρρύνουν μια παραγωγή πιο δυνατή Μακροπρόθεσμα όμως αν πιστέψουμε στι οργανώσει των παραγωγών, πρέπει να είμαστε ταυτόχρονα και ρεαλιστέ ω προ του αριθμού. Λόγω χάρη στην Γαλλία, 46 οργανώσει παραγωγών συγκεντρώνουν 17% του όγκου παραγωγή. Δηλαδή δεν είναι μεγάλο μέρο τη παραγωγή, είναι ένα μόνο τμήμα τη. Αλλά μην ξεχνάμε ότι οι καινοτομίε μπορεί να γίνουν τα ερχόμενα χρόνια σε αυτό το χώρο. Επίση, πρέπει να βρούμε ένα σύστημα ασφάλιση, να προσαρμόσουμε και είναι πολύ σημαντικό, ακόμη και αν το ε, μετατοπίζουμε αυτό στι εθνικέ πολιτικέ, τη φορολόγηση των εταιριών για να μπορέσουν να εξοικονομήσουν τα καλά χρόνια των παχιών αγελάδων ακόμη περισσότερα. Επίσης πρέπει να ε, φροντίσουμε την ε, γεωργική ανάπτυξη. Δεν υπήρξαν αρκετά κονδύλια στην τελευταία ΚΑΠ για την στήριξη των γαλακτοπαραγωγών που είχαν το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής. Ε, η διαφοροποίηση του κόστους είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που να δείτε κάθε φορά που υπάρχει μια κρίση. Δηλαδή ποιοι είναι οι παραγωγοί που θα καταφέρουν να την γλιτώσουν. Εδώ λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε και για την εκτροφία στα ορεινά. Στην περίπτωση τη γνωρίζω καλά, υπάρχουν πολλές περιοχές σε υψόμετρο που στηρίχθηκαν από τους μηχανισμούς της ΚΑΤ. Όχι μόνο με την τελευταία μεταρρύθμιση, ε, και με τα εργαλεία της ΚΑΠ, αλλά υπήρξαν αποφάσεις εξαετίας, επταετίας από ό,τι ξέρω, να μεταφερθούν δημόσια κονδύλια προς όφελος της ορεινής γεωργίας. Είχαμε αυτή τη δυνατότητα, χρησιμοποιήθηκε η δυνατότητα αυτή και έχει δώσει θετικά αποτελέσματα. Όμως έχει δημιουργήσει ένα γαλακτοπαραγωγικό τομέα με δύο κεφαλές, δηλαδή εξαγωγές και άμεσες ε, βοήθειες ε, στι ορεινέ περιοχέ με 100% κατανάλωση των κομιλίων και 50% για όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε αυξήσει την εξάρτηση δηλαδή από τι επιδοτήσει. Δεν θα ε, μιλήσω τώρα για τι ε, τυροκομικέ περιοχέ και την ιδιαίτερη προστασία του. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν από άποψη πραγματιστική. Στη Γαλλία τουλάχιστον πρέπει να ε, ομογενοποιήσουμε την ε, το, την ενιαία πληρωμή, το δικαίωμα στις ενιαίες πληρωμές για τις ε, γαλακτοπαραγωγικές μονάδες. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι χρήσιμες γεωργικές επιφάνειες και το σύνολό τους, τα κονδύλια να, κατα, να κατευθυνθούν στην εξυγχρονισμό των κτηρίων και των υποδομών στις ε, μειονεκτούσες περιοχές που έχουν δυσκολίες αγοράς ε, πρέπει επίση να δούμε τι θα γίνει με τα μοντέλα παραγωγή στι ορεινέ περιοχέ και να ενθαρρύνουμε, και αυτό δεν είναι απλό, να ενθαρρύνουμε τι εξαγωγέ τύρου που είναι ποιότητα σε ε, περιοχέ εκτό τη Γαλλία. Αυτή τη στιγμή μικρό μερίδιο των προϊόντων ποιότητα, που είναι πολλά, φτάνει σε επίπεδο εξαγωγών. Ε, εδώ λοιπόν πρέπει να αυξήσουμε το ανώφλι της στήριξης των νέων παραγωγών σε ορεινές περιοχές, αλλά και την ανάπτυξη των, ε, του ζωικού κεφαλαίου γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων, διότι στις ορεινές περιοχές, στη Γαλλία, πολλές φορές συνεπάρχουν ο τομέας του γάλακτος και ο τομέας του εδώ πέρα ε, πρέπει να δούμε σε τοπικό επίπεδο τι ε, μετατοπίσεις μπορεί να γίνουν ως προς τις εξαγωγές και τη σχέση μας με τον έξω κόσμο. Δεν θα υπάρχει αύξηση της παραγωγής του γάλακτος στη Γαλλία εάν δεν υπάρξει δυνατότητα εξαγωγής περισσότερων προϊόντων στις εξωευρωπαϊκές αγορές. Σε ό,τι αφορά τις αγορές της Γαλλίας, το εμπορικό συζύγιο ε, της χώρας έχει σταθεροποιηθεί εδώ και 10 χρόνια. Δεν έχουμε κερδίσει κανένα τμήμα αγορά επιπλέον, ούτε στην Ευρώπη ούτε αλλού. Αλλά έχουμε βελτιώσει τι εμπορικέ μα επιδόσει σε τρίτε χώρε. Είναι πολύ θετικό. 2,4 δι με δύο γραφήματα πολύ γρήγορα. Σα δείχνω εδώ τι γίνεται στην Κίνα. Σα δείχνω την εξέλιξη των εξαγωγών ε, γαλακτοκομικών προϊόντων προ την κινέζικη αγορά. Και φαίνεται ότι εξάγουμε πολύ παιδικό γάλα και πολύ. Ε, και, και, γάλα, και ορό γάλακτος επίσης. Στο παιδικό ε, γάλα και στο γάλα σε σκόνη βλέπουμε να υπάρχει καλύτερη πώληση από ότι λόγου χάρη παραδοσιακά τυριά που προβλέπονται καλύτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για να ολοκληρώσω ποιο είναι το πρότυπο που πρέπει να προωθήσουμε. Κοίταξα όλα τα στοιχεία και όλα τα επιστημονικά κείμενα και δεν είναι καινούργιες αυτές οι απορίες. Απλώς μια κουβέντα αναχώρα. Η Νέα Ζηλανδία, αυτό που με ευνηδίασε είναι η δυνατότητά του σε 10 χρόνια να παράγουν 10 τόν γάλα παραπάνω ε, χωρίς περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η Ελβετία, δεν είναι γαλακτοκομικό πρότυπο, δεν παράγει ούτε όσο η Μεγάλη Βρετανία. Είναι μια πολύ μικρή χώρα για να δούμε πώς θα μπορούσε να ε, εφαρμοστεί αυτό σε 50 εκατομμύρια τόνους γάλα. Αλλά αυτό που ήταν ε, σημαντικό για όσους γνωρίζουν τις λεπτομέρειες είναι πώς μετατράπηκε η χώρα αυτή. Μεταβλήθηκε τελείως μέσα σε μια 20 ετία και ο Καναδάς που είναι ένα συστηματικό παράδειγμα ε, είναι μια χώρα μικρή, ένας μικρός παραγωγός, ε, με έλλειμμα στο γάλα, αλλά έχει τη γοητεία της ικανότητας που προσέφερε στους γαλακτοπαραγωγούς, μιας τιμής γάλακτος, περισσότερο προσωδοφόρας με μια αγορά πιο ελεγχόμενη. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ε, ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι ασφάλειες λειτουργούν στις Ηνωμένες Πολιτείες στι Ηνωμένε Πολιτείε του προσεχεί μήνε, θα δούμε ακριβώ τι θα γίνει. Δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να έχουμε μια αρνητική θετική αποτίμηση του όλου συστήματος. Πρέπει απλώς να δούμε. Ένα, ότι η βούληση των ε, γεωργών εκεί ήταν ε, προς αυτή την κατεύθυνση και επίση τι προβλέπει ο προπολογισμό σχετικά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Σας είχα εμπιστοσύνη γιατί είπατε ότι τελειώνατε και δεν χρειάστηκε, δεν χτύπησα το σφυράκι. Τέλος πάντων σας ευχαριστώ πολύ. Όπως έχει ανακοινωθεί ο κύριος David Tobin από τις United Dairy Farmers του Ηνωμένου Βασιλείου. Μπορείτε να αρχίσετε σας παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Είμαι διαχειριστής ενός γαλακτοκομικού συνεταιρισμού με πάνω από 50 γαλακτοπαραγωγούς από την Ιρλανδία και την Αγγλία που παράγουν ένα δισεκατομμύριο λίτρα γάλακτος το χρόνο. Την διεύθυνση την έχουν αναλάβει οι γεωργοί και έχουμε έναν απλό στόχο να δημιουργήσουμε κερδοφόρες επιχειρήσεις και βιώσιμο δικαίωμα με βιώσιμες τιμές, εισόδημα με βιώσιμες τιμές. Μία από τις εγκαταστάσεις μας μεταποίησης είναι ιδιαίτερα μεγάλη και οι άλλες 7 ε, είναι εταιρείε που εξυπηρετούν τοπικές αγορές. Ολόκληρη την τροφιμική αλυσίδα καλύπτουμε, όχι μόνο την παραγωγή. Θέλουμε αποτελεσματικούς γεωργούς και αποτελεσματική μεταποίηση και διανομή επίσης αποτελεσματική. Μεταποιούμε το γάλα σε τυρί, ένα τρίτο σε βούτυρο και σε άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα, γιαούρτια κλπ. 45 χώρες, σε 45 χώρες πουλάμε, εκτός Ένωσης ιδιαίτερα, οι περισσότερες στη Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική ή στην Κίνα, και την Άπο Ανατολή. Παλαιότερα πουλούσαμε και στη Ρωσία, αλλά τώρα μας έχει, έχει κλείσει αυτή η αγορά για μας. 80% της παραγωγής μας εξάγεται, διότι έχουμε πολύ μικρή χώρια αγορά. Επομένως υφιστάμεθα τις συνέπειες των αλλαγών από τη διεθνή αγορά, όπως και οι υπόλοιποι γαλακτοπαραγωγοί στην Ευρώπη. 27 here. Hopefully it won't fall further. 27 λεπτά. Γιατί είναι σε αυτό το επίπεδο η τιμή, διότι ο δείκτης της Ένωσης των Γαλακτοπαραγωγών δείχνει ότι συνδυάζει διάφορα, διάφορους δείκτες από την παραγωγή, ένα καλάθι το οποίο είναι λίγο χαμηλότερο από την τιμή που πληρώνουμε Πολλοί γνωρίζετε τον κύκλο της γαλακτοπαραγωγής που βασίζεται στην παραγωγή, όχι στη ζήτηση η οποία μέχρι στιγμής ήταν αρκετά σταθερή, αλλά τώρα βλέπουμε κάποιες αυξήσεις, εκτός βέβαια από το κλείσιμο της ρωσικής αγοράς και τη μείωση της κινέζικης. Οι διακοιμάνσεις των τιμών πριν αρχίσει η Ένωση να καταργεί τα διάφορα μέτρα που έλαμβανε, η αγορά ήταν σχετικά σταθερή και μετά από το 2006 και 2007 όταν καταργήθηκαν οι επιστροφές προς τις εξαγωγές και άλλα η αγορά στην αρχή κινήθηκε πολύ, πάρα πολύ το 2007 και μετά ακολουθήθηκε αυτό από τεράστια ύφεση στην αγορά. Το ενδιαφέρον ήταν ότι τότε υπόθηκε ότι έπρεπε εφόσον υπάρχει κρίση να επιστρέψουμε στις επιστροφές για τις εξαγωγές. Και αυτά τα μέτρα λήφθησαν το 2009 και αυτό βοήθησε στη σταθεροποίηση μιας πολύ σοβαρής κατάστασης της αγοράς, παρόμοιας με την τωρινή. Η ενωσιακή πολιτική σημαίνει ότι αν κάνουμε υπερπαραγωγή θα πέσουν οι τιμές για τους γεωργούς σε όλη την Ελλάδα και θα μειωθεί το εισόδημά τους. Στην πραγματικότητα όμως στον κύκλο αυτό. Αν θέλουμε σταθερές τιμές τότε πρέπει να ελέγξουμε και την παραγωγή, όχι μόνο τη ζήτηση. Στο παρελθόν υπήρχαν πωλήσει γαλακτοπαραγικών προϊόντων από τη Νέα Ζηλανδία που ήταν πολύ φθηνότερα από τα ευρωπαϊκά. Σήμερα όμως τα μαθαίνουμε όλα αμέσως δηλαδή οι αγοραστές μας στη διεθνή αγορά γνωρίζουν αμέσως τις τιμές μας παγκοσμίω. Και άρα δεν μεταφέρονται οι τιμές μόνο μεταξύ περιφερειών αλλά και από διάφορους τομείς μεταξύ τους. Πολύ γρηγορότερα από ό,τι παλαιότερα διότι είναι πολύ πιο ανοιχτά και διαφανή όλα. Μετά τις ε, επιστροφές λοιπόν και τώρα τις ποσοστώσεις υπάρχει πολύ μεγαλύτερη διακύμανση των τιμών. Η τιμή ελέγχει κυρίως την παραγωγή. Τα συμβόλαια μπορεί να παίξουν ένα θετικό ρόλο για τους γεωργούς αλλά μειώνουν, αμβλύνουν την μεταφορά των τιμών από τομέα σε τομέα. Άρα χρειάζεται πολύ καλύτερο έλεγχος τους και της παραγωγής όχι μόνο των τιμών. Για την εφαρμογή της αγροτικής δέσμης στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπήρχαν πολλές επιπτώσεις, κυρίως ή τα σταθερά συμβόλαια με τους γεωργούς αλλά ως προς την ε, προστασία της ε, ετικέτας προέλευσης αυτό δεν έφερε καμία αρχή. Υπάρχει όμως η αρχή μιας σταθεροποίησης και φαίνεται με κάποια μεγαλύτερη σταθερότητα αν όχι και άνοδος. Ξέρουμε ότι η τωρινή κρίση οφείλεται στην υπερπαραγωγή εν μέρει λόγω του καλού καιρού και εν μέρει λόγω υψηλότερων τιμών πέρυσι. Πράγματι μειώθηκε λίγο η παραγωγή, αλλά όσπως έχει σήμερα, τον περασμένο μήνα ας πούμε, είναι πολύ περισσότερη από τη ζήτηση. Στην Ένωση εξάγουμε 9 με, 10, με 11% της παραγωγής μας και πρέπει να βρούμε κάποια αγορά για όλα αυτά έξω από την Ευρώπη. Και οποιαδήποτε μελλοντική ανάπτυξη του τομέα θα βασίζεται στις εξαγωγές. Άρα θα πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί διεθνώς και για τις τιμές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ένα δεύτερο θέμα, το νομισματικό. Θα πέσουν ακόμη περισσότερο οι τιμές του γάλακτος γιατί τα συμβόλαια στην Ευρώπη εκφράζονται σε ευρώ. Στην Ευρώπη βλέπουμε σχεδόν σε κάθε χώρα τους τελευταίους έξι μήνες Χωρίς τις ποσοστώσεις οι περισσότερες θα αναπτυχθούν, θα αυξηθούν γιατί παράγουν μέχρι το επίπεδο των ποσοστώσεων. Η Ιρλανδία είναι εκείνη που είναι πιο γνωστή ως υπόδειγμα αλλά και η Γερμανία έχει μεγάλη παραγωγή και χρειάζεται και με μικρή μόνο αύξηση να δημιουργηθούν, δημιουργούνται αποθέματα. Πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν λοιπόν όλα αυτά Χρειάζεται πιο διαφανής και αποτελεσματική αγορά επιπροθεσμία ώστε να μπορεί να καθοριστεί μια δίκαια τιμή. Αυτές οι αγορές επίσης θα βοηθήσουν στην προώθηση των προϊόντων και στη μείωση του κινδύνου. Υπάρχουν δυνατότητες να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά ακόμη δεν είναι, είναι σε πρώιμο στάδιο. και δεν το εμπιστεύονται ακόμη το σύστημα αυτό η παραγωγή. Πρέπει επίσης να αντικατασταθεί η ρωσική αγορά. Πρέπει δηλαδή να βρούμε κάποια αγορά για τα τυριά μας και ακόμη δεν έχουμε βρει. Ένας τομέας που θα μπορούσε να τον εξετάσει η Κομισιόν για την αγορά νέων, θα ήταν και η αγορά νέων αγορών ή προτιμησιακές συμφωνίες με χώρες σαν την Κίνα. Εξάγουμε στην Κίνα αλλά είναι πολύ χαμηλότεροι οι δεσμοί στην, για τη Νέα Ζηλανδία. Χρειάζεται εδώ κάποια ισονομία. Επίσης πρέπει τα συμβόλαια να μην ε, αφορούν μόνο τους μεταποιητές, αλλά και την προμήθεια των πρώτων υλών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει μια ειδική υπηρεσία για τα λαχανικά αλλά δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τα γαλακτοκομικά εδώ θα μπορούσαμε να εμπνευστούμε με την έννοια των βελτίστων πρακτικών. Τέλος για την τιμή παρέμβασης προς στιγμήν δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει παρέμβαση αλλά ότι η τιμή παρέμβασης αποτελεί μια βάση. Θα μπορούσε δηλαδή να παίξει ένα ρόλο χωρίς πραγματική αληθινή παρέμβαση. Τέλος θα μπορούσε να υπάρξει ένα σύστημα που διαχειριζόμαστε τα περιθώρια και όχι την καθαρή τιμή. Αυτό ίσως είναι ένας δρόμος για το μέλλον και νομίζω ότι θα εφαρμοστεί μόνο με τη συνεργασία των πάντων μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί περιοριστήκατε στο χρόνο σας και για το ενδιαφέρον της παρουσίασής σας. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Άλφρεντ Έντερλε, γαλακτοπαραγωγό από τη Βαβαρία και πρόεδρο της Ένωσης Βαβαρών Γαλακτοπαραγωγών. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για την ατότητα που μου δίνετε να σας παρουσιάσω τη γνώμη ενός που ασχολείται αλλά και εκπροσωπεί τον κλάδο του αυτό σε περιφερειακό επίπεδο. Είμαι επίτιμο μέλος ε, του Προεδρίου της ε, Βαβαρικής ε, Οργάνωσης Γεωργών αλλά συμμετέχω και σε γαλακτοκομικές οργανώσεις σε επίπεδο του ΣΦΑΜΠΕΝ όπου συμμετέχουν 40 γαλακτοκομικά εργοστάσια και όλη η παραγωγή στην ε, βαβαρική Σουαβία. Το σύστημά μας ε, ισχύει εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε μία σημαντική ε, κατανομή σε τομείς της παραγωγής βουτύρου και τυριού στη Νότια Γερμανία. Η προηγούμενη συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για μας. Επίσης, ε, συμμετέχουμε στην ε, προσπάθεια να έχουμε τυριά συγκεκριμένα έμενταλ με ονομασία προέλευσης. Βέβαια είναι περιορισμένες οι ποσότητες της παραγωγής μας. Ως εκπρόσωπος ε, των παραγωγών προσπάθησα να διαθέσω αυτά τα προϊόντα όμως δεν υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον τώρα που λήγουν οι ποσοστώσεις να καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα αγοράζουν. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα πλευρά της συζήτηση. Αυτό μπορεί να ισχύει και για μεγαλύτερες περιφέρειες. Μου θέσατε ορισμένα ερωτήματα. Σας έθελα μια, σας μια αναλυτική γραπτή απάντηση. Ελπίζω να έχει κατανεμηθεί. Οπότε θα πω μόνο μερικά ε, πολύ ε, γρήγορα για τη συνέχιση της παραγωγής. Θεωρούμε ότι θα λήξουν οι καταστάσεις σε ορισμένες περιοχές θα αυξηθεί η παραγωγή ουσιοδός ιδιαίτερα όπου ήδη υπάρχουν οι δυνατότητες των εγκαταστάσεων και δημιουργήθηκαν αυτές οι νέες εγκαταστάσεις ακριβώς εν ώψη της κατάργησης των ε, ποσοστώσεων. Οι αυξήσει παραγωγή βέβαια ε, προκλήθηκαν επίσης από την αύξηση τη τιμή, όπου έγιναν πολύ υψηλές ε, επενδύσεις πρέπει να θεωρήσουμε ότι αν συνεχίσει η μείωση των τιμών τότε θα αξιολογηθούν όλα τα, ε, όλες οι δυνατότητες παραγωγής για να διατηρηθεί κάποια ρευστότητα. Αλλά αν συνεχιστεί η μείωση των τιμών τότε δεν θα, έχει επαρκή ρευστότητα, δεν θα έχουν επαρκή ρευστότητα οι εκμεταλλεύσεις. Από τα συμβόλαια που διαπιστώνουμε διαπιστώνουμε ότι υπάρχει πίεση επί των τιμών αυτό όμως δεν έχει να κάνει με την λήξη των ποσοστώσεων αλλά με γενικότερη μεταβλητότητα των τιμών και τα άλλα γενικότερα προβλήματα που ήδη αναφέρθηκαν Ρωσία, Κίνα κτλ. Συνολικά συμφωνώ με τους προηγούμενους ομιλητές, με ορισμένους, ότι μακροπρόθεσμα φυσικά έχει θετικές προοπτικές η αγορά παγκοσμίω και στο παρελθόν αποφασίστηκε. Ε, στο παρελθόν το διαπιστώσαμε αυτό. Δεν πρέπει βεβαίω όταν εξετάζουμε τις πιέσει επί των τιμών να κάνουμε επιλεκτική χρήση στατιστικών. Τα τελευταία χρόνια είχαμε πολύ θετικέ εξελίξεις παγκόσμιε αγορές, οπότε πρέπει να το δούμε συνολικά το θέμα. Και θεωρούμε επίσης ότι όταν θα αυξηθεί το κατακεφαλήν εισόδημα στις αναπτυσσόμενες χώρες θα αλλάξουν και οι διατροφικές συνήθειες, οπότε οι παραγωγοί μα θα έχουν περισσότερε δυνατότητε διάθεση των προϊόντων του. Δυνατότητε παρέμβαση τώρα, από πλευρά τη Ένωση. Βεβαίω είναι η τιμή παρέμβαση και η ιδιωτική αποθήκευση. Είναι σημαντικό τμήμα των προσπαθειών μας και επίση θα μπορούσαμε να έχουμε και ειδικά προγράμματα. Υπάρχει δυνατότητα στι χώρες που εθίγησαν από το ρωσικό εμπάρκο. Θα μπορούσαν να έχουμε στόχο προσιλωμένα προγράμματα Ταχύτατα βέβαια, χωρίς ε, πολλές συζητήσεις, η Κομισιόν θα πρέπει να δράσει για να βοηθήσει. Οι πιστώσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης πρέπει να προέρχονται από το γενικό προϋπολογισμό και όχι από τις άμεσες ενισχύσεις, γιατί αυτό θα ήταν στην ουσία, τα βγάζουμε από μια τσέπη, τα βάζουμε στην άλλη. Έχουμε περαιτέρω δυνατότητες να βοηθήσουμε τις ε, μεμονωμένες εκμεταλλεύσεις μέσω αυτών των προθεσμιακών συμβολέων. Αυτό θα ήταν σκόπιμο να γίνει γνωστό μέσω ε, εκστρατείας ενημέρωσης της Ένωσης. Πώς πρέπει να διαμορφωθούν οι δυνατότητες παρέμβασης. Ε, συμφωνώ με αυτά που είπε ο Σκόπα της Κόπα Κοζέκα. Ποια είναι τώρα η κατάσταση στη Γερμανία. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η αυξανόμενη συγκέντρωση της μεγάλης διανομής. Έχουμε πέντε μεγάλες ε, ε, εταιρείες σούπερ μάρκετ που ελέγχουν σχεδόν το 80% της αγοράς. Οπότε διαφορετικά αυτό δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Η Γερμανική Αρχή Καταπολέμηση των Μονοπωλίων το ανεγνώρισε και προσπαθεί να το αντιμετωπίσει. Το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η συγκέντρωση οδηγεί ότι μία μικρομεσαία επιχείρηση αν αποκλειστεί από έναν μεγάλο διανομέα δεν μπορεί πλέον να επιβιώσει. Και βεβαίως ε, μπορούν να παίξουν και μεγάλο ρόλο στην, στο καθορισμό των τιμών αυτή η μεγάλη διανομή. Και αυτό δημιουργεί πολύ αρνητικά φαινόμενα. Πρέπει λοιπόν να λυθούν πολιτικά μέτρα και μέτρα καταπολέμησης μονοπωλιακών καταστάσεων. Βεβαίως οι μειονεκτικές, οι μειονεκτικές περιοχές, εγώ ε, έχω σε δασική περιοχή 80 εκτάρια, προσπαθώ να έχω και κτηνοτροφική παραγωγή και γαλακτοκομική παραγωγή. Ξέρω λοιπόν τι λέω όταν μιλάω για μειονεκτικές περιοχές. Η πολιτική για την αγορά του γαλάκτος ε, μόνο εν μέρη μπορεί να βοηθήσει τη διατήρηση της παραγωγής. Χρειάζονται και άλλες συνοδευτικές πολιτικές για να αντιμετωπιστεί πλήρω το θέμα. Ήδη σε αυτέ τι περιοχέ σήμερα το πιο σύνηθε είναι ε, να υπάρχει ε, ε, δραστηριότητα διτή ή και τριπλή των γεωργών, να έχουν και άλλες δηλαδή δραστηριότητες για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Πρέπει λοιπόν να μας βοηθήσετε με τα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε οι νέοι εργαζόμενοι να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις ε, προκλήσεις σε αυτές τις ε, περιοχές. Δουλεύει κανείς πραγματικά με το αίμα της ε, ψυχής του. Πρέπει να είναι πεισμένος. Εάν δεν είναι πεισμένος, δεν είναι αποφασισμένος, δεν το κάνει. Άρα χρειάζεται να μειωθεί και η γραφειοκρατία. Αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ. Θα ενεθάρρυνε τους γεωργούς μας ή τουλάχιστον να μην υπάρξουν επιπλέον ε, γραφειοκρατικές επιβολέ. για παράδειγμα αυτή η απαγόρευση του να δένονται τα μοσχάρια Μα οδήγησε ε, πολλούς, μας οδήγησε σε, ιδιαίτερα πολλούς μικρούς γεωργούς που δεν μπορούσαν να χτίσουν επιπλέον στάβλους να εγκαταλείψουν την παραγωγή. Εάν συνεχίσουμε να επιβάλλουμε τέτοιες γραφειοκρατικές ε, υποχρεώσεις τότε θα συνεχιστεί η εγκατάλειψη των εκμεταλλεύσεων. Δεν είναι δυνατόν να επιβάλλουμε επιπλέον υποχρεώσεις συμπλήρωσης ερωτηματολογίων σε περιοχές που είναι τόσο μικρές εκμεταλλεύσεις. Επίσης και η οδηγία για τα οικοσυστήματα, τη χλωρίδα και την πανίδα μας δημιουργεί μεγάλα προβλήματα και ο τρόπος με τον οποίο καθορίζονται οι περιοχές ειδικού συμφέροντος επίσης δημιουργεί προβλήματα. Πρέπει να δώσουμε περιθώριο δράσης για το πώς θα καθορίζουν τις περιφέρειες τους. Και χρειαζόμαστε και τις πληρωμές από το δεύτερο πυλώνα. Η πλήρης ε, αποδέσμευση των πληρωμών αυτών το δεύτερο τομέα δεν μας βοηθάει ιδιαίτερα για τις μενοητικές περιοχές. Οι πληρωμές αυτές είναι σημαντικό τμήμα του δικτύου ασφαλείας. Το TTIP, οι δυνατότητες εξαγωγών στις ΗΠΑ αντιμετωπίζονται πολύ θετικά από τους μεταποιητές. Πρέπει λοιπόν να πιέσω να διατηρήσουμε τα επίπεδα προστασίας μας, τις προδιαγραφές μας, ιδιαίτερα για την γεωγραφική προέλευση και την προέλευση και την ελεγχόμενη προέλευση, προστατευόμενη προέλευση. Γιατί για τα θέματα αυτά οι καταναλωτές είναι πολύ ευαίσθητοι. Επίσης, μας ρωτήσατε αν μπορούμε να αξιοποιήσουμε το ελβετικό, το καναδικό και άλλα μοντέλα. Πιστεύω ότι δεν μπορούν να μεταφερθούν στη δική μας πραγματικότητα, γιατί η πραγματικότητά μας ε, περιέχει πολύ διαφορετικές καταστάσεις. Και αυτή η πολυμορφία της παραγωγής στην Ένωση είναι το κυριότερο πλεονέκτημά μας και πρέπει να εργαστούμε όλοι για να τη διατηρήσουμε και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να δώσω το λόγο στους βουλευτές. Πρώτα απ' όλα οι συντονιστές μας. Κύριε Ντες, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε Ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές που πήραν το λόγο σήμερα. Τι συμπεράσματα εξάγω. Δεν υπάρχει μία λύση που να ισχύει για όλους. Δεν υπάρχει. Εγώ είμαι από τη Βαβαρία. Η Βαβαρία παράγει γαλακτοκομικά όπως μόλις υπόθηκε και παράγουμε το διπλάσιο γάλα από αυτό που καταναλώνεται στο εσωτερικό μας. Τα 12,5 εκατομμύρια των κατοίκων μας. Άρα θα έπρεπε η μισή μας παραγωγή να εγκαταλείψει τις εκμεταλλεύσεις αν ε, βασιστούμε μόνο στην εσωτερική αγορά. Συμφωνώ λοιπόν με αυτό που είπε ο κ. Έντερλε. Δεν μπορεί να μας δώσει το κράτος λύση. Άκουσα τον Σάλφο Ταραμπέλα που αναφέρθηκε στα 25 λεπτά. Η δική μου ε, οργάνωση παραγών έλαβε 37 λεπτά πολύ πρόσφατα. Το 1995 στην Νότια Γερμανία, να φέρω ένα παράδειγμα, υπήρχε μια μεγάλη γαλακτοκομική ε, εγκατάσταση ήρθε ε, που αντιμετώπιζε μεγάλα προβλήματα. Άλλαξε η διοίκηση και έκανα πολλές επενδύσεις και τώρα πάει πολύ καλά. Άλλες το 95 που πήγαιναν πολύ καλά δεν επένδυσαν ε, τα κέρδη τους από την υψηλή τιμή των γαλακτοκομικών, δεν προσαρμόστηκαν πτώχευσαν όταν σήμερα μέσω των συνεταιρισμών είναι διατεθειμένοι να μην πάρουν πλήρως ε, το κέρδος τους για να γίνουν επενδύσεις από τις γαλακτοκομικές καταστάσεις για να διατηρηθεί ανταγωνιστικότητα επιτυχάνουν. Ενώ άλλοι που δεν είναι διτεθειμένοι να μειώσουν τα κέρδη τους ε, αποτυχάνουν. Καλύτερα λοιπόν να μην παρεμβαίνει το κράτος. Η αγορά μπορεί να τα ρυθμίσει. Τελειώνω, τελειώνω. Χρειαζόμαστε ε, βεβαίως μηχανισμούς για να αντιμετωπίσουμε κρίσεις. Δεν είμαι κατά της ε, ε, αύξησης της τιμής παρέμβασης. Πρέπει να μπορούμε να παρεμβαίνουμε ταχαίως. Μέσω της τιμής παρέμβασης από αυτό συμφωνώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε πολύ γρήγορα να ευχαριστήσω όλους τους εμπειρογνώμονες, ιδίως σε αυτό το δεύτερο πάνελ, μας έδωσαν ε, αφορμές για να συζητήσουμε και να μελετήσουμε και ο συνάδελφος Νίκολσον πιστεύω ότι θα εμπνευστεί από όσα άκουσε σήμερα το απόγευμα. Να ανακεφαλαιώσω εντός ενός λεπτού. Πρώτον, το πακέτο για το γάλα δεν έχει φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο. Το είπαμε επανειλημμένω εδώ στην Επιτροπή Γεωργία. Ήταν ε, ε, μια δεσμή μέτρων που έπρεπε να ασχοληθεί με αυτήν την προσγείωση, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Ε, καμιά φοβερή καινούργια αλλαγή. Ε, προγραμματισμός της παραγωγής των, ε, της τυροκομείας ήταν το μόνο μεγάλο σοβαρό εργαλείο αυτής της, αυτού του κανονισμού και αυτό δεν έδωσε τα πετούμενα αποτελέσματα. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε με την παραγωγή της Ευρώπης πώς θα την πάμε προς τα έξω που υπάρχει ε, ζήτηση. Εδώ έχει κουρεστεί η αγορά εντός. Οι μηχανισμοί πρέπει να μας αποσχολήσουν χωρίς να σκεφτούμε την επιστροφή στις ποσοστώσεις που δεν τις θέλει κανείς. Δεν τις θέλει κανείς γιατί η Ευρώπη θέλει να είναι μια περιοχή ανταγωνιστική και να δράξει τις ευκαιρίες της αγοράς ιδίως των αγορών του εξωτερικού εξωτερικού. Επ' αυτού νομίζω ότι υπάρχει γενικό συμφωνία. Το πρόβλημα όμω είναι εάν πρέπει να πάμε στο εξωτερικό, εκτό Ευρώπη και ενώ τι τρίτε χώρε, όταν λέω εξωτερικό. Ε, πρέπει να υπάρξουν μηχανισμοί ε, διαχείριση τη ε, προσφορά. Δηλαδή μια χώρα που παράγει 10% παραπάνω και δεν είναι σε θέση αυτό το 10% να το θέσει εκτό Ευρώπης σε εμπορία αυτό προκαλεί αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά και ναι. κυρίω ε, πλήττονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσει που δεν έχουν καμία ευθύνη. Ναι. Καμία ευθύνη διότι έχουν διατηρήσει το ίδιο επίπεδο παραγωγή. Οπότε το πρόβλημα είναι να βρούμε ένα μηχανισμό ευελιξίας με στόχου παραγωγή που να εγγυώνται στα κράτη-μέλη ε, ευέλικτο και όχι υποχρεωτικό τρόπο, αλλά να αξιοποιείται το εργαλείο αυτό, να ε, τους προσφέρουν κίνητρα ώστε ο στόχος της παραγωγής να επιτυγχάνεται. Όποιος δεν τον επιτυγχάνει, να αναλαμβάνει τις ευθύνες του με τον έναν τρόπο τον άλλο. Να φροντίζει να θέσει κάπου στην αγορά το προϊόν αυτό ή τέλο πάντων να καταβάλει ένα αντίτιμο. Ε, και δεν ξέρω πώ είναι εύκολο αυτό να μεταφραστεί σε νομοθετική πρόταση, σε νομοθέτημα. Δεν θα είναι απλό, αλλά η προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε εδώ είναι ακριβώ αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ω προ την εθελοντικό περιορισμό τη παραγωγή, η κατάσταση είναι παρόμοια με το πόσο θα πρέπει να περιορίσετε τι παρεμβάσει σα. Ναι. Ναι. Πρόεδρε, Συνήθως ακολουθώ τους κανόνες, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν η σειρά μου. Εκτός αν επιμένετε ότι θέλετε να με ακούσετε. Ε, φυσικά οι πράσινοι δεν θέλουν να με ακούσουν. Ξέρω πολύ λίγα για το European Milk Board, αλλά άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μας είπε η κυρία. Ότι αν παράγουμε πολύ γάλα θα καταστρέψουμε τις τιμές. Εγώ παράγω αυγά και μου είπαν ή να μειώσω τις τιμές ή να μειώσω την παραγωγή μου. Και μείωσα την παραγωγή μου για να έχω υψηλή τιμή. Αυτό έγινε για όλους τους παραγωγούς στην περιοχή μου και ασκήσαμε κάποια πίεση έτσι προς την ε, προμήθεια αλλά δεν ξέρω σε πόσες χώρες λειτουργεί αυτό το συμβούλιο, το board, πόσα λίτρα παράγεται και διακινείται. Θα με ενδιαφέρε να ξέρω τι έχει να μας πει ο κύριος David Dobbin για αυτά, γιατί έχει ένα συνεταιρισμό. Θα εγκρίνατε τέτοια μέτρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι εδώ και πολλά χρόνια συμμετέχω στις συζητήσεις για τα θέματα του γάλακτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά από τόσα χρόνια όλο τα ίδια ακούω όλο τα ίδια επιχειρήματα για να αιτιολογηθεί η πλήρης αλλαγή του τρόπου παραγωγής στην Ένωση. Και πού θέλουν να μας πάνε με αυτή τη φιλευθροποίηση. Στο μοντέλο που επισκέφτηκα επίσης το 2006 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τους μικρούς παραγωγούς που ήταν αυτοί που είχαν 100 αγελάδες και πήγαν να δούμε το βιομηχανικό μοντέλο παραγωγή γαλακτό, τεράστιες εκμεταλλεύσει, 8.000, 16.000 αγελάδε σε πολύ περιορισμένο χώρο, καταστροφή του περιβάλλοντο, ε, των υδάτων, του αέρα, μείωση τη απασχόληση ε, για τι μικρέ εκμεταλλεύσει των 100 αγελάδων και αυτό το βλέπουμε και τώρα, τώρα και εδώ. Όπω υπόθηκε πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Πρέπει να πούμε ανοιχτά ότι το θέμα είναι τι μοντέλο θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, παραγωγή γάλακτος. Και δύο ακόμη. Δεν θεωρώ στην εθελούσια προσέγγιση. Χρειάζονται κρατικές πολιτικές. Η πολιτική γάλακτος ε, συζητήθηκε σε υψηλό επίπεδο πριν από την τελευταία κρίση και εγκαταλείφθηκε αυτά που, εγκαταλείφθηκαν αυτά που προτείνονταν γιατί θα βάζαμε τα προϊόντα μας στο έλεος των κερδοσκόπων. Και αυτές οι εξαγωγές και οι επιστροφές για τις εξαγωγές νομίζω ότι είναι προσβολή για την ανθρωπότητα να λέμε τέτοια πράγματα. Και για το TTIP, εδώ πριν από λίγο στην Επιτροπή Γεωργίας ακούσαμε μία μελέτη όπου μας λέγανε ότι η Γεωργία ακριβώς θα ζημιωθεί από το TTIP. Ποιον κοροϊδεύουμε. Το TTIP το, θεωρούμε ότι είναι λύση για τα προβλήματα που έχουμε στο γαλακτοκομικό κλάδο έλεος να είμαστε ειλικρινείς και πρέπει να πούμε ανοιχτά τι μοντέλο θέλουμε για το μέλλον του γάλακτος στην Ευρώπη και ευχαριστώ πολύ. Housling. Καλά δεν ακούσαμε και πολύ διαφορετικά πράγματα. Αυτοί που είναι υπέρ της φιλευθερωπής της αγοράς ήρθαν και μας ξαναείπαν τα ίδια. Αυτοί που μιλάνε για τη φλευθεροποίηση θεωρούν ότι πρέπει επίσης να υποστηρίζουμε τους γεωργούς μας. Επειδή τους υποστηρίζουμε είναι ανταγωνιστική η γεωργία μας διεθνώς. Αν θέλουμε να παραμείνει στον ανταγωνισμό με τις ε, Ηνωμένες Πολιτείες και Νέα δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε, την υποστηρίζουμε. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Είπατε ότι ο γερμανικός οργανικός γάλακτος είναι θαυμάσιος. Μα δεν βλέπετε ότι μειώνονται οι γαλακτοπαραγωγοί συνέχεια. Τόσο θαυμάσιος είναι. είχαμε διατροτικές αλλαγές ε, τεράστιες, ακραίες και στη δική σας περιφέρεια. Θα καταστραφούν οι δομές εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Μόνο ένα άκουσα αυτό για έναν ευρωπαϊκό οργανισμό γάλακτος. Αυτό θα μπορούσαμε να το αναλάβουμε. Αλλά το συζητήσαμε για το πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει για το μέλλον. Για να ρυθμίσουμε την αγορά. Όλα τα άλλα για την φιλευθροποίηση, τα τροπάρια. Εμείς θα την πληρώσουμε αν υπάρχει πλήρης φιλοθροπής και μόνο που θα ωφεληθούν είναι τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Νταντά. Ευχαριστώ τους εκτό μας προσκεκλημένους σήμερα το απόγευμα. Κάποιοι συγκλίνουν στις απόψεις τους και νομίζω ότι εγώ μπορώ σε 4-5 σημεία αυτή τη σύγκληση όπως προέκυψε μέσα από τα θέματα που ε, αναλύθηκαν. Μια φοβερή πληροφορία. Ο, επίτροπος, ο εκπρόσωπο τη Επιτροπή μα μίλησε για τι τιμέ του γάλακτο το Δεκέμβριο. Δηλαδή, μεγάλη βελτίωση. Την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει για το τιμή του γάλακτο, είχαμε τρει μήνε ε, καθυστέρηση. Οπότε, να κάνω την εξή παρατήρηση. Ε, το παρατηρητήριο. Το παρατηρητήριο και η γνώση τη αγορά είναι ένα θέμα που ήδη ε, έχουμε επιτελέσει μεγάλη πρόοδο από μήνες, χρειάζεται να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα ως προς την εξειδίκευση αυτού του εργαλείου, ώστε να γίνει ένα εργαλείο δημόσιο. Ένα εργαλείο που να επιτρέψει στους μεν και τους δε να γνωρίζουν τις προβλεπόμενες αλλαγέ μεταβολέ στην αγορά. Στο επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν από τρει μήνε, είχατε αναγνωρίσει ότι οδεύουμε προ μια κρίση στι αρχέ αυτή τη χρονιά. Κάτι που το έλεγαν όλοι οι φορεί τη αγορά. Η κρίση ίσω να μην είχε τέτοιε εκτάσει σήμερα. Διότι να θυμίσουμε ότι μόνο 1 έω 2% του πλεονάσματο γάλακτο στην αγορά κάνει, προκαλεί την κατάρρευση των τιμών κατά 5%. Αυτό ε, είναι ένα σημείο στο οποίο θέλω οπωσδήποτε να μείνω. Και ένα άλλο θέμα στο οποίο θέλω να εμείνω είναι η δράση μας σε περίοδο κρίσης. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια σαφή διάκριση μεταξύ των τάσεων των τιμών της αγοράς μακροπρόθεσμα και των εργαλείων διαχείρισης των ε, προσωρινών για να αντιμετώπιστε μια κρίση. Οι τιμέ παρέμβαση αυτή τη στιγμή είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Συμβουλίου και μα το θύμισε κιόλα. Δικό του το παιχνίδι. Τώρα πρέπει να προβλέψουμε τέτοιου κανόνε που επιτρέπουν τη ρύθμιση τη παραγωγή με τρόπο ε, σύντομο, ε, άμεσο για βραχυπρόθεσμε καταστάσει. Αυτό είναι η βασική λύση που έχουμε μπροστά μα. Ιδάλω θα καταλήξουμε σε μια ομαδική ε, καταστροφή. Ο κύριος Σεράου. Ευχαριστώ να ευχαριστήσω και το δεύτερο πάνελ εμπειρογνωμόνων τους 15 προσώπους και ε, ηθήνοντες από το γαλακτοπαραγωγικό τομέα ε, αλλά να πω ότι από την ε, Πορτογαλία έφυγαν τουλάχιστον δύο εταιρείε από τι Αζόρε και το βορρά τη Πορτογαλία και του βλέπουμε εδώ στο πάνελ αυτό των προγνώμων των εταιρεών αυτών στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό εξισορρόπηση τη προσφορά και τη ζήτηση, ιδίω σε ζώνε όπου υπάρχουν και άλλε οικονομικέ εναλλακτικέ. Με φυσικού περιορισμού για την παραγωγή, όπω στην ε, περιοχή των Αζωρών ή με ε, περιοχές όπου το 70% της οικονομίας της γεωργικής περιοχή είναι η παραγωγή του γάλακτος. Έτσι μόνο θα έχουν πραγματικό νόημα τα μέτρα μα. Όμω, για την ευρωπαϊκή προσέγγιση, θα ήθελα να σχολιάσει εδώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε λάβει υπόψη ότι υπάρχει ετερογένεια στην αγορά με την κατάργηση των ποσοστώσεων και ότι θα αντιδράσει διαφορετικώ κάθε μια περιφέρεια τη Ιβύρου. Ε, Ποιο μηχανισμό θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιδράσει ευρωπαϊκά και συνολικά για να ε, αντιμετωπίσει εντοπίσει του τομεί με τι διαφορετικέ αδυναμίε. Ευχαριστούμε ο κύριο Ντότσο. Thank you, uh, Κυρία Ντότς, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η γαλακτοπαραγωγή της Βόρειας Ιρλανδίας έζησαν δραματικά χαμηλές τιμές από το 2014 και μετά. Τώρα είναι 22 πένες το λίτρο, πράγμα που μεταφράζεται σε περίπου 26 σέντ του ευρώ λεπτά. Αυτό πιέζει πάρα πολύ τις οικογενειακές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τους προοδευτικούς γεωργούς που έκαναν μεγάλες επενδύσεις στην επιχείρησή τους. Ακούσαμε πολλές πιθανές λύσεις, αλλά κυρίως μέσω και μακροπρόθεσμες. Δεν λύνουν αυτές όμως τα άμεσα προβλήματα ρευστότητας των γεωργών και στην Ιρλανδία και σε ολόκληρη την Ένωση. Θα ήθελα να ρωτήσω τον καθένα από τους εμπειρογνώμονες, να του ζητήσω να ταυτίσουν τα πιο άμεσα μέτρα που θα μπορούσε να πάρει η Κομισιόν για να υποστηρίξει τους γαλακτοπαραγωγούς και να σταθεροποιήσει την αγορά. Επίσης θα ήθελα να τους ζητήσω να μας πούν και ένα λογάκι ακόμα για το τι θα γίνει την άνοιξη μετά τις ποσοστώσεις εφόσον δεν συμβεί καμία μεγάλη ανατάραξη. Ευχαριστώ. Φυσικά πρέπει να προσαρμόζεται η προσφορά με τη ζήτηση και άρα οι τιμές του γάλακτος να συνδέονται με τις διεθνείς. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος υπερπαραγωγής. Γι' αυτό δεν είμαι πάρα πολύ υπέρ ψηλότερων τιμών παρέμβασης και επιστροφών προς τις εξαγωγές. Αντίθετα πρέπει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης είμαι υπέρ της κατάργησης των Συμφωνώ με τον κύριο Σατελιέ για το ποια είναι τα εργαλεία για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και του κυρίου Άννελε ότι πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία για τα Natura 2000 ας πούμε. Επίσης θέλω να ρωτήσω την κυρία Φανκάμπ αν το σύστημά της αυξάνει την ανταγωνιστικότητα διεθνώς ή αν τη μειώνει. Ευχαριστούμε. Μίλλερ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους εμπειρογνώμονες που μας έδωσαν μια τόσο σφαιρική εικόνα. Μπορώ να εξαγάγω πολύ καλά συμπεράσματα και ως ε, γαλακτοπαραγωγός που έζησα 30 χρόνια με τις ποσοστώσεις πρέπει να πω ότι χαίρομαι που επιτέλους καταργούνται. Μας κόστησαν πολλά χρήματα σε εμάς τους ε, αγρότες για να έχουμε το δικαίωμα να παράγουμε γάλα. Θεωρώ ότι αν θέλουμε να στηρίξουμε τις μειονεκτούσες περιοχές πρέπει να στείλουμε το αναγκαίο μήνυμα που να το συνοδεύσουμε με συνοδευτικά μέτρα και ειδικά προγράμματα. Οι ποσοστώσεις ποτέ δεν περιόρισαν τις διαρθρωτικές αλλαγές. Αντίθετα, Πολλές εκμεταλλεύσεις τα παράτησαν ναι, με ή χωρίς ποσοστώσεις. Ερωτήσεις προς την Κομισιόν τώρα. Πρώτον, θα ήθελε να αυξήσει την τιμή παρέμβασης ε, η Κομισιόν και πώς θα διατηρήσει την νομική βάση ούτω ώστε να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία από το παρατηρητήριο. Ευχαριστώ πολύ. Χόιμπους. Ευχαριστώ. Ακούσαμε πολλές αναλύσεις. Τι ακριβώς μπορεί να αλλάξει. Και πάντα η κόκκινη γραμμή ήταν συμβόλαια, δηλαδή τα βασικά συνθήματα, συμβόλαια και εξαγωγές. Αλλά συμβόλαια που να καλύπτουν την τιμή παραγωγής μπορεί να υπάρχουν μόνο αν λειτουργεί κάπως η αγορά. Τα συμβόλαια δεν αντιμετωπίζουν ριζικά το πρόβλημα αντίθετα οδηγούν σε αβεβαιότητα. Πρέπει να υπάρχει δυνατότητα επαρκής, επαρκούς ε, προσαρμογής της προσφοράς. Και εγώ είμαι 30 χρόνια τώρα παραγωγή, ε, γαλακτοπαραγωγός και μπορούμε να έχουμε εξαγωγές μόνο αν υπάρχουν ε, αγελάδε που να παράγουν γάλα. Γιατί προκύπτουν συνέχεια κρίσεις και όλο πρέπει η παραγωγή να αντιμετωπίσουμε τις ε, συνεχείς κρίσεις. Άρα τα προγνωστικά είναι λάθος και οι απαντήσεις επίσης λάθος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κοιτάξατε σε λάθο κρυστάλλινη σφαίρα. Νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα να έχουμε αυτόν τον οργανισμό ε, εμπορία του γάλακτο. Σάιλε. Ευχαριστώ πολύ. Ο υπουργό μας ήταν πολύ περήφανος ε, για τον κλάδο μας στην Ολλανδία. Είπε έχει πολύ παραγωγή, αλλά έχουν ε, μειωθεί πολύ οι τιμές. Κάποτε παίρναμε 51 λεπτά, τώρα παίρνουμε 30, ενώ ο καταναλωτής πληρώνει τα ίδια. Οπότε η ερώτηση στους πρώτους δύο μιλητές δεν θα έπρεπε να κάνουμε ό,τι μπορούμε τόσο ώστε οι συνεταιρισμοί να έχουν καλύτερη ηγεσία και επίσης και οι οργανώσεις ε, καταναλωτών ούτω ώστε να καταναλώνονται περισσότερο οι παραγωγές των μικρών ε, εγκαταστάσεων στην Ήπεθρο. Αυτό θα μας βοηθούσε και μέσω του δεύτερου πυλώνα οι, τις υποχρεώσεις του Natura 2000 τις έχουμε και στην Ολλανδία. Θέλουμε να διατηρήσουμε τις ε, ε, εκμεταλλεύσεις, αλλά όχι μόνο για την παραγωγή γάλακτος, αλλά και για την προστασία της υπέτρου. Τόσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Αναφερθήκατε και στην κατάσταση των εκμεταλλεύσεων σε μειονεκτικέ περιοχές, ορεινέ κτλ. Συμφωνώ απόλυτα και συμφωνώ και με ορισμένους που είπαν ότι με αύξηση της τιμής παραγωγής δεν δίδεται πλεονέκτημα, δημιουργείται μειονέκτημα για αυτές τις περιοχές. Γιατί η αύξηση τη τιμής παρέμβασης θα βοηθούσε περισσότερο τι περιοχές όπου είναι πολύ πιο εύκολη η παραγωγή. Θα έκαναν περισσότερες ε, επενδύσεις, θα άξαναν ακόμη περισσότερο το μερίδιο αγορά που κατέχουν. Οπότε σε ορνέ περιοχές μόνο ζημιά θα έχουμε. Γιατί χωρί περιορισμό των ε, ποσοτήτων και χωρί ποσοστώσεις δεν βοηθάμε. Να αναφερθώ τώρα στα εξή. Οι όρνε περιοχές θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο στι πιο ευνοημένε περιοχέ δεν έχει κλείσει η εσωτερική προσπάθεια επίτευξης συνοχής. Πρέπει λοιπόν να γίνει ό,τι μπορεί να γίνει ούτως ώστε να μην συνεχίζεται η κατάσταση όπου λαμβάνουν πολύ διαφορετικά ποσά οι διάφοροι παραγωγοί. δεν αντιμετωπίζονται όλοι ισότιμα. Δηλαδή ε, αυτοί οι οποίοι είναι στην παιδιάδα λαμβάνουν περισσότερα. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν, ε, πρέπει να γίνονται θετικές διακρίσεις υπέρ των ε, εκμεταλλεύσεων σε ορεινές περιοχές. Δηλαδή περισσότερη στήριξη για παράδειγμα για τους παραγωγούς και τους μεταποιητές στις ορεινές περιοχές, ούτως ώστε να ευνοήσουμε αυτές τις περιοχές γιατί χρειάζονται αυτή τη στήριξη η Γεωργία εκεί. Μαγκίνας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το σχόλιο που μου έκανε τη μεγάλη εντύπωση προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μου έκανε εντύπωση που και εκείνοι ξυπλάγησαν και ευνηδιάστηκαν που οι τιμέ του γάλακτο ε, έπεσαν στο τέλο του χρόνου γιατί αποδυναμώθηκαν. Η ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Τροπή. Κατά την άποψή σα, η τιμή ε, έπεσε μόνο λόγω τη αγορά και την ε, ζήτηση, το πρόβλημα τη Ρωσία και την αποδυνάμωση τη Κίνα. Εσεί τι κάνατε για να προλάβετε την αύξηση 5% στην παραγωγή του γάλακτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ακούσαμε την πρόταση των ε, του Συμβουλίου για το Γάλα της Ευρώπης, ε, αλλά ουσιαστικά μιλάμε για ποσοστώσεις του γάλα εκτός από το παραθυράκι, έτσι. Είχαμε ποσοστώσεις για 30 χρόνια και όταν ε, τις προβλέψαμε, που ήταν για μια πενταετία αρχικά, περάσαμε σε μια εποχή που δεν έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν. Είναι καιρή και κινδύνου και ευκαιριών όμως. Αυτό που θα ήθελα να μου κάποιο από το πάνελ είναι εάν νομίζετε ότι και τώρα διανύουμε κρίση. Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει πως όχι. Όμως βλέπετε να υπάρχουν ευκαιρίες, διότι νομίζω ότι όλοι γινόμαστε απεσιόδοξοι όταν η αγορά πέφτει. Πέρσι, όταν η αγορά ήταν ψηλά, δεν ακούγαμε απεσιόδοξα σχόλια. Μπορεί κάποιος να απαντήσει. Ο κύριος Βιάγκας, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Η συζήτηση αυτή καλό θα ήταν να συγκεντρωθεί και στο παραγωγικό μοντέλο που έχουμε δημιουργήσει και τι θέλουμε για την Ευρώπη ως προς το μοντέλο παραγωγής. Θα θυμάστε, το 2014 ήταν το διεθνής έτος της οικογενειακής γεωργίας. Ε, Όπω θα ξέρετε, ε, το Παγκόσμιο Έτο τη ε, Οικογενειακή Γεωργία λοιπόν, και η Οικογενειακή Γεωργία η ίδια δίνει πολύ μεγάλη δυνατότητα για την παραγωγή τροφίμων, για, την, ε, για το εμπόριο εγκύτητα, για την ασφάλεια των καταναλωτών, για τη βιοπικιλότητα, για την ε, δημιουργία τη αναπασχόληση και ούτω καθεξή. Έχουμε στην Ευρώπη ένα παραγωγικό μοντέλο που ακόμη βασίζεται στι μικρομεσαίε οικογενειακέ εκμεταλλεύσει. Αυτό πρέπει να, να διαφυλαχθεί. Και έχουμε δει τι γίνεται στην περίπτωση του γάλακτο μεγάλη συγκέντρωση που επηρεάζει αυτή την ισορροπία και μας προσεγγίζει στις μεγάλες ε, εταιρείες των ΗΠΑ. Το θέμα είναι να δούμε κατά πόσον η δομή του παραγωγικού μας μοντέλου θα ληφθεί υπόψη στην λέξη ίσως για το γάλα. Χάρενς Γκαρσία, ευχαριστώ πολύ. Εγώ εξακολουθώ να πιστεύω αυτό που άκουσα, που πίστευα και πριν ε, έρθω εδώ, ότι είναι πολύ ετερογενής η κατάσταση. Δηλαδή, αν κάποιοι μπορούν να παράγουν να ε, παραγάγουν γάλα για την εξαγωγή, γιατί να τους το απαγορεύσουμε. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη τις διαφορετικές καταστάσεις. Οι Ισπανοί μιλάμε κυρίως για τα θέματα με τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν έχετε κι εσείς ε, τέτοια προβλήματα. Και εδώ μπορεί να υπάρχει διαφορετικότητα καταστάσεων. Θα ήθελα να μου πείτε ότι δεν θα έπρεπε πρώτα απ' όλα να ορίσουμε τι σημαίνει κρίση. Δεν είναι το ίδιο το επίπεδο της κρίσης στην Ισπανία με την Κροατία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θα έπρεπε να ορίσουμε τι σημαίνει κρίση για να ξέρουμε τι θα χρησιμοποιούμε για να ενεργοποιούμε μηχανισμούς αντιμετώπισης κρίσης. Και δεν θεωρείτε ότι το παρατήριο τιμών Περιφεροποιημένο, όπως η κυρία Ουγιώα θα ήταν ε, πολύ χρήσιμο και αναγκαίο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Διευθυντής κύριος Κρουτά. Πέντε λεπτά. Και μετά οι εμπειρογνώμονες για δύο λεπτά ο καθένας. Παρακαλώ κύριος Διευθυντής. Ευχαριστώ πολύ. Τέθηκε μια σειρά από ερωτήσεις. Θα ήθελα να πω ε, ότι ήταν εξαιρετικέ οι παρουσιάσει που ακούσαμε και λεπτομερέστατε. Το πρώτο σχόλιο που προήλθε από πολλέ από τι ερωτήσει και από τι παρουσιάσει, ε, εάν είμαστε ή όχι σε κρίση και γιατί δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψει μια κρίση. Στο Συμβουλίο των Υπουργών χθε καθόμουν δίπλα στον Επίτροπό μου και είχα αυτό το προνόμιο, ο οποίο ε, αμφισβήτησε ότι υπάρχει κρίση. Και αν δούμε τι τιμέ ε, και τα κενά του, ε, όπω εμεί πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να είναι, θα είχαμε πολύ καλύτερε τιμέ κατά τον κύριο Νταντέν. Χθε ρωτήσαμε 7 έω 8 κράτη-μέλη γιατί δεν μα έχουν δώσει τι αριθμητικά στοιχεία από τον Νοέμβριο. Δεν τα έχουμε οι αριθμοί που έχουμε και οι μετρήσει μα δεν συνάδουν στο ότι υπάρχει κρίση ευρωπαϊκή. Υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα, υπάρχουν τριγμοί. Ήμουν ο πρώτο που όταν ξεκίνησα με το απόγευμα είπα και εξήγησα προ όλου ότι επεξεργαζόμαστε τα σχετικά ζητήματα και συμμεριζόμαστε τι ανησυχίε πολλών από του γεωργού, αλλά Όντω, το επίπεδο των τιμών είναι πολύ χαμηλό στι χώρε τη Βαλτική και αλλού, αλλά συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη γνώση μα, δεν υπάρχει κρίση. Νομίζω είναι σημαντικό λοιπόν να μην θυποβληθούμε ε, πιστεύοντα ότι υπάρχει κρίση. Δεν θα πρέπει να το αφήσουμε εμεί να το πιστέψουμε. Γι' αυτό χάρηκα που άκουσα και πολλούς σήμερα το απόγευμα να λένε ότι οι προοπτικές είναι καλές. Θα μπορούσα να πω πολλά για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει τους επιχειρηματίες και τους παραγωγούς να βρουν πρόσθετες ε, αγορές, να βρουν εναλλακτικέ της ρωσικής αγοράς που χάσαμε, ίσως και για πολύ καιρό και για τα αμυντικά μας, ε, τα επιθετικά μας μάλλον ε, συμφέροντα, ειδικά και σε σχέση με το TTIP, διότι οι εμπειρογνώμονές μας συμφωνούν, συμφωνούν όταν μιλάμε για τα γαλακτοκομικά, γαλακτοκομικά λέγω, έχουμε ε, με επιθετικά συμφέροντα ως προς το TTIP και την αγορά των ΗΠΑ, αλλά και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και την ιδιαίτερη προστασία με αξία που έχουμε, δεν φοβούμαστε τίποτα. Οπωσδήποτε Πρέπει να εργαστούμε ακόμη σκληρότερα με τους οικονομικούς ε, παράγοντες για να βρούμε περισσότερες διεξόδους. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν έχουμε κρυστάλλινη σφαίρα. Εάν την είχαμε δεν θα καθόμουν εδώ αλλά θα ήμουν στην Καραϊβική σε μια παραλία και θα έλεγα το μέλλον. Ε, εάν ε, λοιπόν σας φάνηκε ότι δεν το έχουμε μελετήσει σοβαρά το θέμα ε, να σας διαβεβαιώσω ότι στον τομέα των γαλακτοκομικών έχουμε κάνει τεράστιες προσπάθειες για να αξιοποιήσουμε ό,τι υπάρχει στα χέρια μας. Δεν θα πάψουμε. Θα συνεχίσουμε να ε, προσπαθούμε. Με ό,τι συνεισφορά έχουμε και με τη στήριξη της Επιτροπής σας θα τα καταφέρουμε ακόμα καλύτερα. Επίσης ένα σημείο για το τι ετοιμασία είχαμε και γιατί δεν αντιδράσαμε. Η απάντηση είναι φυσικά και ήμασταν προετοιμασμένοι. Η απόφαση ελήφθη το 2013 να φύγουμε από το σύστημα των ποσοστώσεων. Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη ελαφρά την καρδία. Η φιλοσοφία που ακολουθούμε για όλη την ΚΑΠ ισχύει και για τις ποσοστώσεις του γάλακτος, για όλα τα προϊόντα το ακολουθήσαμε αυτό. Περάσαμε από τη στήριξη των τιμών στην άμεση στήριξη των προϊόντων. Με ένα κουτί εργαλείων για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει και ιδιαίτερες περιστάσεις. Αυτή την απόφαση λάβαμε έχοντας πλήρη επίγνωση και για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Και τέλος, το 2014, ο τομέας των γαλακτοκομικών φαίνεται να έχει εκτεθεί σε αυτή τη λογική είναι δύσκολο. Θα ξανακάνουμε την ίδια συζήτηση για τη ζάχαρη που, θα ακολούθησε το 2007 και χθε στο Συμβούλιο το συζητήσαμε ήδη μια φορά. Παρόμοιε ανησυχίε. Αλλά και πάλι δεν θα έλεγα ότι συμφωνώ να χρησιμοποιήσουμε τι δυσκολίε των παραγωγών ω. Ε, το με την απομάκρυνση από το σύστημα των ποσοστώσεων προ ένα άλλο σύστημα. Η διαχείριση που είχαμε τώρα προφανώ δεν επαρκεί ούτε οι τιμή τη παρέμβασης και αυτή η συλλογιστική. Είναι παροχημένη η συλλογιστική και λόγω τη νέα αντίληψη για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ μην ξεχνάμε ότι ήμασταν πρώτο εξαγωγέ το 2013 ε, για που και πολλά άλλα προϊόντα. Ω προ αυτά, ε, πρόεδρε, νομίζω ότι απήντησα τι ερωτήσει που απευθύνονταν τουλάχιστον προ εμένα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, γαλακτοπαραγωγή, γεωργή, συνεργατικέ οργανώσει, συνεταιρισμοί. Από ό,τι ξέρω και από όσα άκουσα, βλέπουμε εδώ να περιγράφεται η αρχή μιας κρίσης. Θα επανέλθω λοιπόν για δύο λεπτά στους ομιλητάς και αρχίζουμε από τον καθηγητή Τόιφσεν. Ευχαριστώ. Πολλές ερωτήσεις, πολλές προτάσεις. Πέντε σε δύο λεπτά. Ε, μέσω των οποίων μπορώ να απαντήσω σε πολλές ερωτήσεις. Κατά τη γνώμη μου, η ποσόστοση δεν πρέπει να επανέλθει η ποσόστοση καλύτερα δεν πρέπει να θεωρείται πανάκια, δεν ε, αντιμετώπισε τις κρίσεις. Δεύτερον, να καθορίσουμε την προσφορά ε, μέσω ενός ευρωπαϊκού οργανισμού για το γάλα, δεν είναι ρεαλιστικό. Η μεταβλητότητα των τιμών δεν είναι κρίση οι τιμές μεταβαλλονται άλλοτε είναι χαμηλές και άλλοτε υψηλές άρα είναι θέμα διαχείρισης από κάθε εκμετάλλευση και πρέπει να μπορούν να προσαρμοστούν όταν είχαμε για, για τρία χρόνια υψηλές τιμές ε, δεν είναι τρομερή κρίση εάν έχουμε ένα μήνα χαμηλών τέταρτον η παραγωγή γάλακτος θα συγκεντρωθεί ακόμη περισσότερο στις πιο ευνοϊκές περιοχές. Γιατί δεν είναι μόνο οικονομικά τα πλανεκτήματα μεγάλων επιχειρήσεων και κοινωνικά είναι ωφέλιμο. Άρα θα συνεχιστεί αυτή η συγκέντρωση. Και τελευταίο, η στήριξη των μειωτικών περιοχών είναι απόλυτα αιτιολογημένος πολιτικός στόχος, αν και ως ε, επιστήμων, δεν πρέπει να μιλήσω για το πόσο είναι αιτιολογημένη πολιτική. Αυτό δεν πρέπει να γίνει μέσω πολιτική αγορά και πολιτική παρέμβαση των τιμών. Θα επιτύχει μόνο να διατηρηθεί κάποια περιφέρεια ω γαλακτοπαραγωγός μόνο μέσω ειδικών προσαρμοσμένων για την περιφέρεια αυτή πολιτικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σιέτα Φων Καμπένα. Εάν θέλετε να επιλύσετε την κρίση, θα πρέπει να δείτε τι είναι το πρόβλημα. Ίσως το πρόβλημα είναι ότι απολέσαμε κάποια στοιχεία της αγοράς, είναι επειδή δεν αναπτύξαμε νέες, αλλά υπάρχει το πρόβλημα της μείωσης των, της των τιμών. Και αν δείτε τι γίνεται με τα εργαλεία της κρίσης, που λειτουργούν μόνο όταν υπάρξει κρίση, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για την ε, διαχείριση της ε, Μεθιάς, διότι υπάρχει θέμα κρίσης. Όταν θα ξανααναρρώσει η αγορά θα μπορεί πάλι ο καθένα να κάνει ό,τι θέλει. Όμως το θέμα είναι τι κάνουμε με τους παραγωγούς. ώστε η γαλακτοπαραγωγική βιομηχανία να επεκταθεί και σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η λύση. Ώστε ο γαλακτοκομικός τομέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως το χείριο και στα πολιτικά, να επεκταθεί. Θα πρέπει να συγχαίρουμε τους εαυτού μας που στη γαλακτο κομική παραγωγή μόνο σε, μικρά, ε, μια σε μικρούς θύλακες στην Ευρώπη υπάρχουν προβλήματα και ελλείψεις και ε, τον Σεπτέμβριο πήγα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα συμπόσιο, ήταν όλοι πολύ θετικοί και έλεγαν ότι το μόνο που μειώνεται δραστικά είναι ο αριθμός των γαλακτοπαραγωγών. Αν αυτή είναι η γαλακτοκομική μας πολιτική για την σταθεροποίηση της αγοράς και για να έχουν ένα σταθερό εισόδημα οι κοινότητες των κτηνοτρόφων, αυξανόμενα τα ατομικά οσοδήματα όσων ε, ε, ασχολούνται με την κτηνοτροφία, Ίσως ε, κάτι δεν καταλαβαίνω καλά, ίσως να μην καταλαβαίνω καν την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Και λυπάμαι πάρα πολύ που κατά αυτόν τον τρόπο, εάν δεν ορίσουμε τι ε, σημαίνει κρίση, εάν δεν θέλουμε να λύνουμε προβλήματα ε, βάζοντας όσους ρηπαίνουν την αγορά να πληρώνουν, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Και δεν θα σωθεί και αυτό το κοινοβούλιο, ούτε αυτός ο τόπος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, πολλά σχόλια έγιναν για τον ορισμό της κρίσης και για το ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Υπάρχει μεγάλη ετερεογένεια σε όλη την Ευρώπη, μεγάλη διαφορά μεταξύ του κόστους ε, κίνησης των ε, διαφορών μονάδων παραγωγής. Το θέμα είναι πώς θα ορίσουμε μια περίοδο κρίσης. Εδώ πρέπει να γίνει πολλή δουλειά ε, και κατάντη ανάντι μάλλον και για να δούμε τα διάφορα βάρη ή φορτία που δεν μπορούν να απομειστούν οι γεωργοί η παραγωγή, όπω το κόστο παραγωγή. Δεν υπάρχει απλώ κρίση, όχι απλώ μάλλον δεν υπάρχει κρίση παγκοσμίω. Υπάρχει αύξηση τη ζήτηση. Η ευρωπαϊκή αγορά θα πρέπει να έχει λίγο εφάνταστε λύσει να προτείνει και το βλέμμα στραμμένο λίγο προ τα έξω. Δεν είναι φιλελεύθερη η ομιλία μου υπέρ τη φιλελεύθερη πολιτική, αλλά υπάρχουν δύο φοβερή παραγωγή εκτό ε, Ευρώπη. Η Νέα Ζηλανδία που σε μια δεκαετία μετά παρατηρεί την αγορά τη και η ΗΠΑ που παράγουν προϊόντα χωρί ιδιαίτερε περιβαλλοντικέ ανησυχίε. Η Ευρώπη λοιπόν θα βρεθεί ε, συνεπή και θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία τη επέκταση προ τι εξωτερικέ αγορέ. Ο στόχο δεν είναι να αυξηθεί η παραγωγή προ όλε τι κατευθύνσει. Απλώ να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε να ε, κατευθύνονται στην ζήτηση σε πραγματικό χρόνο. Και έπειτα το θέμα είναι να θα είμαστε σε θέση να βρούμε μορφέ ρύθμιση, και αυτό είναι το θέμα, μορφέ ρύθμιση όχι εξατομικευμένε, αλλά συλλογικέ. Σε έναν κόσμο όπου το δίκαιο του ανταγωνισμού δεν διευκολύνει αναγκαστικά τα πράγματα. Επ' αυτού ε, πρέπει να βρούμε λύσει στην Ευρώπη. Και θα συμφωνήσω με πολλού από όσου είπαν ότι στην, μεσ, στην βραχυπρόθεσμη παρέμβασή μας. Δεν χρειαζόμαστε εργαλεία μόνιμα για τον γαλακτοκομικό τομέα. Είναι εύρωστο ο τομέα αυτό. Έχει περιόδου εφορία που αναπτύσσεται. Αλλά αυτό που είπε ο κύριο Ντε, μια ε, εταιρεία που τα καταφέρνει ή δεν τα καταφέρνει, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την Ευρώπη. Έχει να κάνει και με την ικανότητα των επιχειρηματιών και των διευθυντών των επιχειρήσεων να προβλέψουν σχέδια καλή διάρθρωση μια επιχείρηση. Θα πρέπει λοιπόν την Ευρώπη να χαιρόμαστε που υπάρχουν εταιρείε με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο για του υπολείπου επειδή έχουν καλέ ιδέε οι ίδιοι. Και ω προ τον εξυγχρονισμό όσων πιστεύουν στο μέλλον του γάλακτο, να πω ότι είμαστε στην ίδια πλευρά. Ευχαριστώ. ωραία όλα αυτά. Όμως Πώ τη φαντασία να τη μεταφράσουμε σε κάτι χειροπιαστό για του κτηνοτρόφου μα. Και τώρα ο κ. Τόμπιν. Καταρχήν, υπάρχει κρίση. Αν ρωτήσω του γεωργού τη περιφέρειά μου, θα μου πούνε οπωσδήποτε. Βελτιώνονται τα πράγματα, σταθεροποιούνται οι αγορέ. Μπορεί, αλλά όλοι ανησυχούν ότι θα ξαναπέσει η αγορά την άνοιξη. έχουμε δει ακόμη καμιά βελτίωση. Τι να γίνει τώρα. Πολιτικά είναι αποδεκτό να αφήσουμε τους γεωργούς να καταστραφούν και να μην έχουν ένα δίκαιο εισόδημα. Θα τα λύσει όλα μόνη της η αγορά. Μπορεί, αλλά με τρόπο που μπορεί να είναι κοινωνικά απαράδεκτος. Στο ερώτημα αν το European Milk Board έχει σωστές προτάσεις, ε, είναι, έχουν κάποια αξία αλλά πρέπει εκτός από την κατάργηση των ποσοστώσεων να βρεθεί και κάποιος τρόπος για να γνωρίζουν οι γεωργοί για την ε, τακτοποίηση των τιμών τι είναι κρίση και τι δεν είναι. Το να λέμε ότι θα τιμωρήσουμε όσους υπερπαράγουν και θα βραβευθούν όσοι προσαρμόζονται δεν είναι απλό. Ο ορισμός της ε, έκδηλης κρίσης μπορεί είναι σίγουρο ότι θα λύσει τα πράγματα αυτόματα με την αγορά. Εδώ η πραγματικότητα είναι ότι οι χαμηλές τιμές δεν επιτρέπουν στον ιδιωτικό τομέα να αντιδράσουν. Ο Άλφα Ντέντερλε. Λοιπόν, πολύ σύντομα. Υπόθηκε ότι είπα ότι όλα είναι θαυμάσια. Εγώ είχα καθήκον να πω τα πράγματα όπως είναι. Να αναφέρω λοιπόν τα στοιχεία το 13, που δεν υπήρχε κρίση. Η μέση τιμή ήταν 35,9 λεπτά στην Ελλάδα, 44,2, στη Ρουμανία 26,4. Δηλαδή το θέμα είναι για ποια χώρα μιλάμε θα μπορούσαμε να πούμε ότι στη Ρουμανία υπήρχε κρίση. Αλλά πρέπει να βρούμε και έναν ορισμό. Να συμφωνήσουμε. Οι ποσοστώσεις δεν σταμάτησαν τις διαθροτικές αλλαγές. Το παρατηρήσαμε στην περιοχή μας με πολλή ανησυχία. Θα συνεχιστούν οι διαθροτικές αλλαγές. Το είπα λοιπόν ότι χρειάζονται συνοδευτικά μέτρα ιδιαίτερα στις μειονεκτικές περιοχές. Ούτως ώστε να διατηρηθεί εκεί η παραγωγή. Χρειάζεται ένα δίκτυο ασφαλείας που υποσχεθήκαμε στους παραγωγούς όταν τους είπαμε ότι πρέπει να προσανατολιστούν προς την αγορά. Πρέπει λοιπόν να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας. Βεβαίως, να υπάρχουν ε, μοντέλα για την ε, εξασφάλιση των ε, εκμεταλλεύσεων. Είπαμε ότι είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση στην Ευρώπη. Έχουν μεγάλα προβλήματα όταν οι μεσαίες εγκαταστάσεις εγκαταστάσεις μεταποίησης που έχουν καλά προϊόντα θέλουν να στραφούν προς τις εξαγωγές διαπιστώνουμε ότι τους ζητάνε πολύ διαφορετικά πράγματα διάφοροι αγοραστές ζητάνε πολύ διαφορετικά πράγματα Κινέζοι, Ρώσοι κτλ. Θα ήταν καλό να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση ούτως ώστε οι μεσαίες επιχειρήσεις να ε, μην επηρεάζονται από γραφειοκρατικές υποχρεώσεις. Θέλουμε λοιπόν την υποστήριξή σας και όχι υπερβολικούς κανονισμούς, και γραφειοκρατία γιατί καταστρέφουν τις ευκαιρίες μας για το μέλλον. Ο κύριος Νίκολσον τώρα, που είναι ο εισηγητής μας, μας έχουν δώσει διαρμήσεις κάποιο χρόνο, ευχαριστούμε. Οπότε παρακαλώ εσείς κύριε Νίκος. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, όντως θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να ευχαριστήσω όχι μόνο τους διερμηνείς για τη γενοδορία τους, απλώς θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να μην τους κρατήσω ε, περιτά παραπάνω. Να ευχαριστήσω όλους όσοι έκαναν παρεμβάσεις εδώ σήμερα το απόγευμα. Είναι πραγματικά απίστευτο ότι έχουν περάσει 3,5 ώρες από την ώρα που ξεκινήσαμε. Ευχαριστώ όσους είχαν την υπομονή να μείνουν εδώ, άκουσαν τα πάντα και εγώ τουλάχιστον θαυμάζω όσους τα κατάφεραν. Σε αντίθεση με όσους ε, ήρθαν, κάτσαν κάποιες σημειώσεις και έφυγαν γρήγορα γρήγορα, ασκώντας και αντρεμία κριτική κάποιες φορές. δεν ήταν εδώ τη μεγαλύτερη διάρκεια της ακρόασης. Κατά τη δική μου λοιπόν άποψη, ε, έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που λέγαμε ότι πρέπει να είμαστε πολύ κοντά στην παγκόσμια αγορά. Πρέπει να διατηρήσουμε όμως το δικό μας μερίδιο στην ε, διεθνή αγορά και να το προασπιστούμε. Το θέμα είναι αν θεωρώ μάλλον ότι τα επίπεδα προστασία ε, και του δικτύου ασφαλείας είναι επαρκή. Όχι και δεν συμφωνώ με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον Επίτροπο, αλλά ε, ίσως έχει φύγει ο συνάδελφός σας, να του το μεταφέρετε. Η, κρίση υπάρχει. Υπάρχει πρόβλημα στις περισσότερες εκμεταλλεύσεις, το γνωρίζουμε από τις περισσότερες περιφέρειες και αυτό λέγεται κρίση. Δεν θα αντιμετωπιστεί εάν δεν βεβαιωθούμε και δεν ε, δούμε τον Απρίλιο, τον Μάιο, ποια ακριβώς είναι η κατάσταση. Δεν χρειάζεται βεβαίως πυρηνική φυσική για να καταλάβουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και ότι πρέπει να αναλάβουμε κάποια δράση για να το αντιμετωπίσουμε. Δεν θέλουμε πάλι οι ποσοστώσεις να από και να μπουν από το παραθυράκι. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα παράλληλο σύστημα. Απλώς να υπάρχει δίκαιη στήριξη για όσους παράγουν. Και όντω είναι εκτινοτρόφοι και οι παραγωγοί που υποφέρουν, όχι οι λιανοπολιτέ ούτε οι πολιτέ χοντρική. Η κυρία Μαγκίνε ετοιμάζει μία έκθεση για την Επιτροπή γεωργία για τι βάνομε ε, δραστηριότητε στην ε, τροφική αλυσίδα. Αυτό κύριε Πρόεδρε είναι κάτι που ελπίζω να το κάνουμε και εμείς αυτή την Επιτροπή για να δούμε πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Είναι σαφές ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που είχαμε στο κουτί από το πακέτο το γάλακτος. Πρέπει να πω ότι η παραγωγή πρέπει να είναι υπεύθυνοι δεν μπορούν να κλείνουν μόνο με συμβάσει που μπορούν να του συμφέρουν, αλλά και όταν πάλι του βολεύει μακροπρόθεσμε, πρέπει να, υπάρχει, να υπάρχουν ίσοι κανόνε του παιχνιδιού στην αγορά. Οι διακυμάνσει των τιμών δεν θα ε, εξατμιστούν θα επανέλθουν και θα επανέλθουν. Όπως στον τομέα του χειρίου και των πουλερικών και άλλων τομέων, όλοι χρειάστηκαν να το συνηθίσουν στο παρελθόν το νέο σύστημα. Πιστεύω λοιπόν και με βεβαίως καλωσορίζω το γεγονός μάλλον πιστεύω ακράταντα ότι για όσου λένε ότι χρειάζονται περισσότερε ποσοστώσει. Εάν βλέπετε ως λύση τις ποσοστώσεις, οι ποσοστώσεις προβλέφθηκαν για κάποιο σκοπό, η απόφαση είχε ληφθεί πάρα πολύ καιρό να καταργηθούν. Τώρα είτε συμφωνείτε είτε όχι θα καταργηθούν. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Μια λύση για τα προβλήματα που έχουμε σήμερα οι ποσοστώσεις δεν θα επανέλθουν για όσους τους επιθυμούν, ούτε βραχυπρόθεσμα, ούτε μακροπρόθεσμα. Κατά την άποψή μου λοιπόν, τώρα ποιο ξέρει, ίσως ο κύριος της Επιτροπής μας είπε ότι δεν έχει κρυστάλλινη γυάλινη μπάλα. Ε, κανείς μας δεν έχει. Ε, αν την είχαμε, κάθε τόσο θα τη χρησιμοποιούσαμε και θα βλέπαμε τα πράγματα πολύ διαφορετικά εάν ξέραμε να προβλέψουμε ακριβώς τι θα γίνει λίγο μετά. Όμως, Είναι άλλο να έρχεται κανείς όταν έχει εκ των υστέρων γνώσεις και να επικρίνει τις αποφάσεις που έλαβαν άλλοι στο παρελθόν. Όχι. Οι ποσοστώσεις ε, είχαν προβλεφθεί σε μια περίοδο που υπήρχε μια μεγαλύτερη κρίση που είχε γνωρίσει ο τομέας και δεν τον έστασαν, ε, δεν τον έσωσαν τότε το γαλακτοκομικό τομέα. Γιατί να τον σώσουν σήμερα. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο παρατηρητήριο της αγοράς, να είναι πιο ισχυρό, πιο εύρωστο, εάν μπορεί να αναλάβει ισχυρότερο ρόλο και πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε καλύτερα. Νομίζω, και εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Ντόρφμαν, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στις ορεινές περιοχές. Υπάρχει σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα σε αυτές τις περιοχές και θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί λύση εκεί. Και ε, ξανάρχομαι στο ερώτημα. Έχουμε αρκετά εργαλεία στο κουτί, έχουμε, τα χρησιμοποιούμε αρκετά, χρειαζόμαστε περαιτέρω στήριξη. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Και θέλω αυτό το μήνυμα να το περάσετε και στον Επίτροπο. Δεν θέλουμε να αυτοποβληθούμε και να πιστέψουμε ότι υπάρχει μια κρίση. Ε, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, όντω. Και πρέπει να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για κάποιον που είναι 26 χρόνια μέλος ε, του Κοινοβουλίου και αυτής της Επιτροπής. Έχω ξανακούσει την Επιτροπή να τα λέει αυτά στο παρελθόν. Έχω ε, ακούσει την ε, κυρία Φυσέρα μπορεί να λέει σε αυτή την Επιτροπή ότι ουδέποτε δεν θα χρειαστεί να κάνουμε βεβαιασμένε κινήσει μέχρι να δράσει η Επιτροπή. Το ίδιο κάνετε και τώρα. Πηγαίνετε και πείτε στον Επίτροπο ότι δεν δεχόμαστε αυτά που λέτε. Θα συνταχθεί μια έκθεση εδώ στο επόμενο μήνα και θα ξανάρθω στην Επιτροπή αυτή για να τα συζητήσουμε. Θα τα συζητήσουμε και θα φροντίσουμε να υπάρξει μια λογική θέση επί όλων των θεμάτων. Άκουσα όσα υπόθηκαν, τα έχω σημειώσει και είμαι πολύ ε, αποφασισμένος όταν λέω ότι το πακέτο των γαλακτοκομικών, με συγχωρείτε το πω, ξέρω ότι όλοι θα θέλατε να το πετάξουμε, αλλά ετοιμάζουμε μια ε, έκθεση, θα είναι υπεύθυνη και θα πρέπει να αναλυφθεί δράση αφού ακούστε τι έχουμε και εμείς να πούμε. Αυτά θα προσπαθήσω να κάνω και μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ας αναλάβει ε, τις ευθύνες της. Ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή του σήμερα και ευχαριστώ Πρόεδρε. Για την Προεδρία αυτής της ακρόασης. Ξεπεράσαμε μόνο κατά 5 λεπτά την ώρα μας, δεν είναι και άσχημα. Και αντέξαμε ήδη 3,5 ώρα. Ένα λεπτό μόνο. Το δίκτυο ασφαλείας που, που μας υποσχέθηκαν στην μεταρρύθμιση δεν έχει ακόμη μηχανισμό εφαρμογής και για τις εξωτερικές παραμέτρους. Ε, ε, έχουμε προβλήματα, έχουμε διάφορους παράγοντες εξωτερικούς που παίζουν ρόλο, όπως το ρωσικό εμπάργο ή το TTIP. Και χαίρομαι πολύ που ο κύριος Νίκολσον ξέρει πολλά και για το TTIP. Διότι θα πρέπει να συνδέσουμε την κατάστασή μας και με αυτές τις εξωτερικές ε, ε, δυσκολίες. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές, όλους τους ε, συναδέλφους, τους διερμηνείς. Νομίζω ότι ο χρόνος που αφαιρώσαμε αυτή τη συνεδρίαση χρησιμοποιήθηκε επικερδώς. Ευχαριστώ.